Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το θαυμάσιο βίντεο έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευρά του Προέδρου Αντώνιο Ταγιάννη που θα μας κάνει μια κεντρική ομίλια αργότερα. Χαίρομαι πολύ που ανοίγω αυτή τη ε, συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόσκληση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Μπορώ να σας πω ότι θα μεταφραστεί σε 23 γλώσσες. Οπότε αν θέλετε να ακούσετε οποιαδήποτε διερμήνια, μπορείτε να το κάνετε και επίσης πρέπει να σας πω ότι όπως πολύ συχνά στο Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται και τα δύο φύλλα εξίσου. Η διάσκεψη διοργανώνεται από τον πρόεδρο Ταγιάννη με τις αρμόδιες επιτροπές την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Επιτροπή Αλληλείας και την Επιτροπή Έρευνας και Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα με τη Γενική Διεύθυνση για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και άλλες υπηρεσίες κομισιών. Και καλωσορίζω και τους ε, επιτρόπους Βέλα και Μοέντας που ε, συμμετέχουν στη διοργάνωση και σε αυτήν την ανακτήρια συνεδρίαση. Παράλληλα, είναι θαυμάσιο που είναι εδώ και εκπρόσωποι της νέας γενιάς, α, και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο εκπροσώπους ε, νέων και πολλούς άλλους στην αίθουσα. Γι' αυτό καλωσορίζω θερμά τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό από τα ευρωπαϊκά σχολεία της Βρυξέλλης. Μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας. Ευχαριστώ. Καλώς ορίζουμε τη νέα γενιά. Αυτό καταδεικνύει ότι εκεί ανήκει το κλίμα, είναι στο κέντρο της προσοχής της νέας γενιάς και αυτό είναι θαυμάσιο. Κυρίες και κύριοι, η θαλάσσια πολιτική έχει διάφορες πλευρές δεν είναι δυνατόν να τα συζητήσουμε όλα σε μία μόνο εκδήλωση μισή μέρα, Αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και οι ομιλητές προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και ασχολούνται με διάφορες πλευρές της θαλάσση πολιτικής, έρευνα, οικονομικά θέματα και συμμετοχή των πολιτών. Και έχουμε τρεις συζητήσεις στο κλείστρα Πρώτον, η διακυβέρνηση των ωκεανών για το μέλλον. Ε, τώρα δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένους ομιλητές αλλά θέλω να καλωσορίσω θερμά την πρώην Επίτροπο για την Αλληλεία και τις θαλάσσιες υποθέσει Μαρία Δαμανάκη. Νομίζω ότι σε είδα να κάθεσαι εκεί, σε καλωσορίζουμε. Η κυρία Δαμανάκη ήταν υπεύθυνη για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής που ήταν ένα μεγάλο βήμα προόδου για την Ευρώπη. Η δεύτερη συζήτηση θα ασχοληθεί με τι προκλήσει για να υπάρξουν υγιεινεί και καθαρέ. Ε, συγγνώμη, ε, υγιείς και καθαρές θάλασσες για να αντιμετωπίσουμε τη μόλυνση. Και θα συζητήσουμε την μελλοντική πορεία στο τρίτο γύρο μιλητών για να προωθηθεί η γαλάζια οικονομία όχι μόνο στους παραδοσιακούς τομείς αλλά από και αναδυόμενους νέους τομείς όπως η παραγωγή φυκιών και η παραγωγή ενέργειας από τις θάλασσες. Ε, σε κάθε συζήτηση θα έχουμε ε, την Προεδρία του Προέδρου και Αντιπροέδρου των Αρμοντίνων Επιτροπών και άλλοι ευρωβουλευτές θα κάνουν και σύντομε δηλώσεις. Αγαπητοί φίλοι, δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε διάλειμμα, αλλά αν κατόπιν ε, βρείτε χρόνο, μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις που έχουμε και μπροστά και στις δύο πλευρές του ημικυκλίου. Θα δείτε καταπληκτικά παραδείγματα προγραμμάτων που χρηματοδότησε η Ένωση όπως ο Κοπέρνικος, που ασχολείται ιδιαίτερα και με θαλάσσιες υποθέσεις, ή το πρόγραμμα Μαρίνα και η υπεύθυνη κατάρτιση για τη γνώση των ωκεανών. Και Σήμερα συμμετείχα σε ένα διάλογο για τους ωκεανούς, όπου συζητήσαμε με νέους επαγγελματίε του τομέα, το Marina και το Responsible, και το μήνυμά τους είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στις καθημερινές συζητήσεις ε, των συμπολιτών μας να αναφέρω τα θέματα των ωκεανών. Ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει. Αυτό το, συζητάμε τουλάχιστον όλα Τα τελευταία δύο χρόνια επιτύχαμε να συζητηθούν πολύ περισσότερο οι ωκεανοί και οι θάλασσες και να γίνουν προτεραιότητα. Όχι μόνο λόγω τη μόνη από τα πλαστικά, δυστυχώ αλλά ευτυχώ και για άλλου λόγου. Είχαμε μεγάλε διασκέψεις όπω ο ωκεανό μα τον Παλί, φέτο ε, στην Νορβηγία και επίση μικρέ πρωτοβουλίε που οργανώνουν διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει για το καθαρισμό στι παραλίε. Ε, έχουν γίνει λοιπόν οι θάλασσε θέμα παντού, δεν το γνωρίζουν ακόμη όλοι, αλλά έχουμε κάνει πολλά. Καλό λοιπόν θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει μια επιτροπή για τι θαλάσσιε υποθέσει. Μάρε, όπου να μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα θαλάσσια θέματα. Και οι διασκέψεις που κάνουμε τώρα βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο καλό παράδειγμα θα ήταν το... η διαπολιτική ομάδα που έχουμε για τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα νησιά και τις παράκτης περιοχές. Το ακρονίμιο είναι ΣΥΡΙΚΑ. Το δημιουργήσαμε το 2014 για νέα πλατφόρμα για τα θαλάσσια θέματα και για να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση συνολικά η κοινωνία μας, οι οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Γιατί η ωκεανή και η θαλάσσια πολιτική είναι τόσο σημαντική για μας. Γιατί ζούμε σε έναν γαλάζιο πλανήτη. 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας είναι νερό και είναι ζωτική για το κλίμα. Διότι δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και παράγουν οξυγόνο. Κάθε δεύτερη αναπνοή μα περιλαμβάνει οξυγόνο που έχει παραχθεί στου ωκεανού και είναι πολύ σημαντική για το μέλλον τη ανθρωπότητα. Αυξάνεται ο πληθυσμό μα και χρειάζονται τροφή και από τους ωκεανούς, ενέργεια, μπλε, βιοτεχνολογία και βεβαίως ε, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι το 90% των ε, μεταφορών, αλλά απειλούνται οι ωκεανοί. Χρειαζόμαστε υγιείς ωκεανούς για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτό είναι σημαντικό φυσικά και για μας τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη είναι θαλάσσια ήπειρος. Η ακτογραμμή μας είναι 7 ε, φορές μεγαλύτερη από την ακτογραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνο πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακτογραμμή και είμαστε ηγέτες στην ε, πράσινη αυσιπλοεία, την ενέργεια από τα κύματα, από τα παλαιριακά κύματα και από τις ε, υπεράκτιες ε, ανεμογεννήτριες. Έχουμε εδώ τον καθηγητή Χέρτσιγκ που θα μας μιλήσει αργότερα για τα θέματα αυτά. Αλλά δεν χρειαζόμαστε μόνο περισσότερη έρευνα. Ξέρετε, ξέρουμε περισσότερα για τη σελήνη από ό,τι για τα βάθη των ωκεανών. Θέλουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για τους ωκεανούς. Θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή των ε, αποτελεσμάτων της έρευνας. Και πρέπει η επιστήμη να είναι σε σωστή επαφή με το λαό. Πρέπει να γνωρίζει ο λαός, οι συμπολίτε μας, τα των ωκεανών. Γι' αυτό πιέζουμε για πιλωτικά προγράμματα, για την γνώση, για τις θάλασσες. Και μόνο πριν από μερικές χρόνιες έγινε μια έκκληση από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για τα θαλάσσια θέματα. Και κάτι πολύ σημαντικό. Και η UNESCO προετοιμάζει τη δεκαετία για την ε, επιστήμη των ωκεανών που θα ξεκινήσει το 2021. Θα μα πει ο κ. Διαμήνιν περισσότερα γι' αυτά. Αγαπητοί φίλοι, η πολιτική των θαλασσών μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μακρά παράδοση. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν την ολοκληρωμένη ε, θαλάσσια πολιτική, την πλέη οικονομία, την κοινή γεωρική πολιτική, την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών. Βγάλαμε πρόσφατα ένα φυλάδιο και πρόσφατα είχαμε και οδηγίες για τα πλαστικά ούτω ώστε να καθαρίσουμε τους ωκεανούς μας. Όλα αυτά τα κάναμε σε στενή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμών της Ένωσης. Το Συμβούλιο επίσης, λοιπόν, μαζί με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλά για να προωθηθούν τα θέματα αυτά, αλλά πάντα στηρίχθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα Τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε στα κράτη-μέλη αυτά που αποφασίστηκαν. Ναι, μεν ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Και επίση οι νέοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν μπλε σταδιοδρομίε για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Σε στενή συνεργασία με οργανισμούς όπως ο ε, οργανισμός που θέλει να σταματήσουν οι πλαστικές σακούλες και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες ε, που κάνουν πορείες για το περιβάλλον ή με νέους καινοτόμους ηγέτες που ασχολείται με την αντιμετώπιση των σκουπιδιών στον ειρηνικό. Η Ένωση είναι παγκόσμια πρωτοπορία στην έρευνα και καινοτομία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα προτερήματά μας για να επιτύχουμε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στο επόμενο πλαίσιο ε, για την έρευνα να έχουμε ειδικό κεφάλαιο για τι θάλασσε και του ωκεανού. Επίκυνται οι ευρωεκλογέ, το ξέρετε. Έχουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση για το μέλλον του γαλάζιου πλανήτη. Οι ωκεανοί βέβαια δεν ε, ψηφίζουν, ε, δεν είναι ψηφοφόροι, αλλά είναι πολύ σημαντικοί για μα. Κάποιο που τα ξέρει όλα αυτά, τη σημασία των ωκεανών λοιπόν, θα συμφωνήσει απόλυτα νομίζω ο οποίο φιλοξένησε την διάσκεψή μα για του ωκεανού στη Μάλτα το 2017 είναι ο επίτροπο μα για θέματα αλληλεία, Καρμίνου Βέλα, στον οποίο θα δώσω τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι Γκεζίνε, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε Κάρλος, αγαπητή Τέος Επίτροπε Μαρία, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε εδώ να συζητήσουμε μαζί το μέλλον του γαλάζιου πλανήτη μας. Όπως πολλοί Ευρωπαίοι, μεγάλωσα και εγώ δίπλα στη θάλασσα κυριολεκτικά και έχω πάρα πολύ ε, θερμές αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία και τα καλοκαίρια που περνούσα στις παραλίες, ε, παρθένα νερά, πολύ ωραίες αναμνήσεις ε, και όσο μεγαλώνω τόσο τις θεωρώ πιο σημαντικές αυτές τις αναμνήσεις. Είδα όμως και αρνητικά να συμβαίνουν πίεση στα οικοσυστήματα και στους διάφορους πόρους. Έχω ακούσει φίλους μου ψαράδες να παραπονούνται ότι δεν έχουν τόσα ψάρια να ψαρέψουν. Είδα επίσης ε, να γίνεται λόγος για την αλλαγή του κλίματος, την υπεραλίευση, την ρήπανση. Ε, μπαίνουν στο προσκήνιο αυτές οι συζητήσεις και όλα όσα συμβαίνουν σήμερα μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι πράσινο και γαλάζιο πρέπει να συμβαδίζουν. Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, πριν πέντε χρόνια περίπου, εργάστηκα σκληρά για να περάσω αυτό το μήνυμα και για να δημιουργήσω ένα συνασπισμό για υγιείς παραγωγικές θάλασσες και ωκεανούς. Είτε εδώ, ε, στη χώρα μου, είτε στο εξωτερικό. Συμμαχία από ακτιβιστές, πολιτικούς, επιστήμονες, ε, πολίτες, νέους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει το μέλλον που θα κληρονομήσουν μια μέρα από εμάς αυτό το γαλάζιο πλανήτη. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που βλέπω να είναι γεμάτη σήμερα η αίθουσα γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τη σημασία των ωκεανών, για την οικονομία, για το κλίμα μας, αλλά πάνω απ' όλα για την επιβίωσή μας πολύ απλά. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τα επιτεύγματα της Ένωσης τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρώτα απ' όλα Έχουμε κανόνε που περιορίζουν τη χρήση των πλαστικών μια χρήση. Έχουμε στόχου, ανακύκλωση δεσμευτικού. Όλα αυτά καθιστούν την Ένωση παγκόσμιο πρωταγωνιστή για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Δεύτερον, έχουμε ορίσει πάνω από το 10% ε, των θαλάσσιων περιοχών, των ακτογραμμών, ω προστατευόμενε θαλάσσιες περιοχέ δύο χρόνια πριν από την λήξη τη Διεθνού προθεσμία του 2020. Και αυτό συνεισφέρει στο να έχουμε καλή κατάσταση περιβαλλοντική για τους ωκεανούς μας σύμφωνα και με το ενιαίο θαλάσσιο πλαίσιο, τη σχετική οδηγία. Τρίτον, πιέζουμε για πιο βιώσιμη αλληλεία και αυτό αποδίδει σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αλία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, στην καλύτερη εδώ και δεκαετίε. Τα αλλιεύματα, ε, τα οποία αλλιεύονται σε βιώσιμα επίπεδα, έχουν διπλασιαστεί. 51 ήδη φέτο σε σχέση με 27 όταν αναλάβαμε καθήκοντα και 5 μόλι πριν από 10 χρόνια. Τέταρτον, αναδυόμενοι τομεί ε, τη ε, βιώσιμη θαλάσσια οικονομία είναι πλέον στο προκείμενο. Η ενέργεια του είναι ένα καλό παράδειγμα. Και έχει λάβει και σημαντική χρηματοδότηση για έρευνα, για πειραματισμό. Είναι ένα τομέα ταχαίω αναπτυσσόμενο και περνάμε στην φάση πρώτη ε, διάθεση στο εμπόριο. Επίση, υπάρχουν και άλλες καινοτόμες θαλάσσιε επιχειρήσει ε, και κλάδοι που θα ε, βοηθηθούν από την πλατφόρμα που θα δρομολογήσουμε αργότερα φέτο. Επίση, τα δύο τελευταία χρόνια επενδύσαμε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα, τη θαλάσσια έρευνα συγκεκριμένα. Παραδείγματι το μικρό του τους ενδεχόμενους κινδύνους ε, των μικροπλαστικών για τη θαλάσσια ζωή αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. Και γνωρίζω πως ο συνάδελφός μου, Κάρλος Μοέδας, θα πει περισσότερα για το θέμα αυτό σε λίγο. Δεν έχουμε όμως ε, περιορίσει τις φιλοδοξίες μας μόνο στην Ευρώπη γιατί ε, η ωκεανή είναι μια κοινή ευθύνη παγκόσμια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να αναγγείλω ότι μόλις δημοσιεύσαμε την πρώτη έκθεση προόδου για το τι έχει πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία καταγράφει το τι πετύχαμε από τότε που εγκρίναμε το θεματολόγιο για μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση των ωκεανών τον Νοέμβριο του 2016. Πρόκειται για ένα θεματολόγιο με 50 δράσει ε, που έχει αναζωογονήσει τη διεθνή συνεργασία. Είναι ένα θεματολόγιο που σφυριλατεί και παγιώνει την φήμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενό ε, ως ένα εταίρο αξιόπιστο. Παρέχουμε τεχνική βοήθεια, χρηματοδότηση για βιώσιμη δράση και οικονομική ανάπτυξη και είμαστε στην κορυφή. 600 εκατομμύρια ευρώ περίπου έχουμε ε, διαθέσει για τη στήριξη της αλίας και της ηχθειοκαλλιέργειας, για την υποστήριξη των περιοχών που βασίζονται στην αλία, για πιο καθαρές θαλάσσιες μεταφορές και για βελτίωση των λιμενικών υποδομών και της θαλάσσιας ασφάλειας στις χώρες εταίρους. Βοηθήσαμε σημαντικές αλληλευτικές δυνάμεις να βελτιώσουν τα συστήματα ελέγχου τους ώστε να μπορεί να καταπολεμηθεί καλύτερα η παράνομη αλία και πιο αποτελεσματικά ε, με το σύστημα της χίτρινης και της ε, κόκκινης κάρτας. Επίσης έχουμε διμερείς εταιρικέ σχέσεις ε, με φορείς σημαντικούς χώρες όπως η Κίνα, ο Καναδάς. Επίσης έχουμε ολοκληρώσει μια νέα συμφωνία με την Αρκτική για να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη εμπορική αλληλεία στον Αρκτικό ωκεανό στα ανοιχτά. Επίσης, ε, προωθούμε βιώσιμε ε, γαλάζιες οικονομίες και εντός ε, της Ευρωπαϊκής αλλά και σε άλλες τρίτες χώρες νησιωτικέ μέσω των αρχών της θαλάσσιας βιώσιμης οικονομίας για να προωθήσουμε βιώσιμη οικονομία στο ωκεανούς. Επίκυνται ευρωεκλογέ. Είμαι πεπισμένος περισσότερο από ποτέ ότι οφείλουμε να πούμε στους πολίτες τι κάνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει για τις τοπικέ κοινότητε, για τις οικογένειε, για το μέλλον τους. Και ο ωκεανό είναι το καλύτερο μέρο να ξεκινήσει κανεί. Όπω ε, ε, αρέσει και λέει άλλωστε και ο πρόεδρο Γιούγκερ, θέλουμε να είμαστε μεγάλοι στα μικρά πράγματα. Και τι πιο μεγάλο υπάρχει από τον ωκεανό. Ε, περάσει λοιπόν αυτό το μήνυμα προς τα έξω για να μάθει ο κόσμος ε, πώς εργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις ε, θαλάσσιες περιοχές ε, για ένα γαλάζιο πλανήτη, τον δικό μας γαλάζιο πλανήτη για το μέλλον μας, το δικό μας μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ Καρμένου. Στη συνέχεια μπορώ να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Ξέρετε ότι έχουμε τρία θεσμικά όργανα, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα η Ρουμανία έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Αντριάννα Πέτκου είναι αναπληρώτρια υπουργό Υδάτων και Δασών. Νομίζω περισσότεροι χρειαζόσαστε ακουστικά διότι η προσκεκλημένη μας θα μιλήσει στα ρουμανικά. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ, Γεζίνε. Κύριοι Επίτροποι, κύρια Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διοργάνωση αυτής της εξαίρετης διάσκεψης μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών μας να σώσουμε τους ωκεανούς και τις ανοιχτές θάλασσες έτσι ώστε να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτώμεθα. Θεωρούμε ότι οι ωκεανοί και οι ανοιχτές θάλασσες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Οι ωκεανοί μας δίνουν χώρο, πόρους, ενέργεια και τροφή για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό οι ωκεανοί και οι θάλασσες μπορούν να εξαλείψουν τη φτώχεια προσφέροντας νέες θέσεις βιώσιμες εργασίες. Αυτό όμως το ο βασικό στοιχείο ρύθμισης σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της βιωσιμότητας για τους ωκεανούς. Αυτό αποτελεί υποχρέωσή μας, έτσι ώστε να μην ακολουθήσουν φθήνουσα πορεία οι ωκεανοί, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον που είναι κλειδί για τις πολιτικές μας. Εμείς προσδίδουμε μεγάλη, σημασία στην προστασία των θαλασσών. Για μας η μαύρη θάλασσα προσδίδει πόρους και αποτελεί ένα εξαίρετο οικοσύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ανθρωπογενείς πιέσεις από 200 δις ανθρώπους ως προς την παράνομη δράση τους, καθώς και τη μόλυνση της θάλασσας. Θα πρέπει να προωθήσουμε την βιώσιμη αλληλεία και να διασώσουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης των παρακτήων περιοχών. Παρά τις εθνικές μας προσπάθειες, η προστασία των θαλασσών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την περιφερειακή προσέγγιση που βασίζεται στη σύμβαση για την προστασία της μαύρης θάλασσας κατά της μόλυνσης. Γι' αυτό θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει εταίρος και αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πολλές πιέσεις ως προς την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά αποτελούν μόνιμη απειλή του θαλάσσιου περιβάλλοντος γιατί δεν υπάρχει σωστή διαχείριση θαλάσσιων αποβλήτων. Το θέμα των θαλασσίων αποβλήτων είναι περίπλοκο λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα καθώς και των ιδιοχαρακτηριστικών των θαλάσσιων περιοχών. Η επίλυση αυτών των θεμάτων σημαίνει προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό οι περιφερειακές συμβάσεις έχουν μεγάλη σημασία για την εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών στους ανοικτούς ωκεανούς. Η σύμβαση που αφορά τη Μαύρη Θάλασσα αναφέρεται στην ε, καταπολέμηση των θαλασσίων αποβλήτων και οι όμορες περιοχές καταβάλουν επίσης πολλές προσπάθειες. Η αύξηση των ε, πλαστικών θα πρέπει να καταπολεμηθεί, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα συλλέξουμε μέσα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Έχει μεγάλη σημασία η αποθήκευση, διακίνηση και η ανακύκλωσή τους. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αποτεφρώνονται αλλά να ανακυκλώνονται τα πλαστικά. Θα πρέπει η ανακύκλωση να είναι σημείο κλειδί για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Να επικεντρωθούμε στη γενική πρόληψη ως προς τα απόβλητα και τη σωστή διαχείρισή τους. Γι' αυτό προβάλλουμε και εταιρικέ σχέσεις. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την κατανάλωση σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη μόλυνση από τα πλαστικά και μικροπλαστικά, αυτό το θέμα θα απασχολήσει και το άτυπο συμβούλιο στις 20 και 21 Μαΐου στο Βουκουρέστι. Επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να προγραμματίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις οικονομικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες καθώς και να έχουμε συμμετοχή του κοινού. Να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές που οδηγούν στην θέρμανση των ωκεανών και έχουν επίπτωση στις παράκτιες περιοχές. Η Ρουμανία έχει προβάλει ένα master plan για την προστασία των παρακτίων περιοχών της Μαύρης Θάλασσας, έτσι ώστε να σταματήσει και η διάβρωση των ακτών. Και αυτό αφορά και τη βιωσιμότητα των οικισμών κοντά στη θάλασσα. Επίσης, το Δέλτα του Δούναβη μας έχει απασχολήσει μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης αυτής της ε, μεγάλης ε, λεκάνης απορροής και αυτό αφορά και τα παράκτια ε, ύδατα. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα θρεπτικά στοιχεία διατροφής που υπάρχουν στον Δούναβη και στην λεκάνη του Δούναβη που μειώνονται λόγω του ευτροφισμού. Θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για το οικοσύστημα αυτό της Μαύρης Θάλασσας με βάση την οδηγία πλαίσιο της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο περιβάλλον. Υπάρχει μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση των ωκεανών. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί για την βιωσιμότητα των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών για να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία της βιοπικιλότητας. Είμαι πεπισμένη ότι αυτή η διάσκεψη θα επιτρέψει να επιτελεστεί πρόοδος μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης χρήσης ωκεανών και θαλασσών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό ο Ρουμανικό οδικός χάρτη είναι πολλά υποσχόμενος σε συγχαίρω. Αν κάνετε όλα αυτά που έχετε προγραμματίσει, θα βοηθήσετε πολύ στην υγεία των ωκεανών. Επόμενος ομιλητή, ο Επίτροπο Κάλλος Μουέντας, που είναι αρμόδιο για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία. Και, ε, όπως ξέρετε, ήδη έχουμε πει ότι 500 εκατομμύρια θα πάνε σε ειδικά προγράμματα έρευνα, Αλλά θα συμφωνείτε, κύριε Πίτροπο, ότι θα έπρεπε να είναι και περισσότερα, έτσι δεν είναι, θα ήταν καλύτερα. Έχετε τον λόγο παρόλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και πρώην συνάδελφοι Καρμένου και Μαρία, και κάθομαι εκεί που ε, ήσασταν κι εσείς. Κάθε μέρα, δηλαδή το γραφείο μου είναι εκεί που ήσασταν εσείς, οπότε καταλαβαίνω και το δικό σας το καθήκον. Κοίταζα το κοινό και βλέπω τόσους νέους Νομίζω ότι η δική σας γενιά, η νεότερη γενιά, είναι τόσο τυχερή. Είστε η γενιά που θα δει η επιστήμη να κάνει καταπληκτικά πράγματα, όπως και η τεχνολογία. Θα δείτε θεραπείες ε, για ασθένειες που ακόμη σήμερα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε. Θα δείτε η κβαντική υπολογιστική να αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών. Αλλά θα αντιμετωπίσετε και μεγάλες προκλήσεις. Και η πρόκληση που συζητάμε σήμερα εδώ είναι μία από τις κυριότερες που έχετε ενώπιόν σας. Οπότε απευθύνομαι σε εσά για να σας πω ότι μετά από πέντε χρόνια εργασίας ως Επίτροπος και ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, συναντώντας υπουργούς, πρωθυπουργούς, ε, σημαντικές προσωπικότητες. Όμως, ε, όταν σκέφτομαι την πενταετία που πέρασα, κυρίως θυμάμαι τους νέους που συνάντησα και ένα από τα άτομα που με ενέπνευσαν είναι ένας ε, ιδιαίτερα νέος. Ένας νέος που λέγεται Boyan Slad. Ο Boyan Slad είναι Ολλανδός. Όταν ήταν 16, φανταστείτε το, μόλις 16, πήγε στην παραλία στην ε, Μεσόγειο και είδε πολλά πλαστικά σκουπίδια και είπε «Μα τι έσχος είναι αυτό, κάτι πρέπει να κάνω». Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της γενιάς σας και της δικής μου. Η γενιά σας κάνει πράγματα. Καταλαβαίνει ότι ο ρόλος της δεν είναι απλώς να βρει μια δουλειά, να πάει στο πανεπιστήμιο και τέτοια. Είναι να αλλάξει τα πράγματα. Και η ιστορία του Boyan Slad, η ιστορία της γενιάς σας, είναι ότι ένας νέος, 16 ετών, να θεωρεί ότι είναι δουλειά του να καθαρίσει τις παραλίες και τους ωκεανούς. Και ε, ορισμένοι του λένε, κοιτάξτε, ε, υπάρχουν τόσες τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να καθαρίσουμε τους ε, ωκεανούς. Και ο Μπόιαν λέει, μα αυτοί απλώς ανακυκλώνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην μπαίνουν τα πλαστικά στον ωκεανό. Και εφήβρε μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιεί τα ρεύματα στη θάλασσα για να γίνει κάτι που πολλοί μηχανικοί και πολλοί άλλοι ειδικοί το συζητούσαν αλλά εξέταζαν τα θέματα με συμβατική άποψη. Ο Μπόγιαν προτείνει μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Και αν επιτύχει σε αυτό που επιδιώκει, και βεβαίω ορισμένοι αμφιβάλλουν αν θα επιτύχει, αν είναι σωστή αυτή η τεχνολογία. Αλλά δύο πράγματα που έκανε είναι θεωρώ πολύ σημαντικά. Πρώτον, θεωρεί ότι είναι καθήκον του να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, αποστολή του. Αναλαμβάνοντας από την αποστολή, κατάφερε να ε, βάλει τη συζήτηση αυτή στο επίκεντρο της προσοχής της κοινή γνώμης. Πριν από 15 χρόνια, αν σκεφτούμε πώς ήταν η συζήτηση, θα καταλάβετε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, ε, μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση στην κοινή γνώμη, αλλά η κατάσταση των ωκεανών δεν έχει αλλάξει. 8 εκατομμύρια τόνους πλαστικά μπαίνουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Αλλά η γενιά των παππούδων μου είναι μια γενιά όπου δεν υπήρχαν καθόλου πλαστικά. Οπότε, οι νέοι το καταλαβαίνουν καλύτερα, ότι τώρα 8 εκατομμύρια 8, ε, ε, εκατομμύρια τόνοι μπαίνουν τόσο ε, κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Δηλαδή κάθε χρόνο πάει ο καθένας μας, είναι σαν να πηγαίνει ο καθένας μας κάθε μέρα στην παραλία και να πετάει τρεις πλαστικές σακούλες στη θάλασσα. Ο Μπόγιαν Σλάτ είναι αυτός που κατάφερε οι άνθρωποι να το εξετάσουν. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή συζητούσα με τα παιδιά μου και άκουσαν ε, κάποιες συζητήσεις που κάναμε εδώ για την προστασία των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων των ε, πολιτών. Τα παιδιά μου δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ γι' αυτό. Μια μέρα μου είπαν, μα μπαμπά, έχουμε κάποιον YouTuber, ο οποίος μας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να σταματήσει το ίντερνετ. Και επειδή έρχονται σε επαφή διαφορετικά με το YouTuber από ότι έρχονται σε επαφή με εμένα ε, επηρεάστηκαν από αυτά που έλεγε. Νομίζω ότι ο Μπόγιαν Σλάντ έχει διαφορετικό τρόπο επικοινωνία με τους νέους. Οπότε, προσπαθούμε στον τομέα αρμοδιοτήτων μου να εξετάσουμε τη δουλειά του Μπόγιαν Σλάντ για να τη μιμηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν γίνεται. Δημιουργήσαμε τις αποστολές για την Ευρώπη, έτσι τις ε, ονομάσαμε και θα ήθελα μία από τις αποστολές να είναι για αντιμετώπιση των προβλημάτων των ωκεανών. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι γενικόλογοι να πούμε ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα θέματα των ωκεανών. Πρέπει να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα στους συμπολίτε μας. Πρέπει να τους πούμε τι θα κάνουμε, πώς θα καθαρίσουμε τους ωκεανούς. Και αυτός είναι διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας. Το είπε και ο συνάδελφός μου, ο Καρμένο. Έτσι χρειάζεται να επικοινωνήσουμε τη γενιά σας. Άρα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας να μας πείτε πώς να αλλάξουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική. Και η συγκυρία είναι κρίσιμη, διότι επίκυνται οι ευρωεκλογέ. Ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ όμως. Όταν ήρθα στις Βρυξέλλες το 2014, η κατάσταση ήταν εντελώ διαφορετική. Είχαμε τα προβλήματα των ψευδών ειδήσεων, είχαμε ορισμούς που λέγανε ότι οι ειδικοί δεν μας βοηθάνε. Ενώ τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τη γνώμη σας, αλλά αυτό εξαρτάται από εσά. Εσείς πρέπει να πείτε στους πολιτικούς τι θέλετε, τι επιδιώκετε. Και αυτό βλέπω κάθε Παρασκευή που είμαι στο γραφείο μου να συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί ποια είναι τα σημαντικά θέματα. Ότι δεν αρκεί να λένε οι πολιτικοί ότι κάτι θα κάνουν. Πρέπει να τους πιέσετε. Πώς θα καθαρίσετε τους ωκεανούς, ε, πότε θα το κάνετε, με ποιες τεχνολογίες, ποιος θα τον αναλάβει. Γιατί σε τελευταία ανάλυση εξαρτώμεθα από τους ωκεανούς. Περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε. Η Σίλβια Ρέλ, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, είπε και καταλήγω ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε θαλάσσια όντα. Δεν ζούμε μέσα στη θάλασσα, είπε, αλλά εξαρτώμεθα από τους ωκεανούς σαν να ζούσαμε μέσα στο νερό. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας πω ως μήνυμα. Ότι είμαστε εδώ, μπορείτε να βασιστείτε σε μας, θα ακούσουμε τα αιτήματά σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στην επόμενη περίοδο, όπως κάναμε και σε αυτή την περίοδο. Και θέλω να, ε, να συγχαρώ τον συνάδελφο Καρμένου και το Κοινοβούλιο, την κυρία Μάισνερ, Κάναμε πολλά νομίζω. Αλλά δεν ενημερώσαμε, δεν τα παρουσιάσαμε σωστά στην κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και πραγματικά το νιώθουμε πόσο σας συναρπάζουν οι Δεν ξέρω, ίσως ε, επειδή είστε από την Πορτογαλία όπως και Επιτρόπος ε, Καρμένου Μπέλα από τη Μάλτα. Ε, εγώ θέλω να αναφέρω την Μαρτσέλα Χάνς, γιατί αναφερθήκατε εσείς σε ένα Ολλανδό. Είναι φοιτητρία από το Άχεν, ε, μπορεί να μην την γνωρίζετε. Την ανέφερα όταν έκανα την εισαγωγή μου ομιλία. Ίσως να έχει βρει έναν τρόπο να ξεφορτωθούμε τα πλαστικά της αρέσει να κάνει καταδύσεις και ε, πραγματικά ε, όταν είδε πόσο πλαστικό υπάρχει μέσα στη θάλασσα είπε δεν μου αρέσει αυτό θέλω να το αλλάξω και έτσι δημιούργησε μια πλατφόρμα μαζί με κάποιους ε, μηχανολόγους, μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο με την ιδέα ότι τα μικροπλαστικά με τα κύματα και τα ρεύματα ενώ είναι στην επιφάνεια κανονικά μπορούν να βουλιάξουν στο βυθό. Ε, οπότε αν κάπως με ένα είδος πλατφόρμας που μπορούμε να κάνουμε τα νερά να γαλινέψουν και μπορούν να ανέβουν να επιφάνεια τα πλαστικά, θα μπορούσαμε ίσως να τα ε, περισλέξουμε πιο εύκολα. Είναι ενδιαφέρουσες ιδέες σαν αυτή του Μπόγιαν Σλάντ ή ε, αυτή της ε, φοιτήτρας για την οποία σας ε, μίλησα εγώ. Επειδή μιλήσατε και για την κοινωνία, αυτό το θεωρώ και εγώ σημαντικό. Φυσικά και εμείς είμαστε σημαντικοί, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, αλλά η κοινωνία είναι αυτή και αυτό με κάνει να ε, σας συστήσω και την επόμενη μα ομιλητρία Ζενεβιέβ Πόνς από το Γραφείο των Βρυξελών του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ, από τι ομιλητέ που εκπροσωπεί την κοινωνία ακριβώ. Ζενεβιέβ, έχεις το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ και Ζήνε. Ευχαριστώ και τον Καρμένου για την πολύ σημαντική αυτή πρόκληση που μου απευθύνεται να μιλήσω. Σήμερα θέλω να σας καλησπερίσω όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, κυρίως όμως τη νέα γενιά που εκπροσωπείται τόσο καλά εδώ. Είναι προνόμιο για μένα να απευθυνθώ στην συνέλευση αυτή και είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Η παρουσία μας εδώ είναι άκρος επίκαιρη λίγες ημέρες μετά από τη διαδήλωση ενός εκατομμύριου χιλιάδων νέων ε, που διαδήλωσαν κατά της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δράσουμε και εμείς. Αρκετές ε, ε, είναι οι συμφωνίε και δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει και σίγουρα αυτό θα μα κρατήσει ε, σε δουλειά για δεκαετίες ολόκληρες. Ο ωκεανός είναι η καρδιά του πλανήτη και του κλίματος. Είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη. Ουσιαστικά μας προσφέρει την αναπνοή μας, τον αέρα που αναπνέουμε. Δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται καθημερινά στους ωκεανούς για την επιβίωσή τους. Η προστασία τον ωκεανό λοιπόν δεν είναι επιλογή, σημαίνει επιβίωση. Και αν ο ωκεανός ε, είναι υπεύθυνο για την υγεία του πλανήτη, τότε ο νότιος ωκεανό είναι η καρδιά ε, του ωκεανού. Μιλάμε για ισχυρά πολικά ρεύματα ε, γύρω από την Ανταρκτική που ουσιαστικά τροφοδοτούν τον ωκεανό με πλούσια θρεπτικά ε, συστατικά νερά. Η θαλάσσια βιοπικιλότητα μας ε, παρέχει έμπνευση, οξυγόνο, τρόφιμα. Η πηγή της είναι ο Νότιος Ωκεανός. για όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, πάντοτε με ε, τραβούσε με ήλικε ο ωκεανός. Ε, έζησα την παιδική μου ηλικία στην Τινησία, δίπλα στη θάλασσα και μερικές από τις ε, πιο ε, πρώιμες μνήμες μου είναι ο καιρός που περνούσα με την οικογένειά μου στην Ακροθαλασσιά. Έκτοτε έκανα καταδύσεις ε, σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο και πάντοτε με κατέπλησε η ομορφιά του ωκεανού, αλλά με ανησυχούσε ταυτόχρονα βαθύτατα η υποβάθμισή του. Είτε στη χώρα μου, την πατρίδα μου, όπου οι χελώνες πεθαίνουν επειδή έχουν καταπιεί πλαστικό, ή στο κοραγενές τρίγωνο, όπου υποβαθμίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς η βιοπικιλότητα. Όταν ήμουν επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΒΒΕΦ, αποφάσισα για όλους αυτούς τους λόγους να ενισχύσω τη δράση μας ε, για την προστασία των ωκεανών και πιο πρόσφατα όταν ε, με είχαν προσκαλέσει να συμμετάσχω σε μια ομάδα ε, υψηλού επίπεδου άσκησης επιρροής για τη στήριξη του Νότιου Ωκεανού δεν δίστασα ούτε μια στιγμή. Είμαστε η Ανταρκτική 2020, μια ομάδα ε, έξι εξαμελής από όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον Νότιο ωκεανό, τα νερά που ε, βρέχουν την Ανταρκτική. Είναι πάρα πολύ πλούσιο περιβάλλον αυτό του Νότιου ωκεανού, πιγκουίνι, φάλαινες, φώκες, ε, σε ένα οικοσύστημα που βασίζεται ε, σε πολύ μικρό αλλά πάρα πολλών ειδών κρύλ βιοπλακτών ε, και χιλιάδες επιστήμονες ε, μελετούν αυτό το κρύλ. Το 1959 στην, στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου αποφάσισαν παρόλα αυτά οι χώρες να θεωρήσουν την Ανταρκτική ένα χώρο ειρήνης και επιστήμης. Ήταν μια πολύ γενναία πράξη ε, και δείχνει ότι τελικά μπορούν ε, οι ε, πολιτικές να επηρεαστούν από την Ήπειρό μας και τα νερά της. Τα 25 μέλη της Κομισιόν για τις Επιτροπής για τη Διατήρηση των Πόρων της Ανταρκτικής έχουν δεσμευτεί ακριβώς για αυτό το σκοπό. Να προστατεύσουν δηλαδή τον Νότιο Ωκεανό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος αυτής της Επιτροπής. Και όλα δείχνουν ότι η καλύτερη δυνατή προστασία του Νότιου Κιανού είναι με τη δημιουργία ε, προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών μεγάλης κλίμακας αυτό μα ζητούν οι νέοι, να προστατεύσουμε τον Νότιο ωκεανό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει δύο σημαντικές μεγάλες προστατευόμενε περιοχές στον Νότιο ωκεανό, την Ανατολική Ανταρκτική και την θάλασσα Βέντελ. Η ε, πρόταση για την Ανατολική Ανταρκτική μιλάμε για ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρώτα έγινε από τη Γαλλία το 2011 και περιμένουμε πολύ, ήδη έχουν περάσει χρόνια. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να προστατεύσουμε τώρα τον Νότιο ωκεανό και καθυστερούμε. Έχουμε προβλήματα όχι λόγω έλλειψη σπόρων, τεχνολογία ή επιστήμη, αλλά γιατί ε, την δράση αυτή την ε, επηρεάζουν ε, τα γεωπολιτικά και εθνικά συμφέροντα που θολώνουν αυτά τα παρθένα νερά. Τι περιμένουμε λοιπόν για να δράσουμε. Το 2015 ο Μπαράκ Ομπάμα έδειξε ότι ναι, είναι μεν δύσκολο να προστατεύσει κανεί τον μπορεί όμω να γίνει. Είχε μιλήσει λοιπόν ο Μπαράκ Ομπάμα ε, με τον ηγέτη της Κίνας, τον Xi Jinping, και κατάφερε να υποστηρίξει η Κίνα τη δημιουργία μιας θαλάσσας πρωτευόμενης προχής στη θάλασσα Ρος, στον Νότιο Ωκεανό. Και την επόμενη χρονιά με την ρωσική αυτή τη φορά υποστήριξη επετέχθη συνένεση για την ε, χάραξη των προσδιορισμών της μεγαλύτερης στον κόσμο θαλάσσιας πρωτευόμενης περιοχής στον πλανήτη τώρα να δράσει φέτο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία. Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική. Ε, ο Καρμένου Βέλα, η Φεντερίκα Μογκερίνο, ο Ντόναλτ Τούσκ, έχουν δεσμευτεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσει τον Νότιο Ωκεανό. Ο ε, Xi έρχεται στην Ευρώπη, ε, στο Μονακό αρχικά, μετά στο Παρίσι και ενδεχομένως να μεταβεί και στις Βρυξέλλες εν συνεχεία. Το σημερινό μου μήνυμα, το μήνυμα από την ομάδα Ανταρκτική 2020, το μήνυμα από τους ε, νέους που είναι εδώ παρόντες σήμερα είναι πρέπει να δράσουμε τώρα για το κλίμα και για την απώλεια της βιοπικιλότητας. Και για να το πετύχουμε πρέπει να προστατεύσουμε τον Νότιο Κιάνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζενεβιέβ. Νομίζω ότι όλοι θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την Ανταρκτική, μεταξύ άλλων. Τώρα, ε, έχουμε και την Ντανιέλα Φερνάντες, δεν μπόρεσε όμως να μεταβεί. Έχουμε δύο άλλους εκπροσώπους, νέους, ε, Νίλε Φαν Χόιβέγγεν, που ε, είναι εκπρόσωπος ε, της ε, Ολλανδόφωνης κοινότητας του Βελγίου και ο Σεμπαστιάν Βιλμάρτ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της ε, γαλλόφωνης, του Γαλλόφωνου Συμβουλίου Νεότητας του Βελγίου. Η Νέλε έχει το λόγο πρώτο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Εδώ εκπροσωπούμε τα συμβούλια του Βελγίου νεότητας και θέλουμε επίσης να θίξουμε ένα ζήτημα ύψης της σημασίας, το φυσικό περιβάλλον μας, το σπίτι μας, το μέλλον μας, την Προηγούμενη εβδομάδα πάνω από ένα εκατομμύριο νέοι βγήκαν στους δρόμους έτσι ώστε να ληφθούν θαραλέα μέτρα σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Δεν πρόκειται για τα παιδιά μας ή για τις επερχόμενες γενναίες. Πρόκειται για μας, για το δικό μας μέλλον. Η υγεία και η ευημερία της ανθρωπότητας σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον μας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη ε, έχει θερμάνει τους ωκεανούς ανά μία ατομική ε, βόμβα το δευτερόλεπτο. Δυστυχώς ε, χάνεται, πεθαίνει η θαλάσσια ζωή. Αν δεν σταματήσουμε τις εκπομπές, η Αρκτική θα είναι κατά πέντε βαθμούς ε, θερμότερη μέχρι το τέλος του αιώνα. Μιλάμε για ανεκτά επίπεδα έτσι ώστε ο πολιτισμός να επιβιώσει. Μέχρι το 2100 ο πληθυσμός θα έχει αλλοιωθεί σε σχέση με σήμερα. Σκεφτείτε ποια θα είναι μία εικόνα δορυφόρου του μπλε πλανήτη που δεν θα είναι πλέον μπλε. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις κοραλιογενείς εκτάσεις που αποτελούν ένα 25% της θαλάσσιας ζωής. Όμως το IPCC δείχνει ότι με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό θα, χαθούν, θα χαθεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο κοραλιογενής ευλάστησης. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται κατά πολύ στις χώρες του ΩΣΑ. Κάτι το οποίο ε, δείχνει ότι το δικαίωμα στο ε, νερό πρέπει να υπάρχει, καθώς και να απαγορευτεί η γλυφοσάτη. Πώς ε, δεν μπορείτε να είσαστε δραστήριοι. Η Ευρώπη έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά αυτό δεν θα μας περισσώσει. Μιλάτε για την γαλάζια οικονομία. Αυτός ο νέος όρος είναι μία, δεν θα είναι δεν θα πρέπει να είναι μία σήμανση. Θα πρέπει να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρακτικές που σχετίζονται με τους ωκεανούς. Δεν θα πρέπει να προφήσουμε δράσεις που είναι επιζήμιες στο περιβάλλον. Θέλουμε να δεσμευτείτε όλοι προς αυτό. Οι ωκεανοί είναι ένα νέο ελντοράντο. Είναι πόροι, είναι αναψυχή είναι ε, θρεπτικά συστατικά μεταξύ πολλών άλλων, από τα οποία εξαρτώμαστε πλήρως και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Η προστασία των ε, οικοσυστημάτων των ωκεανών είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές για την επιβίωση βιώσιμων οικοσυστημάτων για τους ανθρώπους, τη φύση και τις επιχειρήσεις. Σας παρακαλούμε να το κάνετε σοβαρά σας προτρέπουμε να ισχύσουν οι κανόνες αλίας στον τομέα αλίας για να μην γίνεται χρήση πλαστικών στις ε, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. η παγκόσμια διακυβέρνηση των ε, ωκεανών δεν θα αρκέσει από μόνη της. Η καταπολέμηση... τη αλλαγής. Η καταπολέμηση της φτώχειας ε, είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Πρέπει να υπάρξει διαρθρωτική δράση. Πρέπει να επαναδιαμορφωθεί το σύστημα ανάλογα με την φυσική, φυσιολογική πραγματικότητα με την φυσική πραγματικότητα του πλανήτη και των συμπολιτών. Το θέμα δεν είναι να καθαρίσουμε μόνο του ωκεανού. Είναι να σταματήσουμε να του μολύνουμε Ξέρουμε την κατάσταση. Ξέρουμε και τις λύσεις. Αλλά ε, τα παραβλέπετε όλα αυτά. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια θέματα. Ε, πρέπει να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα της φορολογικής δικαιοσύνης όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φόρο για τον άνθρακα. Θα πρέπει η Κομισιόν ε, να καταπολεμήσει επίσης την ε, φόρο αποφυγή κατά προτεραιότητα στην επόμενη θητεία και να θέσει ένα τέρμα στο φορολογικό ντάμπινγκ και τα κοινωνικά ζητήματα βέβαια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι γνώμονας στις ε, εν λόγω πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια διαφορετική θεώρηση για τα δημοσιοοικονομικά. Η χρηματοδότηση ε, να κρίνεται με βάση το πόσο συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή να επενδύουμε εκεί που μετράει. Δεν μιλάμε όμως μόνο για επιχορηγήσεις δημοσιοοικονομικά. Πρέπει να κατανοήσουμε το εμπόριο ε, ως ένα παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να έχουμε δυσανάλογη συγκέντρωση πλούτου ούτε διαιώνιση ανθιγυνών τρόπων ζωής. Για παράδειγμα, μπορούμε να υιοθετήσουμε τον δείκτη ανθρώπινη ανάπτυξη, που είναι ένα βασικό δείκτη επιτυχία και όχι απλά η ανάπτυξη με βάση το ΑΕΠ να είναι το κριτήριο. Πρέπει επίση το πολυμερέ εμπορικό σύστημα να μεταρρυθμιστεί στο πλαίσιο αυτό και οι κανόνε του ΠΟΕ, ώστε να λάβουν μεγαλύτερη προτεραιότητα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποια μικρά βήματα προηγουμένω, όπως η πρόταση για αύξηση του ενωσιακού προπολογισμού και των ταπανών για ε, το κλίμα κατά 25%, όμω αυτό δεν αρκεί. Είναι σαφές. διότι θα πρέπει να μετριαστεί η αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να δοθούν πόροι για την οικολογική μετάβαση. Για εβδομάδε, κατεβαίνει ο κόσμος ε, και διαδηλώνει. Άρα χρειάζεται συστημική αλλαγή, όχι κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν αιτήματα που σχετίζονται συγκεκριμένα με του ωκεανού. Ζητούμε όμω πέραν αυτού τη διαγενειακή δικαιοσύνη και την ισότητα να την θεωρήσετε σημαντική κατευθυντήρια γραμμή για τι πολιτικέ σε όλα τα επίπεδα. Οι επιστημονικέ μαρτυρίε, τεχνικέ λύσει, η κρίσιμη μάζα ε, είναι κάτι που το έχουμε. Το έχουμε επιτύχει. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να επιδειχθεί πολιτικό σθένος και είναι η τέλεια στιγμή χρονική να γίνει αυτό, διότι η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική. Το μέλλον μας είναι αυτό το οποίο παίζεται στην κυριολεξία. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ε, διαλέξετε το μέρος της ιστορίας στο οποίο θέλετε να είστε. Μπορούμε να εργαστούμε μαζί για να προστατεύσουμε το μέλλον ε, και των ε, νυν και των μελλοντικών γενιών. Ας είστε κι εσείς μέλος κομμάτι αυτής της Ευχαριστώ. Νέλε και Σεμπαστιά, ακούσαμε αυτά που μας είπατε, μας συγκίνησαν ιδιαίτερα και εν γέννη η συνεισφορά σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να μετατρέψουμε την πολιτική σε πραγματικότητα, αλλά προσπαθούμε. Λίγη λοιπόν τώρα η, εναρκτήρια, ε, η έναρξη της διάσκεψης θα πάμε για την οικογενειακή φωτογραφία έξω στο άτριουμ. Πριν όμως από την οικογενειακή φωτογραφία θα έχετε ένα νέο ε, πάνελ υπό τον Αλέν ε, Καντέκ. Δυστυχώς όμως άργησε η πτήση του και γι' αυτό η Ντάρια Μάτο θα αναλάβει το επόμενο πάνελ και θα ήθελα όλοι οι πάνελιστ στη συνέχεια να έρθουν να μας αντικαταστήσουν. Άρα τώρα θα πάμε για την οικογενειακή φωτογραφία και μερικοί θα επανέλθουν. Ο Ντάριο Μάτο θα είναι... Ο Γκάμπριελ Μάτο θα αναλάβει το πρώτο πάνελ το οποίο θα αρχίσει σε 10 περίπου λεπτά.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 Γεια σας, σας καλωσορίζω. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για δύο λόγους. Ακουστικά παρακαλώ, να τα χρησιμοποιήσετε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εγώ είμαι ένας από, τους 500, από τα 550 εκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν Ισπανικά. Άρα θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Το δεύτερο είναι γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα διερμηνέων ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Mi colega η συνάδελφος η Γκεζίνε Μάισνερ μας είπε ότι ο Αλέν Καντέκ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να προεδρεύσω σε αυτό το εξαιρετικό πάνελ ομιλητών. Ε, λυπούμεθα που δεν βρίσκεται εδώ ο Αλέν, αλλά θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες, τους εκπροσώπους, τους εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους μου, ευρωβουλευτές. Εφόσον άλλαξε λοιπόν η σειρά παρουσίασης, θα μιλήσω και εγώ στην πρώτη φάση συζήτησης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τρία τέταρτα του πλανήτη ε, αφορούν την, το νερό, δηλαδή απαρτίζονται από ύδατα και σε όγκο και σε ε, κυβικά. Πρόκειται για το 70% των υδάτων που απαρτίζουν τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο με 25 χώρες και περιφέρειες, θαλάσσιες περιφέρειες και βεβαίως αυτό περιλαμβάνει και τα Κανάρια νησιά που είναι απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή. Πέρα λοιπόν από την ε, νομιμότητα και τη θεμητότητα συμμετοχής μας θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στον αλληλευτικό τομέα τι εννοούμε όταν μιλάμε για διαχείριση των ωκεανών, διακυβέρνηση των ωκεανών, τι σημαίνει αυτό, τι προϋποθέτει. Θα ήθελα να σας μιλήσω, να σας σκιαγραφίσω τι σημαίνει καλή διακυβέρνηση των ωκεανών. Η καλή διαχείριση περιλαμβάνει και αφορά την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αλία δεν έχει σύνορα και αυτό ακριβώς σημαίνει και γι' αυτό υπάρχει κοινή αλλιευτική πολιτική. Άρα η διασυνοριακή διάσταση των ωκεανών δείχνει ότι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα, στο πιο ευρύ πλαίσιο αλλά και πιο περιορισμένο. Καλή διαχείριση επίσης σημαίνει σωστή συμμετοχή των οικονομικών φορέων. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω ιδιαίτερα. Θα πρέπει να ακούσουμε την επιστημονική κοινότητα της ΜΚΟ και ολόκληρο τον τομέα και θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να συμμετέχουν ε, δραστικά γιατί θα δράσουμε όχι για τους οικονομικούς φορείς αλλά με τους οικονομικούς φορείς. Το δεύτερον ε, αφορά την ανάγκη χρήσης εύκολων όρων που να αποτελούν επίκληση. Δηλαδή μιλάμε για εκφόρτωση, για χώρους εκφόρτωσης φόρτωσης και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Δεν πρέπει όμως να εμείνουμε στην ορολογία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι σημαίνουν όλα αυτά, ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα και να μην χρησιμοποιείται η δημαγωγία για το απόλυτο κέρδος, διότι αυτό θα μας πλήξει άμεσα. Οι θαλάσσιες ε, περιφέρειες, θαλάσσιες περιφέρειες, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιφέρειες αποτελούν χήμερα. Έχουν ευεργετήματα βεβαίως και αποτελούν ένα μέσον διαχείρισης αλλιευτικών δραστηριοτήτων και για μία προστασία των θαλάσσιων περιοχών, αλλά δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Πέμπτο σημείο. Δεν θα πρέπει να εντυπωσιάζουμε με όρους οι οποίοι είναι δυσνόητοι και δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Εδώ ε, αναφέρομαι στο MSY, το οποίο για πολύ καιρό απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, τους επιχειρηματίες, τους επιστήμονες και τους οικονομικούς φορείς. Και νομίζω ότι σήμερα καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να δούμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορούμε να το αποδώσουμε καλύτερα και να το θέσουμε σε εφαρμογή. Δηλαδή την μέγιστη αυτή βιώσιμη απόδοση. Μη χρησιμοποιώντας, μη χρησιμοποιώντας ε, περίεργους όρους. Επίσης υπάρχει ένας ε, άλλος όρος για την βέλτιστη χρήση των ωκεανών. Έχει μεγάλη σημασία η χρήση ε, των πόρων όπως προβάλλουν οι εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς. Μιλώ για τις ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, για την αρχή της βιοπικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη αποφάσεων στο μέα της διαχείρισης της αλίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε και να ενισχύσουμε τα ε, παγκόσμια μέσα που έχουμε ή περιφερειακά μέσα. Γιατί πολύ συχνά όταν οι προσπάθειες δεν αποδίδουν δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει νομοθεσία αλλά υπάρχει θέμα εφαρμογής του νόμου και αυτό σχετίζεται άμεσα με την αλληλευτική πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχουν ορόσημα και πλαίσια για τον ευρωπαϊκό αλληλευτικό στόλο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία εάν λάβουμε υπόψη τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της βιωσιμότητας ε, χρήσης του ε, στόλου μας, ο οποίος δεν πρέπει να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ηγετική θέση έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες και τις ε, προκλήσεις μέσα στα πλαίσια της βιωσιμότητας των πόρων. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την αλία και τον αλλιευτικό στόλο. Η υπεραλίευση, οι κλιματικές αλλαγές, καθώς και η παράνομη, αδήλωτη και άναρχη αλίευση. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες προσπαθήσαμε να απαλείψουμε αυτή τη μάστιγα μέσα στα πλαίσια της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τρίτες χώρες θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε τα αλλιεύματα, τα παράνομα αλλιεύματα να μην φτάνουν σε εμάς. Αυτό αφορά και το ένατο σημείο που είναι και το τελευταίο. Τι γίνεται σε σχέση με την υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την πρόκληση, πρόκληση στον τομέα της ηχθειοκαλλιέργειας, ιδιαίτερα όταν οι θάλασσές μας πλήττονται από τις θαλάσσιες μεταφορές και την εκμετάλλευση των πρώτων υλών, την μόλυνση των θαλασσών και τις κλιματικές αλλαγές. Για όλους αυτούς τους λόγους που είναι ε, ολίγιστοι σε σχέση με το σύνολο, θα πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση των ωκεανών. Η υγεία των ωκεανών έχει μεγάλη σημασία για την ανθρωπότητα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους διαχειριστούμε και να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους πόρους, να έχουμε καθαρούς ωκεανούς, ε, παραγωγικούς, ασφαλείς και υγιείς και προπαντός προστατευόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και τώρα θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδιοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Ο κάθε ένας από τους ομιλητές θα πρέπει να μιλήσει γύρω στα τέσσερα λεπτά. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην Εντάρ Ματσάδο που είναι καλός φίλος και Γενικός Διευθυντής στην ε, Γενική Διεύθυνση Αλίας και Θαλασσών. Ευχαριστώ αγαπητέ Γάμπριελ και αξιόλο, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε Βέλα, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι η συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης ε, μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Και σήμερα έχουμε τόσους νέους εδώ είναι επίσης κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας χαροποιεί. Νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση που λαμβάνει η χώρα εδώ στο Κοινοβούλιο είναι προήμιο σύστασης μιας επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Αλία και τους ωκεανούς. Νομίζω πως θα ήταν καλή ιδέα για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία και θα μας ωφελούσε όλους. Ευχαριστώ και συγχαίρω πολλούς ε, ευρωβουλευτές για τις προσπάθειες ε, που έχουν κάνει όπως, που έχουν κάνει, όπως η κυρία Ροντούστ και ο κύριος Σάντους για να είναι προτεραιότητα το θέμα αυτό για το Κοινοβούλιο. Όπως είπαν και διάφοροι ομιλητές ήδη προηγουμένως, οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι ζωτική σημασία ε, για όλους μας. Είτε μένετε κοντά στην παραλία είτε στο εσωτερικό μιας περιοχής είναι ζωτική για την ε, ζωή. Αλλά ε, υφίστανται πιέσεις, είναι ευαίσθητοι και χρειάζονται καλύτερη προστασία, φροντίδα, διαχείριση γιατί τους έχουμε παραμελήσει συνολικά ως παγκόσμια κοινότητα για πολλά χρόνια. Εμείς πριν από τέσσερα χρόνια, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρωτήσαμε τους Ευρωπαίους και διεθνεί εταίρου αν θεωρούσαν το διεθνές πλαίσιο για την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών το τρέχον τότε ήταν επαρκές και αποτελεσματικό σχεδόν όλοι απάντησαν όχι. Όχι επειδή το υπάρχον διεθνές πλαίσιο που έχει κέντρο τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο των θαλασσών δεν είναι σωστό, αλλά γιατί υπάρχουν κενά από πλευράς διεθνών ε, μέσων, ορισμένα είναι και ανεπαρκή και αναποτελεσματικά και δεν υπάρχει επαρκή συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων που έχουν δημιουργηθεί ε, όλα αυτά τα χρόνια. Και μόνο μέσω ισχυρής διεθνούς συνεργασίας που ε, στη σημερινή συγκυρία δεν είναι από τα πιο δημοφιλή ε, θέματα. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, παγκόσμια φύση των προβλημάτων αυτών. Μόνο ενωμένοι, μόνο συνεργαζόμενοι μεταξύ χωρών, μεταξύ, πέρα από σύνορα μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή για πρώτη φορά η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπό την ηγεσία του Επιτρόπου Βέλα και της ε, υπάτης εκπροσώπου Μογκερίνη. Μόνο λοιπόν που τότε, τότε που για πρώτη φορά υπήρξε ένα έγγραφο για την ε, παγκόσμια διαχείριση των ωκεανών, υπήρξε μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η ε, κατάσταση όπως ήταν και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, όπως είπε και ο Επίτροπος Βέλλα στην εισαγωγή του, δημοσιεύουμε για πρώτη φορά μια έκθεση προόδου για το σε τι βαθμό και με το τι τρόπο επιτύχαμε τους στόχους που θέσαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Στην έκθεση αυτή είναι προσβάσιμη. Θα δείτε ότι οι υποσχέσεις μας μετατρέπονται σε δράση και στον ε, αλληλευτικό τομέα. Λοιπόν, να τονίσω την πολύ σημαντική συμφωνία, καταρχάς, που συνήφθη τον περασμένο Οκτώβριο για μια νέα συμφωνία. Λοιπόν, μια νέα συμφωνία λοιπόν για την αλία στον, στην Αρκτική που απαγορεύει την ε, αλία για 16 χρόνια ε, στην κεντρική Αρκτική και ε, θα μπορούσε κατόπιν να επεκταθεί άλλα 16 χρόνια αυτή η απαγόρευση αν συμφωνήσουν οι συμβαλόμενοι. Δεύτερον, η Ένωση και όπως είπε ήδη ο Γκάμπριελ έχει πολεμήσει σκληρά για να εξαλειφθεί η παράνομη αλία και έχουμε αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό όργανο σε ενωσιακό επίπεδο που μας επέτρεψε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά πολλών ε, από τους εταίρους μας και να εξαλειφθεί η παρουσία αλλιευμάτων που έχουν αλλιευθεί παράνομα στις ευρωπαϊκές αγορές. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε εξάλλου ένα δίκτυο εταιρικών ε, συμφωνιών με τρίτες χώρες για θέματα αλλίας και αυτό βασίζεται στη νέα κοινή ελευτική πολιτική που θέτει στο κέντρο της προσοχής μας την βιωσιμότητα και την ε, υγεία των ε, ε, διαφόρων αλλιευτικών ειδών. Έχουμε συμφωνίες με τη Μαυριτανία, με το Μαρόκο, το Πράσο Κροτήριο, τη Γουνέα Μπισάου και επίσης σε αυτή τη νέα γενιά συμφωνιών υπάρχει και η διάσταση της θαλάσσιας οικονομίας, της βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης. Τέταρτον, προωθούμε μαζί με τους εταίρους μας την ανάπτυξη μια βιώσιμη γαλάζιας οικονομία. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά και ορισμένοι από του ομιλητέ στην ανακτήρια εκδήλωση το ανέφεραν. Πρέπει όμω να είμαστε προσεκτικοί. Η γαλάζια οικονομία πάντα πρέπει να εξετάζεται από την πλευρά της βιωσιμότητας για να αποφύγουμε τα λάθη που έγιναν για την ε, γεωργία και κτηνοτροφία. Τώρα, για να είναι αξιόπιστη σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε αξιόπιστες στο εσωτερικό μας. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω τις προσπάθειες που έχουμε μαζί με τα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο και με τον κλάδο της αλίας. Και έχει υπάρξει τρομερή πρόοδος, ούτως ώστε από θέματα να παραμείνουν σε υγιή κατάσταση. Ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τα αποθέματα σε τόσο βιώσιμο επίπεδο όπω τα έχουμε σήμερα. Με συγχωρείτε, ήδη ξεπέρασα το χρόνο μου. Θα σταματήσω εδώ. Αλλά θα έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε και περαιτέρω αν υπάρχουν ερωτήσει. Για άλλη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω που συνεργανώνετε με την Επιτροπή αυτή την εκδήλωση και με χαρά να συμμετάσχω στην περαιτέρω συζήτηση και σα ευχαριστώ πολύ.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 ε, σπάσουμε τα στεγανά και να δούμε διακλαδικά, διατομεακά το θέμα των ωκεανών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχουμε συλλογική ευθύνη να προσφέρουμε λύσεις ε, για ασφαλείς, ε, υγιείς, βιώσιμους στη διαχείρισή τους ωκεανούς. Πώς θα βρούμε καινοτόμους τρόπους να διαχειριστούμε τους ωκεανούς. Εμείς στηρίζουμε τη λεγόμενη διατομιακή προσέγγιση. Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των τομέων. Είναι μια συνεργατική ε, προσέγγιση που τη βλέπουμε και στην έκθεση πρόοδου για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών που εγκρίναμε στις 15 ε, Μαρτίου μετά από δύο χρόνια δράση και μετά το policy paper που είχε κατατεθεί στα τέλη του 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται στην διαχείριση των ωκεανών και στο θαλάσσιο πολυμερέ σύστημα γιατί θέλουμε να εφαρμοστούν σωστά οι φυστάμενοι κανόνες και να πληρωθούν τα διοικητικά κενά. Θέλουμε επίσης διευκόλυνση τη συνεργασία και ανάληψη νέων πρωτοβουλειών. Είμαστε πεπισμένοι πως οι ωκεανοί θα πρέπει να είναι υψηλά στο διεθνές θεματολόγιο στο πλαίσιο και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Ε, όταν είναι ρευστά τα πράγματα, και όταν υπάρχει μια παγκόσμια βεβαιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στο να είναι προβλέψιμος, ε, ε, αξιόπιστος πρωταγωνιστής στο διεθνές προσκήνιο, σε στενή συνεργασία βέβαια και με άλλους φορείς. Στηρίζουμε μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες. Και αυτό το δείχνει και η υποστήριξη που παρέχουμε στο θεματολόγιο του 2030 και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, και υπάρχει και η παγκόσμια στρατηγική εσωτερικό έγγραφο της Ένωσης ε, για την ε, κοινή εξωτερική πολιτική. Εκεί οι ωκεανοί έχουν μεγάλη προτεραιότητα. Τα δύο τελευταία χρόνια προβάλαμε περισσότερο και το θέμα της παγκόσμιας διαχείρισης των ωκεανών στις συνομιλία με τρίτε χώρες, τα περιφερειακά μας προγράμματα και στρατηγικές και αυτό το πράξαμε διότι πιστεύουμε πως η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, για ασφαλείς οδούς, ε, εμπορίας αγαθών, για ένα ασφαλές θαλάσσιο περιβάλλον και για τη διαχείριση των ωκεανών συνολικά υπέρ της υγείας ε, και της σταθερότητας ε, συνολικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Όπως μόλις είπε ο καλός μου φίλος ε, Ζωάου, Αγιάρ Μασάδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά πολλές χώρες να καταπολεμήσουν την παράνομη αλία στα εδάφη για να υπάρχει μεγαλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών συνολικά στις θαλάσσιες περιοχές. Επίσης υπάρχει συνεργασία για την περισυλλογή των μικροπλαστικών και των θαλάσσιων απορριμμάτων σε συνεργασία παραδείγματος χάρη με τις ασιατικές χώρες, την Νοτιοανατολική Ασία, με τις χώρες του ΑΖΕΑΝ. Επίσης έχουμε συνεργασία για την προστασία της Αρκτικής και της Ανταρκτικής όπως προαναφέρθηκε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της έρευνας, της συλλογής δεδομένων. Έχουμε επενδύσει σοβαρά στην επιστημονική συνεργασία και στα προγράμματα δορυφορικής παρακολούθησης μέσω του Κοπέρνικους, για παράδειγμα. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε ενεργοί και ε, να αναλαμβάνουμε εκ των προτέρων δράση για την προστασία των θαλασσών ε, ε, και προστατεύοντας κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, Ατλαντικό, Ασία. Θέλουμε να Προωθήσουμε επίσης ε, το σεβασμό στα νομικά δεσμαυτικά μέτρα και συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Θέλουμε να προωθήσουμε το διάλογο για όλα αυτά τα θέματα. Είναι όλες αυτές πρωτοβουλίες που δείχνουν πώς ανταποκρινόμαστε συνολικά στο θεματολόγιο 2030 και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε και μεταξύ αυτών το στόχο 14 που αφορά τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση ωκεανών, θαλασσών ε, και θαλάσσιων πόρων εν γέννη. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και θα πετύχουμε πρόοδο στον στόχο 14 αν έχουμε πρόοδο και στους άλλου παρότι ο 14ος αυτός στόχος έχει πολλά να προσφέρει για την επίτευξη και των άλλων στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει πρόκληση λοιπόν να λάβουμε κατεπίδουσα δράση για να σώσουμε του ωκεανού. Πρέπει όμω να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία και ε, να αναλάβουμε περισσότερε πρωτοβουλίε για να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί. Έχουμε συλλογικέ ευθύνε. Ε, δεν πρέπει να αποστρέφουμε το βλέμμα από αυτέ. Επίση, η ζωή στου ωκεανού, ε, η ζωή των ωκεανών, δεν είναι απλά αυτό. Είναι η ζωή του ίδιου του ανθρώπου, είναι η ζωή ε, των τοπικών κοινωνιών που ζουν δίπλα στη θάλασσα, που συμβιούν ε, ουσιαστικά με τους ωκεανούς. Ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, την ευημερία συνολικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος και όλα αυτά θα προστατεύσουν τον πλανήτη μας. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας συνεισφορές και προτάσεις γιατί μπορούμε να πετύχουμε μόνο αν συνεργαστούμε ε, όλες οι κοινωνίες και όλοι οι παγκόσμιοι εταίροι και οργανισμοί. Ευχαριστώ πολύ. the... Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κάθε συνάδελφος μπορεί να μιλήσει για τρία λεπτά το ανώτερο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Χωσέ Ινάσιο Φαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Γκαβριέλ Μάτο. Θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχήν τον αγαπημένο μου επίτροπο Καρμένου Βέλα και σας ευχαριστώ για την εργασία σας για την διατήρηση των ωκεανών μας. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω την Γκεζίνε Μάισνερ, τη συνάδελφο και τέλος, για να μην ξεχάσω κανέναν, θα ήθελα να χαιρετήσω τον συνάδελφο Ρικάρδο Σάντας, ε, του ε, τη συνάδελφο Κλάουδια Μοντέρο Γκιάς και τον ε, Ζουάου Μασάδο, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για την αλλιευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η Πορτογαλία έχει μακρά παράδοση στους ωκεανούς και έχει πολλούς ανθρώπους στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Κοινωνία των Πολιτών. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται την ευθύνη της για την χρήση των ωκεανών μέσα στα πλαίσια της ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και δυνάμει του στόχου 14. Μετά το τέλος της διαδικασίας διακυβέρνησης το 2017 ανέκυψε μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να μιλήσω για τρία στοιχεία άξονες για να παραμείνει ο πλανήτης μας γαλάζιος. Ε, διπλωματία για το κλίμα, προστασία του περιβάλλοντος και μπλε πόροι, οικονομική πόροι. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την υπερεκμετάλλευση των πόρων για να μην υπάρχει τέτοια πίεση στα λιευτικά αποθέματα. Θα πρέπει να έχουμε πιο συνειδητή αλία που να μην βασίζεται στο κέρδος και την διφαγία αλλά τη βιωσιμότητα. Έτσι μόνο οι ωκεανοί θα παρέχουν πόρους για τους Ευρωπαίους και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε και την υδατοκαλλιέργεια. Μία άλλη έννοια είναι οι επιπτώσεις του Brexit για να δούμε τι θα γίνει με την απώλεια υδάτων χωρίς να υπάρξει πίεση ως προς τα αλλιευτικά αποθέματα άλλων περιφερειών. Θα ήθελα να σταθώ στην έρευνα και την ενέργεια την καθαρή ενέργεια και την βιοτεχνολογία έτσι ώστε η έρευνα να μετατραπεί σε καινοτομία και να δημιουργηθούν και νέες ευκαιρίες στην πλέ οικονομία. Πιστεύω ότι η, ο, η ενέργεια των ωκεανών θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποτροπή ε, διοξιδίου του άνθρακα και να δημιουργήσει και 500.000 θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να μειωθεί και η χρήση ορυκτών καυσίμων. Όμως ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτή η εκμετάλλευση οδηγεί σε κλιματικές αλλαγές. Οι Ευρωπαίοι τόνισαν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν σε μία οικονομία χαμηλής χρήσης του άνθρακα έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπεράκτιες ε, επιχειρήσεις εξόριξης και να υπάρχει χαμηλή χρήση ή και μηδενική του άνθρακα. Εάν ε, συνεχίσουμε να ρίχνουμε ε, λίματα καθώς και όσο υπάρχουν πετρελαιοκυλίδες ή ρήψη φαρμακευτικών προϊόντων, τότε θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα υγείας. Αυτό αφορά όχι μόνο περιβαλλοντική αλλά και οικονομική ζημία. Έχουμε έναν νέο κανονισμό για τη χρήση εξοπλισμού μοναδικής χρήσης και θα οδηγήσει σε αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά με βάση αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Μόνο το μέλλον θα το ε, δείξει. Αυτό που μετράει τώρα είναι να μαζεύουμε τα λίματα και να τα δεσμεύουμε, τα λίματα που υπάρχουν στους ωκεανούς και να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου, μεθανία και μαύρου άνθρακα. Επίσης, η θαλάσσια δραστηριότητα οδηγεί σε συγκεκριμένες διαρροές, πετρελαιοκυλίδες και ούτω καθεξής. Και αυτό ε, έχει μεγάλη επιρροή και στον ευτροφισμό και στα πλανκτόν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά, αυτά στις αρνητικές απόρριες θα πρέπει να έχουμε αποκλειστικές οικονομικές ε, ζώνες που να είναι 25,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο μέσα στα πλαίσια της ε, φιλόδοξης οικονομικής διακυβέρνησης των ωκεανών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ένας φάρος δράσης στα πλαίσια του Διεθνούς Θαλάσσιου Οργανισμού. Τέλος, ε, για την Αρκτική, οι κλιματικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε ε, αλλαγές μεταξύ Βόρειου Ειρηνικού και Βόρειου Ατλαντικού. Θα πρέπει λοιπόν να αποτρέψουμε την ε, οικολογική καταστροφή με τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα πυρηνικά Έχουμε έναν εξαιρετικό γαλάζιο πλανήτη, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας απασχολούν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δώσω το λόγο στην κυρία Ουλρίκε Ρόντουστ. Την παρακαλώ να πάρει το λόγο για τρία λεπτά. Βέβαια το καταλαβαίνω πως δεν είναι δυνατό, αλλά, ε, αλλά ξέρω ότι θα κάνετε την πρώτη. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι ωκεανοί δεν γνωρίζουν σύνορα. Μας υποχρεώνουν να έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Μας καλούν να μην χτίζουμε τείχους και να απομονώμεθα. Αυτό για μένα είναι ήδη μία αξία αυτή καθ' Τα μέτρα για την ε, πολιτική των θαλασσών έχουν να κάνουν με την αλληλεία, με την εξόριξη βάθους και την χρήση της Αρκτικής. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία μεταξύ διαφόρων ε, δραστηριοτήτων και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ηγετικό ρόλο στη διεθνή πολιτική για τις ε, θάλασσες. Η απάντηση είναι απλή, απλούστατη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω ε, είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια δύναμη η απώλεια θαλάσσιας ε, βιοποικιλότητας και η αποδυνάμωση των οικοσυστημάτων της θάλασσας παίζει μεγάλο ρόλο στην, ε, στο κλίμα. Τις τους τελευταίους μήνες τα λίματα στη θάλασσα έχουν γίνει προτεραιότητα. Επιτέλους, σε μία ε, αποστολή διαπίστωσα ότι ένα ε, ε, ψάρι μπορεί να φάρ καταπιεί πολλά ε, απορρίμματα. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να πνίγουμε τα ψάρια. Και επίσης έχουμε και τις εκπομπές από, το, από τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα βλέπω αυτά στη χώρα μου στην περιοχή μου, μπροστά στην πόρτα μου στο Σλέσφι Χολστάιν. Στα πλαίσια τη παγκόσμια της ε, ε, γενική ανακοίνωση για τη διεθνή πολιτική των θαλασσών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο δεσμεύονται να δράσουν από πλευρά τη Ένωση. Αυτό θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του G7 και των περιφερειακών συμβάσεων για τι ε, θαλάσσιες περιοχέ. Όπω αναφέρθηκε ήδη, αυτή αυτός ο διεθνή συντονισμό έχει κεντρική σημασία. Για το πρόβλημα είναι αναγκαστικά παγκόσμιο. Και αν δούμε και τους στόχους ανάπτυξης του, των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του G20, του G7 και τις διάφορες άλλες ε, περιφερειακές συμφωνίες, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει να υπάρξει μία συνολική προσέγγιση. Αυτή την προσπάθεια πρέπει να την αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερε απαντήσει πρέπει να δώσουμε, για παράδειγμα, για την ε, αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών στη θάλασσα. Από πού όμως να ξεκινήσουμε. Πολλά έχουμε να κάνουμε και είναι πολύ μικρές οι ουσίες, ε, είναι τα μικροπλαστικά και δυστυχώς το 94% των λιμάτων καταλήγουν στη θάλασσα και στο βυθό των θαλασσών. Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί λοιπόν με απλά μέσα. Δεν είναι απλό βεβαίω. Αλλά εμεί εδώ συγκεντρωμένοι πρέπει να έχουμε ένα μόνο στόχο. Να διασφαλίσουμε το μέλλον του γαλάζιου πλανήτη μα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα της θάλασσας. Αλλά όχι μόνο με νέους νόμους. Έχουμε αρκετούς νέους νόμους. Πρέπει να δράσουμε με συνέπεια για να εφαρμόσουμε αυτούς τους νόμους. Να ελέγξουμε την εφαρμογή τους και ενδεχομένως να υπάρχουν και κυρώσεις και μάλιστα σοβαρές κυρώσει. Χρειαζόμαστε τις ε, θάλασσες και τους ωκεανούς για να επιβιώσουμε. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Ουλρίκε. Σεβάστηκες και το χρόνο σου. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, διάφορους εμπειρογνώμονες ε, και ενδιαφερομένους φορείς και θα ακολουθήσει βέβαια και μία ώρα ερωταπαντήσεων στη συνέχεια, ώστε να μπορέσει να ανταλλαγή απόψε μεταξύ ακροατηρίου και πυρογνωμόνων. Σε κάθε πυρογνώμονα θα δώσω 5 λεπτά το πολύ. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Στίβ Τρέντα από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης για 5 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω ενώπιόν σας. Σας ευχαριστώ επίσης ε, που διαθέτετε και χρόνο για να μας ακούσετε. Ε, θα κόψω την ομιλία μου ε, για να μην περάσω το πεντάλεπτο, άρα αφήνω τα εισαγωγικά και πηγαίνω στην ουσία. Η γαλάζια καρδιά του πλανήτη μας αντιμετωπίζει προβλήματα και για να τα αντιμετωπίσουμε πρέπει να βελτιώσουμε την διαχείριση. Βλέπω τρία βασικά θέματα που θα μας επιτρέψουν να το πετύχουμε. Πρώτον, νομίζω θα ήταν ένα ασφάλμα να μην έλεγα ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τι δράσει, του οργανισμού με τι δράσει για το κλίμα. Θα πρέπει να βαθμίσουμε τι προσπάθειε ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην ξεπεράσει την αύξηση των δύο βαθμών ε, καλύτερα το 1,5 βαθμό η θερμοκρασία στο πλανήτη. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση των ε, ανανάσιμων πηγών ενέργεια, σε, σε μείωση των εκτοκαυσίμων για μηδενική ε, σε άνθρακα οικονομία και πρέπει να τα λάβουμε αυτά τα μέτρα παντού και στι θάλασσε και του ωκεανού. Το δεύτερο, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν νέα μέτρα για να προστατευτεί η βιοπικιλότητα στα ανοιχτά, στο βάθο των ωκεανών. Έχουμε κάνει πρόταση, αλλά στα δύο τρίτα ε, των ε, ωκεανών ε, και πάνω από το 90% της εδάτενης μάζας δεν είναι ακόμα προστατευμένο. Πρέπει να προστατεύσουμε τουλάχιστον το 30% των εδάτων των ωκεανών για να μπορέσουμε και εμείς να ωφεληθούμε από τις πολλές περισσότερες που έχει να μας παράσιο και να θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη για να δείξουν ηγετική στάση και να προωθήσουν τις ε, ε, δράσεις και που, που σε επίπεδο ΙΕ ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο για οικολογικά αντιπροσωπευτικό δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων ε, περιοχών. πρόκειται για μια ευκαιρία που δεν θα δοθεί σε πολλές γενιές για τη διατήρηση, για την πραγματική βιώσιμη χρήση και την προστασία των ζωτικών πόρων όρων για αυτή τη γενιά και τις μελλοντικέ γενιές. Επίσης, ε, απευθύνω έκκληση στο να είμαστε διαφανείς ε, για την ε, βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης. Υπάρχουν κάποιοι που αδίστακτα κερδοσκοπούν ε, και πολλές φορές δρούν χωρίς να μπορεί κανείς να τους εντοπίσει. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε σε όλες ε, τις χώρες ε, τις αρχές που θα μπορούν να ελέγχουν για να βλέπουν ποιος, που, πώς κάνει τι. Και θέλουμε να έχουμε απλές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της διαδικασίας διαχείρισης της αλίας. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, την ενιαία δημοσίευση ε, βασικών ε, πληροφοριών για τις άδειε αλίευση ε, των σκαφών. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και δεν είναι και δαπανηρό, είναι δωρεάν. Επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί παγκόσμιο αρχείο μητρό των νεολογημένων σκαφών. Θα πρέπει να πάρουν δράση οι περιφερειακή οι περιφερειακοί ε, ε, και γενικώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να έχουμε ε, καταγραφή όλων των σκαφών. Και αυτό έχει πάρα πολύ μικρό κόστος, αλλά μπορεί να μεταμορφώσει την κατάσταση. Επίσης, σημαντικό είναι και σε ό,τι αφορά την εξόρυξη ε, στα νυχτά και σε όλα τα άλλα επίπεδα να ε, βοηθήσουμε ώστε να μην παρακάμπτουν με τις σημαίες ευκαιρίες ορισμένοι ε, τους κανόνες, να μην απειλείται έτσι η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια, η βιοπικιλότητα. Αυτά απαιτούν την δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε τα μητρώα, τα αναλαμβάνουν ε, την ε, ευθύνη για ε, τα κράτη, μάλλον αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Υπάρχουν δέσμες μέτρων που μπορούμε να εφαρμόσουμε ευθύ αμέσως και μπορούμε να είμαστε πρωταθλητέ και πρωτοπόροι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε που ιδρύθηκε άλλωστε η Ένωση, έδειξε ότι είναι μια δύναμη για το καλό, πολλές φορές χρησιμοποιεί και ε, την, ε, το εμπορικό τη σήμα, αν θέλετε, για να δώσει το καλό παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε δυναμική ηγεσία στο παγκόσμιο προσκήνιο, να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη αλία το κάναμε, χρειαζόμαστε αντίστοιχο όραμα και ε, πρωτοβουλία για εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας των Παρισίων για μια νέα συμφωνία των Εθνών για ε, τα βαθέα ύδατα και να μην υπονομεύονται πλέον οι προσπάθειες που γίνονται από ορισμένους. Ευχαριστώ. Thank you very much, Steve. Now I'm going... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω λόγο στην πρώην ε, Επίτροπο Μαρία Δαμανάκη που είναι επικεφαλής του οργανισμού Nature Conservancy. No. Okay. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γκάμπριελ. Είπα ότι όσο μεγαλώνω, μου είναι πολύ πιο εύκολο να μιλώ όρθια. Κύριε Επίτροπε Βέλα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αγαπητή κυρία Μάισνερ, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το κτίριο και να βλέπω να τα καταφέρνει τόσο καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ζωντανή, αλλά και δυναμική και ε, ζωντανή, ζωηρή όπως η ωκεανοί. Είμαι πολύ ευτυχής και ελπίζω το ίδιο να συνεχίσει και μετά τις επόμενες ευρωεκλογές. Ας το ελπίσουμε τουλάχιστον. Εδώ θα σας μιλήσω για να σας πω ότι εκπροσωπώ μια μεγάλη περιβαλλοντική οργάνωση, μία από τις μεγαλύτερες που έχει έδρα στις ΗΠΑ, τη Nature Conservancy, εκπροσωπούμε, είμαστε μάλλον παρόντες σε 72 χώρες και είμαστε μοναδικοί γι' αυτό. Από τότε που έφυγα από τις Βρυξέλλες έχω μεταβεί παντού. Αυτά που θα σας πω λοιπόν ε, είναι πράγματα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε και είμαι πολύ υπερήφανη γιατί όπου και να πήγα είδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ηγετική ε, δύναμη για την διακυβέρνηση των ωκεανών και την βιωσιμότητα των ωκεανών και ήθελα να πω ιδιαίτερα στους νέους ότι θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα μου υπενθύμησε ότι την τελευταία φορά που ήμουν εδώ ε, ψηφίσαμε την ε, νέα κοινή αλλιευτική πολιτική, η οποία και ισχύει. Άρα τα καταφέρνουμε. Παρακολούθησα τους ε, νέους που μας είπαν «Κάντε κάτι». Μα κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όπως είπε και ο Επίτροπος Βέλα, έχουμε προοδεύσει και προσβλέπουμε στο μέλλον με αισιοδοξία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και καταφέρνουμε πολλά. Χρειαζόμαστε περισσότερα φυσικά. Απειλούνται οι ωκεανοί, βεβαίως, και έχουμε και τις κλιματικές αλλαγές να αντιμετωπίσουμε. Το κλίμα έχει αλλάξει άρδιν, άρα όπως είπε και ο κύριος Λέφερ, δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε σε σχέση με τον βιώσιμο αναπτυξιακό στόχο 14 αν δεν τον συνδέσουμε με άλλους ε, στόχους. Οι κλιματικές αλλαγές ισχύουν και μας ε, κατακλείζουν. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Ζουάου, χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία για να τα καταφέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ένας μείζων οργανισμός, αλλά οι ωκεανοί δεν έχουν σύνορα. Είναι μία έννοια που ξεπερνάει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Νομίζω ότι εάν θέλουμε να κοιτάξουμε προς το μέλλον, θα ήθελα να βασιστώ σε τρεις στόχους. Μπορούμε να συνεργαστούμε επ' αυτών και είμαι σίγουρη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα λάβουν υπόψη αυτή την τάση. Ένας βασικός στόχος είναι 30-30, ε, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε το 30% των ωκεανών μέχρι το 2030 και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για την βιοπικιλότητα αλλά και για την ίδια τη γαλάζια οικονομία, γιατί αν οι ωκεανοί δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η υγεία των ωκεανών έχει μεγάλη σημασία, 30% λοιπόν μέχρι το 2030. Μετά έχουμε την ε, σύμβαση, της συνθήκη ανοιχτών θαλασσών. Συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη και συνεργάζομαι και εγώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ηγετική δύναμη υπέρ της Σύμβασης Ανοιχτών Θαλασσών με βάση την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης και της βιωσιμότητας και φυσικά αποτιμώντας το τι συμβαίνει. Βεβαίως χρειαζόμαστε και χρηματοδότηση, το είπαν και οι νέοι μας. Τα χρήματα είναι κάτι το σημαντικό, το ξέρετε, αλλά για να προστατεύσουμε τους ωκεανούς υπάρχει και ένα εμπλεκόμενο κόστος. Δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει πια δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό θα πρέπει να μοχλεύσουμε τα χρήματα που διατίθενται για τους ωκεανούς. Ε, υπάρχει με ένα ιδιαίτερο ομόλογο το επωνομαζόμενο ε, γαλάζιο γαλάζιο ομόλογο στις Σεϊχέλες. Τώρα θα μεταβώ στο Μεξικό και θα δείξω τι γίνεται στο Κανκούν, τι γίνεται στις ε, κοραλιογενείς περιοχές και φυσικά υπάρχουν και πριμοδοτήσεις εκεί όπου χρειάζεται. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε καινοτομίες και χαίρομαι για τη Γενική Διεύθυνση ε, ΜΑΡΕ προβάλλει την καινοτομία. Πολλά αλλάζουν και χαίρομαι γι' αυτό. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον Επίτροπο Μοέδας που μίλησε για την Σίλβια Έρλ, η οποία κατοικεί στις ΗΠΑ και η οποία είπε ότι οι άνθρωποι είναι όντα, σκεπτόμενα όντα. Ο Πλάτωνας είχε πει προερχόμαστε από τη θάλασσα και θα επιστρέψουμε στη θάλασσα. Το ξέρουμε αυτό. Αποτελεί μία πραγματικότητα. Είμαστε θαλάσσια όντα λοιπόν, ας είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και ας κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστούμε και εμείς Μαρία. Mr. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μάτινσεν από, τη από την ΦΑΟ και το Διοικητικό του Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μάισνερ, Επίτροποι, Προηγούμε παρελθόντες και παρόντες, για να ε, παραφράσω και τα λόγια του κυρίου Φαρία. Κυρίες και κύριοι, Τέσσερα είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Εάν θέλουμε βιώσιμη διατροφή και ε, επιστημιστική ασφάλεια για όλους. Τα τέσσερα βασικά ζητήματα καταρχάς επηρεάζονται και από τέσσερις μείζονος σημασίας παράγοντες. Πρώτα απ' όλα η αύξηση του πληθυσμού και όπως όλοι ξέρουμε θα φτάσουμε τα 10 δις το 2050 το δεύτερο είναι η κλιματική αλλαγή. Όλοι καταλαβαίνουμε την ε, σημασία και τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει στους ωκεανούς και τις κοινότητές μας. Το τρίτο είναι η βιοπικιλότητα που σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με το μέλλον και με τις λύσεις. Και το τέταρτο είναι η ρήπανση. Το πλέον προφανές ε, φαινόμενο είναι αυτό των πλαστικών και μετά βεβαίως έχουμε να κάνουμε και με τα απόβλητα που προέρχονται από την ξηρά. Το 10% μόνο έχει να κάνει με την δραστηριότητα των ίδιων των ωκεανών και τους ωκεανούς και με τα απορρίμματα των ε, αλληλευτικών εργαλείων ή της αλίας. Και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτά τα τέσσερα βασικά ζητήματα όλα έχουν να τέσσερις υποδιαιρέσεις κοινωνικο-οικονομικές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως σκέφτομαι τα δικαιώματα των πληθυσμών, των κοινοτήτων, τα θέματα του φύλου, της ισότητας των φύλων. Οι μισοί άνθρωποι στον κόσμο στην τον τομέα της επεξεργασίας των προϊόντων της αλίας είναι γυναίκες και η νεολαία. Η απασχόληση της νεολαίας, που είναι ένα άκρο σημαντικό ζήτημα. Κάτι λίγο πιο καθημερινό, το θέμα των ποιοτικών στατιστικών. Διότι σε αυτές βασίζουμε όλες τις αποφάσεις μας. Και το τρίτο είναι πιο ανησυχητικό είναι η επισητιστική ασφάλεια. Βλέπουμε νέα στοιχεία να αναδύονται με διαφορετικό ένδυμα κάθε φορά. Ας πούμε η αντίσταση στα αντιβιωτικά που έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις αλλά αφορά και την αλία και τους ωκεανούς προφανώς. Και θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω το τέταρτο στοιχείο που συμπεριλαμβάνει τα τρία προηγούμενα το τεράστιο χάσμα ανάπτυξης τη διαφορά που ακόμα παραμένει μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών. Τα τέσσερα αυτά μείζονο σημασία ζητήματα έχουν να κάνουν με τις θάλασσες και κυρίως την παράνομη, άναρχη και μη ρυθμισμένη αλία. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο τμήμα του μεγαλύτερου παζλ και είναι μία ανοιχτή πληγή. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και τα υπόλοιπα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προσπάθειές μας. Έχουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο που ανέφερε πριν ο Στίβ. Έχουμε τις διάφορες υποσυμφωνίες που ανέφερε προηγουμένως και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προηγουμένως και όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν ε, υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά τη. Αλλά και από χώρες όπως η Σουηδία ξεχωριστά. Ε, ένα μέρος της λύσης είναι οι οργανισμοί προγραμματισμού της αλίας. Εάν χρηματοδοτηθούν σωστά, μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως μόνο ένα μικρό τμήμα τους χρηματοδοτείται σωστά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Το δεύτερο θέμα είναι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που το καθορίζουν ως αρμοδιότητα και προνόμιο τα εθνικά κυρίαρχα κράτη-μέλη. Τα τελευταία 25 χρόνια επιτύχαμε πρόοδο, ιδίω στο ε, νότιο ημισφαίριο και σε ένα μέρος του βορείου, όμως στο νότιο ημισφαίριο τα πράγματα αντιστράφηκαν. Η πρόοδος οπισθοδρόμησε η αλληλευτική ένταση και δραστηριότητα προχώρησε από τα βόρεια στα νότια. Η κατάσταση των αποθεμάτων δεν βελτιώνεται. Δεν ε, τα πάει και άσχημα, αλλά δεν μπορούμε να επιζήσουμε με το 1 τρίτο των ε, αποθεμάτων να αλλιεύεται. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Εδώ γίνονται δύο ζητήματα. Οι απομακρυσμένες θάλασσες και οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Απλώς πρέπει τώρα να το εφαρμόσουμε και χρειαζόμαστε και τους απαραίτητους πόρους. Το τρίτο ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Οι παράκτιες κοινότητες, οι γαλάζιες όπως έχουν ονομαστεί, οι μικρή κλίμακας αλία, οι κοινότητες που βασίζονται στην αλία ε, κοινότητες μεταναστών, 25% ε, των ανθρώπων που ζουν από την αλλιευτική βιομηχανία βασίζονται σε αυτέ τι δραστηριότητε. και τα μισά από θέματα τα αλλιεύει ο αναπτυσσόμενο κόσμο. και τα καταναλώνει ο ανεπτυγμένο. ενώ το άλλο μισό το αλλιεύει ο ανεπτυγμένο κόσμο και έχουμε 95% του πληθυσμού. Είναι περίπλοκο αυτό το ζήτημα και αυτή η ισορροπία εδώ. Χρειαζόμαστε νέε λύσει και εργαζόμαστε σκληρά για να το πετύχουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε υποστήριξη υποστήριξη από οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τέταρτο ζήτημα έχει να κάνει με την αυξημένη ε, προσφορά ε, των προϊόντων στο μέλλον, κυρίως από την πηγή της υδατοκαλλιέργειας. Χρειαζόμαστε πιο πολλά ψάρια για τον πληθυσμό που αυξάνεται. Δεν θα τα ε, πάρουμε από την αλεία στις θάλασσες και τους ωκεανούς, θα προέλθουν από την υδατοκαλλιέργεια. Ε, εδώ και την υδατοκαλλιέργεια. Εδώ υπάρχει θέμα οικολογικό αποτυπώματος των παραγωγικών συστημάτων της υδατοκαλλιέργειας. Εάν όμως το βάλουμε στόχο, μπορούμε να σχεδιάσουμε τέτοια παραγωγικά συστήματα που δεν θα βαραίνουν τόσο πολύ το περιβάλλον. Το αποτύπωμά τους θα είναι ε, καλύτερο από ό,τι σήμερα. Και θα έχουμε βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων και στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο κ. Πασκουάλ Γοναντεφέο, Διευθύνων Σύμβουλος της Κονοτέκο ΕΣΠΕ. Για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πω ότι είναι ε, για μένα πραγματικό προνόμιο να βρίσκουμε εδώ. Είμαι πρόεδρος ενός τερμινάλ του Μιλάνου του λιμένα της Νάπλης που ανήκει σε μια πολυεθνική εταιρεία που εξυπηρετεί το εμπόριο και συνδέει χώρες από όλο τον κόσμο. Επίσης είμαι πρόεδρος ε, της περιοχής της ε, Καμπανίας. Εκεί συγκεντρώνονται όλες οι επιχειρήσεις ε, της επιμελητίας και συνδέουν τους λιμένες με τις οδικές μεταφορές και σε μία από τις πιο σημαντικές ενώσεις της Ιταλίας που εδώ και πολύ καιρό ασχολείται για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Σήμερα υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη σχετικότητα ε, για την θαλάσσια οικονομία, το, η έννοια της γαλάζιας οικονομίας ε, που αρχίζει να αναδύεται σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ε, χάρη στην μεταποίηση των ουσιών που γίνονται εμπορεύματα. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με άλλους παγκόσμιους οργανισμούς εργάζονται για να ρυθμίσουν μία σειρά δράσεων που να καθιστούν το κλάδο μας πιο βιώσιμο. Έτσι λοιπόν ε, είναι γνωστή η στόχη. Το 2020 προβλέπεται μείωση του ποσοστού ε, του θείου ε, από το 3,5% στο 0,5%. Όμως δυστυχώς πρέπει να αναφέρω ότι στο παρελθόν οι πολιτικές των κυβερνήσεων ε, συχνά δεν επένδυσαν σε υποδομές που να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μεταφορών μέσω της θάλασσας, που ρηπαίνει περισσότερο, υποστηρίζοντα αντίθετα τρόπους μεταφοράς ε, χερσαίου ε, με κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος για τις μελλοντικέ γενιές σήμερα. Η συνειδητοποίηση της σημασίας μιας ε, φόρου ανάπτυξη των λιμένων και για των θελέσεων μεταφορών ε, αναδύεται λένε και περισσότερο. Ε, αποτελούν παράδειγμα των πολιτικών ε, των ναυτιλιακών εταιριών που στοχεύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε αυτές οι πολιτικές έχουν να κάνουν με τη χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και στη δραστική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται στα λιμάνια. Ε, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα της εταιρεία του ομίλου όπου συμμετέχω. Έχουμε μια ε, εταιρεία που ανήκει στην MSC. Έχουμε εγκαταστήσει ε, μηχανές για να υπάρξει αναγέννηση βιώσιμη και οικονομική ε, των αποβλήτων που παράγονται επί του σκάφους και είναι δυνατόν να μειώσουμε ε, τον όγκο μέχρι τον 90%. Και αυτά χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα ε, και πάρα πολλά τερματικά στους λιμένες έχουν στρέψει τις πολιτικές τους προς την απόκτηση μέσων να τροφοδοτούνται δηλαδή τα πλοία με ηλεκτρισμό, ηλεκτρικό ρεύμα και αντικαθιστούν τα παραδοσιακά καύσιμα. Επίσης εφαρμόζουν τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον έλεγχο των μηχανών. Σε αυτή την επτική, οι εθνικές και κοινοτικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν με τις governance των λιμένων, προκειμένου να παρέχονται περισσότερες κατάλληλες υπηρεσίες και ενεργειακά αποδοτικές που ε, να ε, βοηθούν τις, ε, ευκαι... τις οι πολιτικές των ε, θεσμικών οργάνων θα έπρεπε λοιπόν να ακολουθούν δύο άξονες, την υλοποίηση δημοσίων υποδομών, ε, δηλαδή ε, εξοπλισμό για ε, ηλεκτρικό ρεύμα και ε, να υπάρχουν ε, αποθήκευση φυσικού αερίου, πολυτροπικές διασυνδέσεις με την επικράτεια, παραδείγματο χάρη στην Ιταλία και με κάποια καθυστέρηση έχουν ξεκινήσει διαγωνισμοί για να δημιουργηθούν αυτές οι αποθήκες για το ευρωπημένο φυσικό αέριο. Και από την άλλη θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι οικονομικοί φορείς που ε, ασχολούνται μόνο με την ναυσιπλοεία, με τις θαλάσσιες μεταφορές, ε, να κάνουν αξιοσημείωτες επενδύσεις. Δηλαδή, ε, να δοθούν και κίνητρα σε αυτούς τους επιχειρηματικούς φορείς να επενδύσουν σε τεχνολογικές λύσεις που να εμπνέονται από τη γαλάζια οικονομία. Λέγεται ότι η γαλάζια οικονομία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επομένως, η αναγκαιότητα υπάρχει για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά όλοι μαζί. Όμως ε, υπάρχει και υποχρέωση, λαμβάνοντας ε, υπόψη την ιστορική στιγμή που θα βιώσει η χώρα μου αυτή την εβδομάδα, να προσέξουμε τι ε, προσφέρεται από την Κίνα. Η λεγόμενη πρωτοβουλία Bent Elrod. Η Κίνα, και θέλω να το επενθυμίσω, την προηγούμενη δεκαετία παρουσιάστηκε σε όλο τον κόσμο το παγκόσμιο εργοστάσιο με χαμηλό κόστος εργασίας ε, και ε, ποιότητα παραγωγής. Έτσι λοιπόν μπόρεσε να αγοράσει τις τεχνολογίες δυτικών εταιριών και αφού κατέκτησε την τεχνολογία, προέβη σε αναβάθμιση στην αλυσίδα αξίας και στην ποιότητα των προϊόντων και παρουσίασε στον κόσμο νέες τεχνολογίες πιο πολύπλοκες από τις δυτικές. Το 2014 ξεκίνησε ένα τεράστιο φαρανικό σχέδιο ε, χρησιμοποιώντας 120 ε, δισεκατομμύρια ε, στις παγκόσμιες αγορές και αυτή τη στιγμή μόνο 70 χώρες, αλλά σκοπεύει να συνάψει 100, συμφωνίες με 120 χώρες για να δημιουργήσει το Silk Road, αλλά και το One Belt, One Road, για να, συνδεθεί, συνδεθούν με την αγορά της. Ε, βλέπουμε ότι η παρουσία στο ιστορικό της Ένωσης των κρατών που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Κίνα, πέρα από το ότι θα υπάρξουν μειονεκτήματα και απώλεια της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές μπορεί και να αποδυναμώσει πολύ τη δράση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας. Και δεν είναι τυχαία και η προσοχή που δίνεται στην Ελλάδα ε, δυστυχώς έχει παραχωρήσει ένα στρατηγικό λιμένα στην Κίνα, τον Πειραιά και δυστυχώς ε, υπάρχει και επιρροή και στις πολιτικές αποφάσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιες ε, χώρες ε, που στην αρχή, κάποιες χώρες που έδειξαν θυσισμό, όπω το Πακιστάν, Σιέρα Λεόνε, το Μπαγκλαντές ε, και άλλε, στη συνέχεια κύρωσαν τι δεσμεύσει του, επειδή αυτά, αυτά τα προγράμματα, τα σχέδια των υποδομών θα χρεώναν υπερβολικά τις χώρες. Σήμερα μιλάμε στην Ιταλία και για την ανάλυση κόστου-οφέλου. Αφού έκαναν τέτοιες αναλύσεις, γύρισαν την πλάτη στην οδό του μεταξιού. Εγώ, όντα Ευρωπαϊστή, εύχομαι η Ευρώπη να παραμένει πάντοτε πιο ενωμένη για να έχει την ικανότητα και την πολιτική βούληση να υλοποιήσει όλε τι απαραίτητε δράσει και να δώσει του αποφασιστικού αγώνε για να κερδίσει την, αυτήν τη γαλάζια οικονομία. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους ε, ομιλητές. Αρχίζει αμέσω η συζήτηση, ερωτήσει και απαντήσει Άμε χάλια από χρόνο που δείχνει ότι δεν είμαι καλός πρόεδρος γιατί δεν σας διέκοψα. Ας προσπαθήσουμε στο γύρο των ερωταπαντήσεων να κερδίσουμε χρόνο. Παρακαλώ ποιος θέλει το λόγο να σηκώνει το χέρι του και να περιμένει να του δίνεται ο λόγος. Σας παρακαλώ να κάνετε ερωτήσεις πάρα πολύ σύντομες και όχι μεγάλες τοποθετήσεις ε, για το τι πρέπει να γίνει. Συγκεκριμένες ερωτήσεις να συστήθετε πρώτα και να μας πείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας κάθε φορά. Ο Τζουζέπε Σκινότη από την Nova Meet, παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλωσορίζω και όλους τους προσκεκλημένους και όσους ήρθαν, κυρίως τους νέους. Πολύ γρήγορα, είμαι ο κύριος Σόντι, πρώην μηχανικός και εργάζομαι για το Nova Meet. Και ασχοληθήκαμε με τις εναλλακτικέ προϊόντων ψαριών και κρέατος που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο εμπορευματοποίησης. Μας ενδιαφέρει στην Ευρώπη να δούμε πώς ε, έχει αυξηθεί στη διατροφή μας κατανάλωση προϊόντων κρέατος και ψαριού. Τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Οργανικού Υγείας δείχνουν ότι είναι, δείχνουν ότι είναι ανησυχητικά ε, όσα συμβαίνουν για όλους μας και ότι είμαστε στην, κα, κακό δρόμο για να προστατεύσουμε τους ωκεανούς. Υπεραλίευση, απώλεια της βιοπικιλότητας, ε, ρήπανση από τα μικροπλαστικά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ωκεανοί υπάρχουν εδώ και δύο εκατομμύρια χρόνια, ενώ η ανθρωπότητα ενώ και δύο εκατομμύρια μόλι χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν το 2019 πρέπει κάτι να αρχίσει να κάνει για αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Έχουμε και δυνατότητε και ευθύνε. Είναι και τύχη που θα μπορούσαμε ε, να μείνουμε στην ιστορία ω η πρώτη γενιά ανθρώπων που αντέστρεψαν την τάση των αλλαγών του κλίματο για τα παιδιά μα και το μέλλον και Προτού ε, γίνουμε 10 δι άνθρωποι στον πλανήτη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει νέε ευρωπαϊκέ τεχνολογικέ λύσεις για να χειριστεί καλύτερα του πόρου των ωκεανών μα. Στην Ευρώπη έχουμε ταλέντο, δημιουργικότητα και τη δύναμη για να φέρουμε αυτέ τι λύσει στην αγορά και να σώσουμε του ωκεανού μα. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερο, η καλύτερη κινητήρια δύναμη για να σώσει τους ωκεανούς μας. Ε, παρά τη μεγάλη κρίση τη ανθρωπότητα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Let's do it. Να ξεκινήσουμε από σήμερα κιόλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ομαδοποιήσουμε λίγο τις ερωτήσεις ανά για να δοθούν απαντήσει. Το έδρανο 115. Επειδή δεν ξέρω τα ονόματά σα, θα λέω το αριθμό του εδράνου στο οποίο κάθεστε. Εξαιρετική η διάσκεψη. Υπάρχει ένα ταμπού. Το οξυγόνο δεν το συζητάμε το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, συζητάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι ζωή το οξυγόνο. Η θάλασσα μας δίνει το οξυγόνο. Μήπως θα πρέπει να αρχίσει μια πολύ μεγάλη έρευνα για το οξυγόνο και μάλιστα την παραγωγή οξυγόνου από τους ωκεανούς. Ευχαριστώ. 248. Pierre Dumoulin, je représente... Pierre Dumoulin, εκπροσωπώ μια ε, τοπική ε, ε, επιτροπή στις Βρυξέλλες γιατί δεν μιλάμε για όλα τα πυρομαχικά. 35.000 ε, ετών στα ανοιχτά του ΚΝΟΚ ε, ανάμεσα στην ε, Σκοτία και την Ιρλανδία και στη Βαλτική. Έχουμε δανούς ψαράδες, τραυματίες και πάρα πολλά επεισόδια. Οι δανοί ψαράδες υφίσταται πολλές μεγάλες δηλητηριάσεις και έχουν πρώτες βοήθειες κατά των δηλητηριάσεων ε, τύπου υπερίτη ε, στα σκάφη του, στα λεφτικά. Η Φιλανδία ήδη δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οβίδες έχει βγάλει ε, από εκεί που περνάει το, ο αγωγός Nord Stream 2 στα χωρικά της Ήδατα και αλλού. Είναι πολλά τα τοξικά πυρομαχικά στην Αδριατική, στην Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή οι Άπωνες είναι οι μόνοι ε, που ανακτούν ε, αυτά τα πυρομαχικά για να τα καταστρέψουν ε, από τα βάθη των ωκεανών. Δεν θα μιλήσω για τις λίμνες της Ελβετίας ή για την Αμερική. Αυτά θα τα αναλάβει ο κύριος Τραμπ. Θα πρέπει η Ευρώπη επιγόντως να βιαστεί, αν δεν θέλουμε να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, να βιαστεί τι εννοώ. Στο Οικαιογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας έχει γίνει μια έρευνα που λέει αν, βγει το 1 έκτο, το αν δεν βγει το 16% ε, θα πεθάνει για 30 χρόνια η Βαλτική, αν αδρανίσουμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιληφθεί. Ε, με ρομπότ θα μπορούσε να γίνει αυτό, οι Κινέζοι ενδεχομένως, μια Αμερικανική εταιρεία, ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Θα απαντήσουμε στι τρει αυτέ ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ ερωτήσεις να κάνετε, όχι τοποθέτηση και εξήγηση 1,5 λεπτό, γιατί δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Ποιο θέλει να απαντήσει. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Γκαμπριέλ. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Ήδη εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον ορίζοντα 2020, ε, λέει ο Ζωάγκυρα Ματσάδο, για την έρευνα στους ωκεανούς. Και αυτά που σας είπα, ε, το ακούσαμε και στην εισαγωγή από τον Επίτροπο, τον κύριο Μοέδας. Στο νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπης, όπου αυξάνεται, ε, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο προπολογισμό, έχουμε αυτό τον ειδικό στόχο ε, για τους ε, ωκεανούς. Να έχουμε αυτή την έρευνα χάρη στην πολιτική ηγεσία των Επιτρόπων Βέλα και Μοάδας, σε αγαστή συνεργασία. Και ο συνάδελφος Ζάιρικ Πακέ είναι στο επόμενο πάνελ και θα μπορέσει σίγουρα να σας πει περισσότερα. Αυτή είναι όμως η πρώτη φορά όπου θα έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα αναγνωρισμένο παγκοσμίω ως από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα και θα έχουμε ειδικέ αποστολές αυτή τη φορά για τους ωκεάνου Ευχαριστώ. Άλλος. Um, je voudrais parler à monsieur... Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο που μίλησε προηγουμένως και να πω για τις τοξικές ουσίες και για τα πυρομαχικά κατάλοιπα. Υπάρχουν χειρότερα προβλήματα στους ωκεανούς. Υπάρχουν τα πυρηνικά απόβλητα, λόγω χάρη. Ξέρετε ότι στη δική μου τη χώρα, την Πορτογαλία, αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε ε, ολόκληρες ε, δεξαμενές με τοξικά απόβλητα από πυρηνικά εργοστάσια. Και αυτά καλά θα, καλό θα να τα συζητήσουμε. Το έχω ξαναπεί στο Κοινοβούλιο. Το έχω πει. Δεν είναι μόνο ε, τα τοξικά πυρομαχικά απόβλητα που ή μπορεί να είναι ανώδυνα. Ε, εδώ και στις ευρωπαϊκές ακτές έχουμε τέτοια προβλήματα όπως τα μπιτόνια που σας είπα που ανακαλύπτουμε. Και καλό θα ήταν να το δούμε εν ώψη και της ερχόμενης εβδομάδας. Άλλα σχόλια, κυρία Δαμανάκη. like just to say Θα ήθελα απλώς να πω ότι έχει δίκιο ο κύριος εκεί. Δεν έχουμε αρκετά επιστημονικά στοιχεία, ούτε αξιολογήσεις που μπορεί να συνδέουν ε, την κλιματική αλλαγή με τα μεγάλα βάθη των ωκεανών. Έχουμε μελετήσει τις παράκτης περιοχές, ε, τα ε, κοραλιογενή νησιά και άλλους βάλτους δημοθάλασσες κοντά στη θάλασσα, αλλά για τα μεγάλα βάθη των ωκεανών δεν έχουμε μελετήσει την κλιματική αλλαγή. Αν υπάρξουν επιστημονικά στοιχεία, σίγουρα θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις προσπάθειες. Και τα πανεπιστήμια μπορούν να βοηθήσουν και τα Ινστιτούτα και συμφωνώ με τον ΖΟΑΟ. Ο κύριος Μάτο. Α, η κυρία και Ρόντος. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τα τοξικά ε, πυρομαχικά και τις τοξικές ουσίες. Ε, εγώ είμαι από το Σλέσφικ Χολστάιν ε, ε, που βρέχεται από τη Βαλτική. Και στη δική μου περιφερειακή πολιτική, στην Περιφερειακή Βουλή, συζητούμε και με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κρατηδίου από τότε που ασχολούμαι με την πολιτική και βλέπετε από τα γκρίζα μου μαλλιά ότι είναι πολλά τα χρόνια. Έχω μάθει λοιπόν πάντα ότι το Ταμείο είναι μείον Ό,τι και να θέλεις, ό,τι, όσο και μεγάλο να είναι το πρόβλημα, ε, ο ένας ε, το παραπέμπει στον άλλον και ε, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε χρήματα. Γι' αυτό χαίρομαι κάθε φορά που ακούω διαμαρτυρίες και δυνατές φωνές που διατρανώνουν θα πρέπει να πιάνουν περισσότερο τόπο τα χρήματά μας. Συμφωνώ απολύτως. Επιγόντως θα πρέπει να δράσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε νόμους λογικούς για την αλεία. Ε, ε, ότι και δεν μπορούν μετά να ψαρεύουν οι επειδή είναι καταδηλητηριασμένα τα ψάρια. Ε, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για ερωταπαντήσεις γιατί μιλήσαμε εμείς πολύ. Θα πρέπει να δώσουμε τώρα το λόγο στο δεύτερο πάνελ για τις ε, καθαρές θάλασσες και ο Σας Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ από το πρώτο πάνελ. May I invite the speakers for panel two on the stage. Να καλέσω τους ομιλητές να έρθουν ε, στο πάνελ, παρακαλώ. Hello everyone. Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να σα καλέσω να καθίσετε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο πάνελ. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και θα έρθει και ο πρόεδρο Ταγιάννη, ο οποίο θα μα απευθυνθεί. Στι 5 παρατέταρτο προβλέπετε. Εν τω μεταξύ, να σα συστηθώ. Λέγομαι Αντίνα Βαλεάν. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου να προεδρεύω στο πάνελ αυτό με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τους συναδέλφους, ε, μέλη του Κοινοβουλίου και εμπειρογνώμονες. Ο τίτλος ε, του πάνελ είναι «Η επίτευξη υγιών καθαρών θαλασσών και ωκεανών». Θα ακούσουμε τις εισαγωγικές παρατηρήσεις μου και κατόπιν ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Κοινοτομία θα μας απευθυνθεί, ο Ζανερικ Πακέ, κατόπιν θα ακούσουμε την Γιώνα Ντρέικ, ε, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα τελευταία έτη στο να διατηρήσουν την ηγετική θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και κατόπιν θα ολοκληρώσουμε με ομιλητέ από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Δυστυχώ δεν θα έχουμε πολύ χρόνο για διάλογο. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας δύο λόγια. Δυναμή του δικού μου ρόλου. Ξέρουμε ότι οι ωκεανοί αποτελούν το 7% της επιφάνειας του πλανήτη και ε, το 97% του είδους καλύπτει πάνω από το 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, θάλασσα μας δίνει κινητικότητα, ψυχαγωγία, φάρμακα, αλλά επίσης οι ωκεανοί ρυθμίζουν το κλίμα, μας δίνουν οξυγόνο και ε, απορροφούν μεγάλο ποσοστό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Με άλλα λόγια, οι υπηρεσίες που προφέρονται από τους ωκεανούς είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Οι, ανθρω... οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στο οικοσυστήμα των ωκεανών λόγω της κλιματικής αλλαγής, της οξύνησης, της υπερελίευσης, της ρήπανση ε, ε, ε, και των σκουπιδιών, της καταστροφής, των οικοτόπων και των χωροκακτητικών ειδών. Όλα αυτά έχουν καλυφθεί από νομοθεσία και από έγγραφα με κατευθυντήριες γραμμές. Εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε αναλάβει δράση προκειμένου να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας των νομοθετημάτων. Οι συνάδελφοι στη συνέχεια θα σας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία που έχει συμπεριλάβει το Κοινοβούλιο στην νομοθεσία προκειμένου να βελτιώσει το καθεστώς των ωκεανών. Όμως η θέση σε ισχύ της νομοθεσίας αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Σε ό,τι αφορά τις γενικές πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική πριν 11 χρόνια έθεσε τον στόχο κλειδί να διασφαλίσει ένα καλό περιβαλλοντικό καθεστώς ε, όλων των ε, θαλάσσιων υδάτων μέχρι το 2020. Σε επίπεδο ε, Ηνωμένων Εθνών, ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 14, δηλαδή να χρησιμοποιούνται οι ωκεανοί και θάλασσες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει τεθεί στο θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς ε, έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μα Πέρσι, η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για την εξολόγηση προγραμμάτων των κρατών μελών για τα μέτρα που είχαν πάρει δυνάμει τη οδηγία πλαίσιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχαν καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε τα κράτη-μέλη για να αναπτύξουν ε, τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, η εξολόγηση δείχνει ότι όλες ε, οι πιέσει στο περιβάλλον στο θέλασσο περιβάλλον δεν καλύπτονται κατάλληλα από τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Τα ίδια τα προγράμματα έχουν ε, ψηλά ποσοστά φιλοδεξίας ε, να πετύχουμε ένα καλό περιβαλλοντικό καθεστώς μέχρι το 2020. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι το 2017 πολλές πολιτικές ε, ε, είχαν τεθεί σε εφαρμογή και παρά αυτό το γεγονός, παρά δηλαδή το ότι υπήρξαν θετικά αποτελέσματα, οι πιέσεις ε, στο θαλάσσια περιβάλλοντα συνεχίσουν να αυξάνονται. Πράγματι, η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2015 ε, της ε, περιβαλλοντικής στρατηγικής μας έδειξε ότι έχουν γίνει πολλές ε, προσπάθειες αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σε κάποιους τομείς δείχνει ότι συνεισφέρει στο στόχο 14 το SDG, δηλαδή έχει δεσπίσει προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές. Ε, σε ό,τι αφορά ε, τα ε, θαλάσσια απόβλητα. Είχαμε το 1998 την πρώτη σχετική νομοθεσία. Από τότε η ρήπανση με πλαστικά των ωκεανών έχει διαβλάβει τέτοιο μέγεθος και θεωρείται ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε περισσότερο πλαστικό από ψάρια στους ωκεανούς. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια ευρεία σειρά εργαλείων όπως ε, χάρη ε, κανονισμούς ε, για την συλλογή των αποβλήτων και τον οδηγία για τις εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων στους λιμένες. Και αφού έχουμε συνεισφέρει στην υιοθέτηση του πακέτου για τα απόβλητα το 2018 που θα αυξήσει τους στόχους ανακύκλωσης, και πρόσφατα, ε, τον προηγούμενο Δεκέμβριο, θετήσαμε για την οδηγία για τα πλαστικά μία χρήση. Εκεί θέτουμε πιο αυστηρούς κανόνες για τα πλαστικά προϊόντα και τη συσκευασία μεταξύ που είναι μεταξύ των 10 ε, πρώτων προϊόντων που βρίσκουμε στις παραλίες. Η οδηγία θα απαγορεύσει ε, τη χρήση κάποιων πλαστικών μιας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικέ και συγκεκριμένα μέτρα θα εισαχθούν για να μειωθεί η χρήση των λοιπόν πλαστικών προϊόντων ε, που απορρίπτονται και για τα οποία δεν υπάρχουν εναλλακτικέ. Είναι λοιπόν σαφέ ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και φροντιδικαιανή και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με ισχυρή διεθνή συνεργασία. Υποστηρίζουμε πλήρω την ανάπτυξη νομικών δεσμευτικών μέσων όπως η βιώσιμη χρήση και η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνική δικαιοδοσία δυνάμει τη Η μείωση τη ανθρώπινη πίεσης στου ωκεανού είναι μια δέσμευση που θα πρέπει να αναλυφθεί σε όλα τα επίπεδα από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι τον μεμονωμένο καταναλωτή. Και με αυτέ τι εισαγωγικέ παρατηρήσει, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζάνερικ Πακέ, τον Γενικό Διευθυντή τη διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έρευνα και η καινοτομία. Παρακαλώ. Κύριε Πακέ, έχετε πέντε λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτό το πάνελ. Και εφόσον μίλησε ήδη ο Επίτροπος, λίγα λόγια για το πού βρισκόμαστε στην έρευνα σχετικά με τους ωκεανούς. Κοιτάζουμε το μέλλον και την προετοιμασία του επόμενου προγράμματος πλαισίου για τον ορίζοντα της Ευρώπης. Αυτό υπόθηκε και στην προηγούμενη σύνοδο και θα το ακούτε και από όλα τα μέλη του πάνελ. Οι ωκεανοί μεταβάλλονται ε, ε, εκ βάθρων από όλε τις απόψεις κυρίως από την άποψη τη μετεωρολογική. Ε, οι νέε κανονικέ συνθήκε είναι το απρόσμενο των αλλαγών του καιρού. Οι καταιγίδε ε, διαρκώ είναι διαφορετικέ. Είδατε ότι ο τυφώνα στη Μοσαμπίκη είναι ένα περιστατικό που δεν θα είχε λάβει χώρα ούτω υπό άλλε συνθήκε. Και βεβαίω ο καιρό επηρεάζει και το τι γίνεται στου ωκεανού. Το θέμα του οξυγόνου στους ωκεανούς. Οι ωκεανοί ε, παράγουν τον αέρα που αναπνέουμε. Και αυτό όμως αλλάζει. Οι ωκεανοί παράγουν τα τρόφιμα που καταναλώνουμε αλλά και εκεί επισυμβαίνουν αλλαγέ, Οι ωκεανοί είναι η μεγαλύτερη αποθήκη, η δεξαμενή άνθρακα που διαθέτουμε. Επίσης, η σχέση των ωκεανών σε σχέση με το λιώσιμο των πάγων ε, μεταβάλλεται, ε, αλλάζει η στάθμη της θάλασσας και ο ρυθμός ανώδου της και εκεί θα συνεχιστούν οι αλλαγές. αλλά τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ήδη το 2016 το μέσο επίπεδο της θάλασσας ήταν 20 εκατοστά παραπάνω από ό,τι πριν από έναν αιώνα. Και με τις τωρινές τάσεις υπολογίζουμε 60 εκατοστά συνολικά παραπάνω μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτή τη στιγμή η ωκεανή είναι η ισχυρότερη πηγή βιοπικιλότητας. Αυτό είναι γνωστό για τον πλανήτη μας και το γονιδιωμά του, αλλά αυτό μεταβάλλεται γοργά. Οι ωκεανοί όμως είναι και το νέο σύνορο που αν ξεπεράσουμε θα μετρήσουμε κατά πόσο είμαστε καινοτόμοι. Υπάρχει το θέμα της γαλάζιας οικονομίας που μπορεί να φτιαχτεί με βάση τους ωκεανούς μας. Ενέργεια, υλικά, ε, ηχθειοκαλλιέργεια και βιολογικά προϊόντα, όλα αυτά είναι στοιχεία που έχουν σχέση με τους ωκεανούς και θα μπορέσουν να ενισχύσουν και την οικονομική μας πρόοδο. Εάν όμως μεταβαλλόνται τόσο ε, βαθιά οι ωκεανοί και είναι τόσο σημαντικοί για το μέλλον μας, ξέρουμε αρκετά καταλαβαίνουμε αρκετά άραγε για τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Ε, εδώ ακούσαμε να λένε όλοι οι ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μέχρι το 2030 έχουμε μία δεκαετία για τους ωκεανούς, για να αφοσιωθούμε στο θέμα των ωκεανών, να τους καταλάβουμε, να τους μελετήσουμε και να βρούμε λύσεις. Το παράδοξο όμως είναι ότι Ξέρουμε πολύ περισσότερα για το ηλιακό μα σύστημα και το διάστημα από ό,τι για του ωκεανού. Οι ωκεανοί πρέπει να χαρτογραφηθούν πλήρω και δεν γίνονται αρκετά προ στιγμή ε, ούτε διεθνώ ούτε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν το Horizon Europe, θέτοντα ω στρατηγικό τομέα ε, του ωκεανού στι προτεραιότητε του προγράμματο, θα βοηθήσει για του στόχου των φυσικών πόρων. Δεν μπορούν ε, βεβαίω τα ευρωπαϊκά προγράμματα να αντιμετωπίσουν ε, όλε αυτέ τι ανάγκε μόνα του. Χρειάζονται συνδυασμένε προσπάθειε, αλλά ήδη αναφέρθηκε σήμερα το απόγευμα η ανάγκη ευρωπαϊκή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ασχοληθούν με αποστολές έρευνας που θα ε, αφορούν εν μέρη τους καθαρούς ωκεανού και θάλασσες. Και αυτέ οι αποστολές θα αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα. Διότι όχι μόνο θα επιστήσουν την προσοχή των συμπολιτών μας στο θέμα των ωκεανών, αλλά θα αποσχολήσουν και τις ευρωπαϊκές ε, μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Η Ευρώπη πρέπει να καθορίσει τι γραμμή πλεύσης θα ακολουθήσει εμεί τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τι απαντήσεις θα δώσουμε στα προβλήματα των ωκεανών να μένονται λοιπόν από εμά πολύ συγκεκριμένε προτάσει ε, για να πετύχουμε τα αποτελέσματα και με λύσει που θα εφαρμοστούν για να είναι χειροπιαστά τα αποτελέσματα. Η πρώτη φάση ξεκίνησε. Η πρώτη αποστολή έχει μια επιστημονική ατζέντα, όχι μόνο ε, και ερευνητική ατζέντα, όχι μόνο βάσει του Horizon 2020, γιατί εκεί θέλουμε να συντονίσουμε τι προσπάθειε μεταξύ κρατών μελών σε όλη την Ευρώπη και με δημόσιε και ιδιωτικέ ε, συνεργασίε αλλά χρειάζεται όλοι οι φορείς να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια βαθιά αλλαγή, πραγματική αλλαγή, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή την ατζέντα, αυτόν τον κατάλογο προτεραιοτήτων, με την πολιτική για του ωκεανού, όπω είπε και η κυρία Βαλέαν. Διότι δεν μπορεί η έρευνα μόνη τη να αλλάξει τα πράγματα στην πράξη, αλλά η χάραξη πολιτική βάσει των γνώσεων που η έρευνα έχει προηγουμένω προσφέρει και των λύσεων που μπορεί να προτείνει. Αυτά θα κάνουν την πραγματική διαφορά. Να διασυνδέσουμε την έρευνα και την επιστήμη με τι ε, πολιτικέ προτεραιότητε. Αυτό είναι η ουσία. Και αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν και οι ωκεανοί μα και εκεί όπου υπάρχει και συγχρηματοδότηση. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε για του ωκεανού ε, στην μελέτη τη μελλοντική χρηματοδότηση του Horizon 2020. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διαπραγματεύσεων για το Horizon 2020. Θα ολοκληρωθεί μάλλον τι επόμενε ώρε η σχετική διαπραγμάτευση για το Horizon 2020. Και όσοι ε, ενδιαφέρονται για το θέμα των ωκεανών, α ενώσουν τι δυνάμει του για να συζητήσουν τι προτεραιότητε του ορίζοντα 2020 για την ερχόμενη χρονιά. Οπότε όταν άρχισε να τρέχει στι αρχέ του 2021 το πρόγραμμα αυτό, να ξέρουμε ποιε είναι οι προτεραιότητε που πρέπει να κάνουμε για αυτέ. Η Ευρώπη είναι ναυτική, είναι θαλάσσια. Έχουμε τη μεγαλύτερη ακτή παγκοσμίω, 68.000 χιλιόμετρα. Δυο φορέ περισσότερα από τη Ρωσία και τρει από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, έχουμε τον πολιτισμό και την κουλτούρα μα να βασίζονται στου ωκεανού. Είμαστε μια ένωση ωκεανών. Και εδώ τα προγράμματά μα θα πρέπει να συνδυαστούν με φιλοδοξότερε κρατικέ και δημόσιε πολιτικέ. Οι ωκεανοί βρίσκονται στην καρδιά του περιβαλλοντό μα. Ευχαριστώ. Okay, okay, understood. Um, okay, Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πακή. To madam Drake. Και με χαρά θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τζέικ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλεάν για την ευκαιρία που μου δίνετε ο πλανήτης μας καλύπτεται κυρίως από τη θάλασσα. Ε, άρα ε, η καλή κατάσταση των θαλασσών είναι απαραίτητη για την ίδια τη ζωή ε, στη γη. Το είπαν πολλοί προλύσαντες και ο Ζαν τώρα μόλις. Σήμερα όμως έχουμε έρθει εδώ για να αποτυπώσουμε ε, την κατάσταση, τι έχουμε κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωρίσουμε πού βρισκόμαστε και τι απομένει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Η θάλασσα πάνω απ' όλα είναι η πηγή ε, πολλών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που παράγουν υπηρεσίες και αποφέρουν πόρους από τους οποίους τόσο πολύ σήμερα εξαρτώμαστε. Ωστόσο αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες είτε είναι αλληλεία, ναυτιλία, γεωργία, ενέργεια και πολλές ακόμα ασκούν πιέσεις στη θαλάσσια ζωή, στους οικοτόπους και απειλούν πολλές φορές την πρωταρχική ε, λειτουργία των ωκεανών μας, που είναι να διαφυλάξουν και να διατηρήσουν ζωντανό τον ίδιο τον πλανήτη μας. Πολύ συχνά ε, είμαστε πολύ φιλόδοξοι, έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και σεμνινόμαστε γι' αυτό, γιατί όντως πρέπει να είναι καθολικό, προστατευτικό και να μπορεί να εφαρμόζεται. Όλοι αυτοί είναι στόχοι ένα πλαίσιο για την αλία, για το περιβάλλον ε, και ε, ε, καθώς επίσης με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις όλα αυτά συνδέονται και συνδυάζονται. Μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά χάρη σε αυτό το πλαίσιο ενωμένα τα κράτη-μέλη προοδευτικά κάνουν κάποιες βελτιώσεις έτσι ώστε να φτάσουμε στους στόχους. Βήματα ε, για να είμαστε ε, πιο συντονισμένοι και με στρατηγική να προστατεύουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Ας πούμε, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να έχουν μια καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, δηλαδή μέχρι το 2020 θάλασσες καθαρές, παραγωγικές και υγιείς. Ε, αν δούμε όμως τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος, αν αποτυπώσουμε την κατάσταση, απομένουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν. Και είναι μάλλον απίθανο να είναι σε καλή κατάσταση το περιβάλλον ε, ε, παντού και πουθενά και για όλα αυτά τα θέματα μέχρι το 2020. Αυτό επίση αντανακλά τη συνολική εικόνα των ωκεανών που βρίσκονται σε ανισχυτική κατάσταση. Ε, βέβαια όλα είναι προβλήματα εφαρμογής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τόνισε αυτό επανειλημμένα σε διάφορες εκθέσεις. Ε, αυτό όμως οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Και οι άλλοι παράγοντες ποιοι είναι, για παράδειγμα. Χρειάζεται περισσότερη καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε αποτελέσματα επιτόπου. Επιτρέψτε μου εδώ να σας αναφέρω το παράδειγμα των πλαστικών μιας χρήσης προηγήθηκε το πρώτο πάνελ που αναφέρθηκε στη διακυβέρνηση, που και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Δεν θα επιμείνω τώρα σε αυτό. Η περιφερειακή συνεργασία είναι βεβαίως κομβική σημασία για ε, την επιρροή μας στη θάλασσα, όπως είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρήπανση και η απώλεια της βιοπικιλότητας είναι αχαλήνοτη. Εμείς έχουμε εισβάλλει στη θαλάσσια ζωή με τις δικές μας δραστηριότητες, υποβαθμίζουμε το πολύτιμο οικοσύστημα και τους οικοτόπους, αλλά δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ε, τα οικοσυστήματα και να ε, βοηθήσουμε ε, να ανακτώνται τα είδη και να αναπαράγονται αν ορίσουμε προστατευόμενες περιοχές για τη θαλάσσια ζωή. Άσυλα. Ε, χάρη στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των θαλασσών, τώρα έχουμε περίπου, περίπου 11% των θαλασσών να καλύπτονται, ενώ παγκοσμίω αυτό το ποσοστό είναι στο 7%. Χρειαζόμαστε όμως μια ε, γερή όθηση για να γίνεται σωστή διαχείριση με σωστά μέτρα συντήρησης και διαχειριστικά σχέδια έτσι ώστε να έχουμε και οικολογικά ωφέλη και κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη. Τα απορρίμματα, τα απόβλητα στη θάλασσα είναι σύμβολο της ε, αναπαραγωγικής και αναποτελεσματικής μας οικονομίας. Τα ρίχνουμε στη θάλασσα και στις ακτές τα σκουπίδια αντί να τα ανακυκλώνουμε και να τα επαναχρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια βάση ε, στους λιμένες για την καταπολέμηση της ρήπανσης των θαλασσών από πλαστικά. Ωστόσο, ε, ε, επίκυνται και άλλες προσπάθειες. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν γενικά την οικονομία και την ε, ποιότητα της ανακύκλωσης των πλαστικών. Έχουμε νομοθεσία για την μία χρήση για αλευτικά εργαλεία που χάνονται στη θάλασσα και επίσης Έχουμε βελτιωμένους κανόνες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων. Γνωρίζουμε όμως αρκετά για τη θάλασσα, τα είπε ο Ζαν Ερίκ προηγουμένως. Προφανώς υπάρχουν κενά γνώσεις που θα πρέπει να καλύψουμε και εδώ ε, αυτό αφορά την αλία, τα ίδια τα απόβλητα στη θάλασσα, το θόρυβο στο βυθό, τον υποβρύχιο θόρυβο και ε, ε, την καινοτομία και τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα και για τις υδατοκαλλιέργειες. Τέλος, είναι ε, σίγουρα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι γίνονται τόσο πολλά για τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Επίσης, μπορούν ακόμα να γίνουν πολύ περισσότερα και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από κοινού φωτίζουμε αυτή την πτυχή, τις απειλές και τις ευκαιρίες. Θα πρέπει από κοινού να δούμε πώς θα προστατεύουμε τους ωκεανούς, πώς θα δρούμε, πώς θα δρέπουμε τους καρπούς όλοι και πώς θα σεβόμαστε τους ωκεανούς γιατί πραγματικά αξίζουν τόσο πολύ το σεβασμό μας. Thank you. Ευχαριστώ πολύ και τώρα με χαρά ανακοινώνω ότι θα πάρει το λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος Αντώνιο Ταγιάννη. Ζητώ συγγνώμη. Θα πρέπει να κατέβουμε στην πρώτη σειρά των εδρών και θα επανέλθουμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ημικύκλιο του Ευρωκοινοβουλίου. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Κιασίνε Μέσνερ, ειδική επιτετραμένη του Ευρωκοινοβουλίου μας για τις θαλάσσιες υποθέσεις. Βρίσκεστε στην καρδιά της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης και είστε και ο διευθυνονού, ο κύριο Βέλα, ο κύριο Μουέδας, ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, ο κ. Καντέκ, ο πρόεδρο τη Επιτροπή Αλία, η κ. Βάλεαν, εκπρόσωπο τη Επιτροπή ΕΜΒΗ, ο κ. Χένκελ, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ήτρε. Για μένα είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε να υποδεχόμαστε στο υποκύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω από χίλιε πολίτε, ερευνητέ, επιστήμονε, πολιτικού ηθήνοντε, επιχειρηματίε και εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και των ενώσεών τη. Στην αρχή τη θητεία μα διοργανώσαμε 11 ε, συνόδου διασκέψει υψηλού επίπεδου μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτική κληρονομιά, την Αφρική, την ε, ψηφιακή κοινωνική διάσταση, τη μετανάστευση και το καθεξής. Ήρθαν πολίτες, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, ενώσεις, φορείς για θέματα που είναι κέρια σημασία για την Ευρώπη και τους πολίτες μας. Σήμερα θελήσαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα ύψης της σημασίας. Το μέλλον των ωκεανών μας. Πρόκειται για μια ε, σύνοδο που θελήσαμε με μεγάλη αποφασιστικότητα να διοργανώσουμε και ευχαριστώ και την ε, δική μου ε, υπετετραμένη την ε, κυρία Μάισνερ για την διοργάνωση και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε, λέγαμε πριν τις ευρωεκλογέ. Το συζητάγαμε διαρκώ. Ένα γεγονό τέτοια σημασία. Δεν μπορούσαμε να μην επιμείνουμε στη διοργάνωσή του. Είναι για το περιβάλλον, είναι για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, τα πλαστικά. Είμαστε στην πρώτη γραμμή στην προστοφυλακή. Για να εξασφαλίσουμε το μέλλον του πλανήτη μας πρέπει εμείς οι κυβερνώντες να είμαστε σε θέση να δράσουμε χωρίς να χάνουμε χρόνο. Η ε, διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η περιβαλλοντική της διεύθυνση πρέπει να είναι υπόδειγμα για όλους τους διεθνείς παράγοντες. Θέλουμε περισσότερες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος για να αναλάβουν την, κοινωνική τους, την κοινωνική ευθύνη, να προωθήσουν την καινοτομία, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε ένα σημαντικότατο ψήφισμα το οποίο ε, βλέπει θετικά την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν καθαρό πλανήτη για όλους. Θέλουμε μια οικονομία σε άνθηση, σύγχρονη, ε, περιβαλλοντικά ουδέτερη. Θέλουμε την απαλλαγή από τον άνθρακα με το στόχο μηδενικών εκπομπών ε, και τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου στο 2050 παροτρύνουμε τα κατημέλη να αναλάβουν δεσμεύσει για να πετύχουν το στόχο αυτό. Ε, αναγνωρίζουμε όμω ότι υπάρχουν και κίνδυνοι από τι κλιματικέ αλλαγέ. Βάσει του Ευρωπαϊκού Οργανού Περιβάλλοντο, μεταξύ του 2010 και 2016, οι μέγιστε απώλειε τη Ένωση λόγω των μετεωρολογικών και ακραίων καιρικών συνθήκων έφτασαν τα 12 δι ευρώ, 8. Εάν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα, και με υψηλές εκπομπές ε, το ετήσιο κόστος των πλημμυρών μπορεί να φτάσει τα χίλια δις ευρώ μέχρι το 2020 μέχρι το 2100. Μέχρι το 2030 το 50% των ακατοικούμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειψιδρίας. Γι' αυτό χρειάζεται μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση για να συμπεριληφθούν τα περιβαλλοντικά θέματα σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης, Συμπεριλαμβανομένη της ε, πολιτικής μας για το εμπόριο. Όλες οι εμπορικές μας συμφωνίες θα πρέπει να ε, είναι πλήρως συμβατές με τη Συμφωνία των Παρισίων είτε για να βελτιώσουμε τη διεθνή δράση κατά των κλιματικών αλλαγών, είτε για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν συνθήκες ε, και όροι ισοτιμία στη δράση των επιχειρηματιών μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά μα ε, διεθνώ και όλε μα προσπάθειε για το κλίμα, για την οικονομία να ενισχύονται ε, αμοιβαίω. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τι λύσει για το περιβάλλον, για την ψηφιακή μα δράση, για την καθαρή ενέργεια, να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τι μελλοντικέ δεξιότητε και να δημιουργήσουμε εκατομμύρια θέσει εργασία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε με αυτόν τον τρόπο τους ωκεανούς και να τους ρηπαίνουμε. Θα πρέπει την ευφυή χρήση των ωκεανών και την πάυση της ρηπανσής να τους θέσουμε μεταξύ των στόχων της χιλιαρτίας του ΟΗΕ. Είμαστε μεταξύ των πρώτων που ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Στην διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς, τον Ιούνιο πριν από δύο χρόνια, ε, μπορέσαμε να καθορίσουμε 19 σοβαρούς στόχους, φιλόδοξους στόχους για να σταματήσει η απόρριψη από στη θάλασσα, να παρακολουθείτε η κατάσταση των υδάτων και να προχωρήσουμε στη διακυβέρνηση των ωκεανών. Θέλουμε νομοθετικά εργαλεία διεθνού επίπεδου ε, για την βιοπικιλότητα στη θάλασσα και την παράνομη ηλία. Θέλουμε ένα μοναδικό νομοθετικό πλαίσιο για όλες τις δράσεις που έχουν σχέση με τους ωκεανούς. Σήμερα έχουμε πάνω από 150 εκατομμύρια τόνου ωκεανούς, πλαστικού στους ωκεανούς μας. Κάθε χρόνο καταλήγουν στη θάλασσα επιπλέον 8 τόνοι. 8 εκατομμύρια τόνοι. Ε, με αυτό το ρυθμό μέχρι το 2050 στις θάλασσες θα έχουμε περισσότερα πλαστικά από τη ψάρια είναι μια ζημιά περιβαλλοντική αλλά και οικονομική γιατί πλήττει τον τουρισμό και την ε, αλία. Το 70% των ε, αντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα, των ε, διαφόρων προϊόντων είναι μιας χρήσης. Γι' αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση τέτοιων πλαστικών μέχρι το 2021. Αυτό ζήτησε το Κοινοβούλιο. Το πακέτο μα για την ε, κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε την περσινή χρονιά αλλάζει τον τρόπο παραγωγή μα. Θέλουμε ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή του που είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον. Εάν ανακυκλώσουμε ένα εκατομμύριο τόνων πλαστικού, θα απαλλάξουμε του δρόμου μα. Είναι μάλλον σαν να, να βγάζουμε του δρόμου μα ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα. Την, περασμένη εβδομάδα στην Αυλομέλεια του Στρασβούργου εγκρίναμε μια οδηγία που δεν θεωρεί αυτομάτω ω παραγωγό έναν αλία ο οποίος ε, φέρνει και ε, εκφορτώνει απόβλητα που τυχαίως πιάστηκαν στα δίχτυα του. Έτσι μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της αποκομιδής και δίνουμε τη δυνατότητα να μην ε, μένουν τόσα πολλά απόβλητα στις θάλασσες. Δίνουμε κίνητρο στα σκάφη να ασχολούνται με τα ίδια τους τα απόβλητα και την αποκομιδή τους και να τα πηγαίνουν στα λιμάνια όπου θα δημιουργηθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις. Γι' αυτό ελπίζω τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν θα δυνατόν πιο γρήγορα αυτή την οδηγία. Με περίπου 5,5 εκατομμύρια εργαζομένου, υποστηθέμενη αξία των 500 δι ευρώ ετησίω, η γαλάζια οικονομία είναι προφανώ κέρια σημασία για την Ευρώπη. Κάποιοι τομεί όμω έχουν και άλλα περιθώρια ανάπτυξη. Σήμερα το 75% του εξωτερικού μα εμπορίου και το 37% των συναλλαγών στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά γίνονται μέσω θαλάσση. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία για να έχουμε θαλάσσιε μεταφορέ που να είναι αποτελεσματικότερε. Ο νέο προπολογισμό τη Ένωση για το 2021 έω 2027 θα πρέπει να προβλέπει μέτρα υποστήριξη αυτού του σκοπού, αυτή τη στρατηγική. Οι καθαρέ θάλασσε και οι καθαρέ ακτέ θα πρέπει να είναι κριτήρια δύναμη τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, είναι ένα πόρο οικονομικού, εμπορικού και τουριστικού χαρακτήρα, μοναδικό παγκοσμίω. Σε ό,τι αφορά την μηχανή τη Αλία, αυτή προσφέρει στου Ευρωπαίου καταναλωτέ περίπου 6,5 εκατομμύρια τόνο ψαριού ετησίω και δίνει δουλειά σε 350.000 Ευρωπαίου. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον τομέα τη αλεία και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία. Θα πρέπει <clears throat> να διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην βιώσιμη αλεία. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει, σε όλη αυτή τη θητεία μάλλον, εργαστήκαμε για τον κανονισμό, για την συλλογή δεδομένων και αυτόν για, την για τον εξωτερικό μας στόλο, τον εξωενωσιακό. Ε, για να ολοκληρώσω, πολλές ευρωπαϊκές ε, ανακαλύψεις και προτάσεις και πρωτοποριακά βήματα ήταν αποφασιστικά για την διαφύλαξη του πλανήτη, όπω ε, τα βιοδιασπόμενα πλαστικά, τα ανακυκλώσιμα υλικά και η τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών. Με το πρόγραμμα Κοπέρνικο ε, συγκεντρώσαμε θεμελιώδη στοιχεία για να καταλάβουμε καλύτερα τον πλανήτη μα και να μπορούμε να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Να γιατί η διαστημική πολιτική χρησιμεύει και για να προασπιστούμε τη φυσική μας κληρονομιά, να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να έχουμε καλή και σωστή διαφύλαξη του πλανήτη. Οι υπηρεσίε του Κοπέρνικου είναι ένα σημαντικό πόρο για την διαχείριση των αστικών περιοχών, την βιωσιμή ανάπτυξη, την προστασία τη φύση, τον περιφερειακό χωροτοξιακό σχεδιασμό, τη γεωργία, την αλεία, την υγεία, την ε, προστασία των πολιτών, τι οικοδομέ, τι ε, μεταφορέ και τον τουρισμό. Γι' αυτό ζητάμε μεγαλύτερε προσπάθειε ε, και περισσότερε επενδύσει για καινοτομία και έρευνα. Είναι αλήθεια ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει αύξηση στο πακέτο αυτό που ήταν ορίζοντα 2020 και τώρα θα ονομάζεται ορίζοντα Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε φιλοδοξότεροι. Η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου προβλέπει κι άλλη αύξηση επιπλέον σε αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήσαμε από το 50% να φτάσουμε στα 120 δις ευρώ και ζητήσαμε το 30% όλων των δράσεων προβλέποντας τον επόμενο προπολογισμό της Ένωσης, ε, δηλαδή το 35% του ορίζοντα Ευρώπη, να αφορά μέτρα βιωσιμότητας. Για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις οικονομίες κλίμακας και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να έχουμε κοινού πόρους στο ύψος των προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Και επιμένω, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο. Δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από την Ευρώπη και να λένε ότι είναι δικό μας το φταίξιμο. Τώρα πρέπει να, ε, παίξουν το, να πάρουν μέρος στο παιχνίδι αυτό και τα κράτη-μέλη. Το περιβάλλον, η έρευνα, η καινοτομία, η βιομηχανία, η βιομηχανία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένε. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι ενώσει και επιχειρήσει είναι το κλειδί για, την ε, ε, για το σωστό συνδυασμό περιβάλλοντο και καινοτόμου ανταγωνιστική ε, οικονομία. Θέλουμε μια Ευρώπη που να είναι φίλη των ωκεανών. Θέλουμε να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο και από την σκοπιά τη ε, περιβαλλοντική διπλωματία, όπω κάναμε με την COP24 στο Κατόβιτσα το Δεκέμβρη, και με συγκεκριμένε δεσμεύσει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια όλων σα. Είναι μια πρόκληση που καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε και να την κερδίσουμε μαζί, να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Ε, οι ευχαριστίε μου, οι ευχαριστίε όλου αυτού του κοινοβουλίου πηγαίνουν και κατευθύνονται προ εσά. Εσά που δώσατε αυτέ τι μάχε. Η δική μου η δέσμευση προ του συναδέλφου του κοινοβουλίου είναι ότι μπορείτε και όλων μάλλον των συναδέλφων του Κοινοβουλίου ότι μπορείτε πάντοτε να υπολογίζετε σε εμά και στην υποστήριξή μα. Σα ευχαριστώ. Okay, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο πάνελ. Είχαμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε την αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ε, Γενική Διευθύνση για το Περιβάλλον, την κυρία Ντρέικ. Τώρα να δώσω το λόγο στου επόμενου ομιλητέ. Ε, είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ασχοληθεί με το θέμα θα ξεκινήσω με τον Μάρκ Ντέμεσμάκερ, αλλά θα πρέπει να σας ζητήσω να περιοριστείτε στα τρία λεπτά. Αυτό απαιτεί η οργάνωση της διάσκεψης. Παρακαλώ τρία λεπτά κύριε Ντεμεσμάκερ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Στα αγγλικά, καλησπέρα σε όλους σας. MEP for ECR Group. Είμαι ευρωβουλευτής από την ομάδα ECR Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας. Ασχολούμουν σε αυτή τη θητεία με όλα τα θέματα της κυκλικής οικονομίας και το, τη νέα ρύθμιση για τα πλαστικά μιας χρήσης. Πολλά ε, ακούστηκαν ήδη. Το πλαστικά είναι ένα υλικό πολύτιμο και χρήσιμο και έχουν τη θέση τους στην κοινωνία μας. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε πλαστικά σήμερα είναι και αφορητός αλλά και πανάκριβος. Επιπλέον, η ανακύκλωση πλαστικών και η συλλογή τους παραμένει πολύ χαμηλή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 5% της αξίας των συσκευασιών, των πλαστικών συσκευασιών παραμένουν στην οικονομία μας. Άρα το 95% της αξίας χάνεται. Και είναι βασική πρόκληση να διαχειριζόμαστε τα πλαστικά με τρόπο βιώσιμο όσο και ε, υπεύθυνο σε όλη την αλυσίδα. Η στρατηγική για τα πλαστικά θα πρέπει να είναι μοχλός για να ενθαρρύνει και να κινητροδοτεί για νέα μοντέλα, για νέες λύσεις, ε, κοινέ δεσμεύσεις και δράσεις από όλους τους ε, ενεχομένους την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία όχι απλώς να τα ξαναπούμε αλλά να προχωρήσουμε και σε δράσεις. Θα δούμε τι θα βγει από τον τριμερή διάλογο και τη συμφωνία για τα πλαστικά μιας χρήσης ε, στον οποίο κατέληξαν μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις το Δεκέμβριο ε, που δεν θα ξεχάσω ποτέ ούτε εγώ ούτε ο Επίτροπος Βέλα. Πάντω ήταν καλό το αποτέλεσμα και είμαι πεπισμένο ότι αυτή η νομοθεσία είναι κρίσιμη για τη μετάβασή μα προ την κυκλική οικονομία, αλλά και προ ένα βήμα στο να κρατήσουμε τα απορρίμματα αυτά τα πλαστικά μακριά από τι θάλασσε τα πελάγια και του ωκεανού μα. Ιδιαίτερα τα πλαστικά απόβλητα είναι μεγάλο πρόβλημα πέρα από τα υπόλοιπα σκουπίδια για τι θάλασσε και του ωκεανού. Και όπως είπε και ο πρόεδρο, πρέπει να αποφύγουμε να καταλήγουν στη θάλασσα τελικά, ε, να έχουμε περισσότερα πλαστικά ψάρια η στο μέλλον. η δέσμη ε, μιλάει για τα 10 κοινότερα ε, προϊόντα πλαστικών που βρίσκουμε στις ακτές μας στην Ευρώπη και το Κοινοβούλιο χαίρεται που θα απογορευθούν ε, τα προϊόντα ε, από όξο αποσπόμενα πλαστικά. Το θέμα είναι ότι δεν, δεν ε, ε, διαλύονται αυτά, αλλά γίνονται ε, πάρα πολύ μικρά σωματίδια πλαστικού. Τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να μειώσουν τους πλαστικούς περιέκτες τροφίμων και τα πλαστικά κυπελάκια μιας χρήσης, ποτήρια δηλαδή. Επίσης το κόστος καθαρισμού είναι πολύ μεγάλο και δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Έχουμε δεσμευτικό στόχο για ε, ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών ποτών μέχρι ε, το 2029 κατά 90%. Τα πλαστικά μπουκάλια ε, αναψυκτικών ποτών και τα λοιπά είναι αυτά που βρίσκουμε περισσότερο στις ακτές μας. Και καταφέραμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη μέχρι το 2030 μέχρι το 2030 να είναι το 30% ανακύκλωσιμο προϊόν στις συσκευασίες. Επίσης, τα πλαστικά φίλτρα τσιγάρων είναι το, το δεύτερο μετά τα μπουκάλια ε, που βρίσκουμε. Μέχρι 500 λίτρα νερού μπορεί να ρυπάνει μία πλαστική γόπα από τσιγάρο και θα πρέπει οι καπνοβιομήχανοι να τα ξέρουν αυτά και να ε, πληρώνουν το κόστος της συλλογής σε δημόσιους χώρους. Είναι σίγουρα μια πολιτική συγκυρία πάρα πολύ σημαντική, την υποστηρίζουν οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών για να περάσουμε σε μια μετάβαση, σε μια κυκλική οικονομία με ανακύκλωση πλαστικών. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε αυτές τις οδηγίες και η μετάβαση ε, στην κυκλική οικονομία θα μας κάνει να κάνουμε τις χωματερές χρυσορυχία. Και τελικά αυτή η σούπα των πλαστικών στους ωκεανούς μπορεί να γίνει ένα τεράστιο γαλάζιο λιβάδι. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρικάρτο Σερόσεντος, ο οποίο είναι μέλο τη Επιτροπή Αλίας. Ελπίζω να μείνετε στα τρία λεπτά. Ο κύριος μου είχε δώσει υπόσχεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν 20 ε, χρόνια, ε, Πορτογαλός ε, ποιητής εδώ εκείνησε το φεστιβάλ του Σιροπαρλιά και είπε στη γλώσσα μου μπορώ να ονειρευτώ τη θάλασσα. Θα μιλήσω πορτογαλικά λοιπόν. ο Homo sapiens ε, με συνεχή και προοδευτικό τρόπο και στη συνέχεια με επιταχυμένο τρόπο και στη συνέχεια με στιγμίο τρόπο τον 20ο αιώνα έγινε, στην, ε, μετατράπηκε στην κύρια μετασχηματιστική δύναμη της γεωλογίας του πλανήτη που μας ε, οδήγησε στο να μπούμε σε μια νέα γεωλογική εποχή, το ανθρωπόκαινο δεκάδες επιταχυμένης ανάπτυξης και βιομηχανική κοινοτομία μα έκαναν να ξεπεράσουμε τουλάχιστον 4 από τα 9 όρια του πλανήτη. Οι θάλασσες και ωκεανοί που είναι στοιχεία σταθεροποιητικά για βιοκαιοφυσικών διαδικασιών και κυρίω ρυθμίζουν το κύκλο του άνθρακα σήμερα είναι αποδυναμωμένε τα προβλήματα πάνε πολύ πέρα από την υπερελίευση και από τη ρήπανση και τα χωροκατακτητικά είδη υποφέρουν και από οξύνηση, από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και πολλοί από αυτούς τους παράγοντες ελοπιδρούν με άλλους συνυπάρχοντες παράγοντες όπως η αύξηση του επίπεδου του νερού της θάλασσας, η απώλεια βιοπικιλότητας και η αύξηση περιοχών χωρίς οξυγόνο και πολλά από αυτά τα προβλήματα μπορεί να φαίνονται περιφερειακά και σίγουρα υπάρχουν τέτοια περιφερειακά ζητήματα. Το γεγονό είναι ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, από μια παγκόσμια σκοπιά. Ε, ο αντίκτυπο των ανθρώπου ε, πάνω στο θαλάσσιο συνστόσο του πλανήτη δεν έχει πολιτικά σύνορα. Οποιαδήποτε απάντηση είτε σε χώρια ύδατα είτε στην ανοιχτή θάλασσα θα πρέπει να γίνει από κοινέ πολιτικέ. Η παγκόσμια διακυβέρνηση και η τεχνική επιστημονική γνώση είναι οι πυλώνε για ένα βιώσιμο μέλλον. Χρειαζόμαστε συντονισμένα προγράμματα στις θαλάσσιες επιστήμες για να καταλάβουμε το ρόλο των ε, ωκεανών. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ένα στόχο marketing. πρέπει να είναι μια δέσμευση που θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να λάβει υπόψη τα διάφορα επίπεδα ανάπτυξη μεταξύ περιοχών και χωρών. Ε, οι χώρε που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ε, για να έχουν χειρότερε περιβαλλοντικέ συνθήκε είναι οι λιγότερο αναπτυγμένε. Όμω αυτοί συνεισέφεραν λιγότερο στην κατάσταση του πλανήτη. Πρέπει να έχουμε προοδευτική και συνεχή εστίαση στην παιδεία, στην κατάρτιση και στην έρευνα για να επιτρέψουμε ότι η νέα γενιά ε, των διαχειριστών των ωκεανών ε, ε, ασκούν τα δικαιώματά τους και τα καθήκοντά τους με μεγαλύτερη υπευθυνότητα για έναν υγιή ωκεανό. Ε, συνεχίζει να λειτουργεί το ρολόι και δεν έχουμε ωραίες ε, ατράκτους. Μπορούμε να καταλήξουμε σε γενοκτονία για ορισμένε περιοχές του ωκεανού και κατόπιν ε, για τον πολιτισμό μας. Στη συνέχεια ε, πρέπει η, να έχουμε την ηθική ευθύνη μια γενιά ε, που κινητοποιείται. Σας ευχαριστώ αυτή τη νέα γενιά, αποτελεί ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ και που σεβαστήκατε και το χρόνο. Τώρα, η επόμενη ομιλήτρια είναι η Κλαούδια Μοντέριο Ντεαγκιάρ, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών. Έχετε τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους παρόντες και τους επιτρόπους και δεν μπορώ παρά ανακλέψω κάποια δευτερόλεπτα από τα τρία λεπτά για να απευθυνθώ και να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ για όλη τη δέσμευσή της και το έργο της ε, για το γαλάζιο κόσμο, για τον κόσμο των θαλασσών και των ωκεανών. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σεράου Σέντος, ε, παρά τις πολιτικές διαφορές που προσχωρίζουν. Είναι ένας ε, Πορτογάλος, ο οποίος χάραξε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο στον τομέα της θάλασσας και κατόπιν πρέπει να καταλευτούμε όλες αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι ωκεανοί καθώς ε, βρίσκονται ε, σε προτεραιότητα του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίω ε, για να το προωθήσουμε στις επόμενες ευρωεκλογέ. Πρέπει να δείξουμε ότι ανησυχούμε για την κατάσταση αυτή, ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν αποδείξει ότι θέλουν να δράσουν απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται και επίσης να ε, απαριθμίσουμε όλους τους ακτιβιστές που αναφέρθηκαν εδώ. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, τον David Attenborough το, με το πρόγραμμά του στο BBC ε, ευαισθητοποιεί για να εργαστούμε περισσότερο για αυτή την προβληματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των πλαστικών στους ωκεανούς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες προκλήσεις πρέπει να συνεχίσουμε να προτείνουμε στρατηγικές ε, προσερμογής, μακροπρόθεσμες για την καταπολέμηση των απορριμμάτων αλλά και την κλιματική αλλαγή. 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω ε, δαπανούμε για τι θαλάσσιε έρευνε, προωθώντα νέε υπηρεσίε και νέα προϊόντα για την γαλάζια οικονομία. Ε, Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται περισσότερες επιστημονικές γνώσεις και στοιχεία που να αναλύουν περισσότερο το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Ρίζων Ευρώπης ε, ε, θα παρέμβει στους ωκεανούς και θέλουμε να μπλοκάρουμε το δυναμικό των θαλασσών. Αυτό μπορεί να είναι το κλειδί για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Όλοι χρειαζόμαστε, είμαστε απαραίτητοι για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις πρέπει να συνεχίσουμε, όπως κάναμε και στην Επιτροπή Μεταφορών, σε μια γνωμοδότησή μας, εκφράζεται αυτό, να συνεχίσουμε τη στρατηγική για να ε, υπερασπίσουμε την περαιτέρω χρήση του γραπημένου φυσικού αερίου, αλλά και να αντικαταστήσουμε ε, τις πηγές ενέργειας που ρηπαίνουν περισσότερο. Θα πρέπει να έχουμε πιο διατομικές προσεγγίσεις και να ε, επικεντρωνόμαστε στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Επίσης, σε αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, θα πρέπει να εστιάσουμε και να αναφερθώ και στις άκρως απομακρυσμένες περιοχές ε, δεδομένου στις τοποθεσίες τους στον Ατλαντικό και στον Ινδικό ωκεανό είναι θεμελιώδης για την μελέτη και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, του αντικτύπου στα θαλασσικά οικοσυστήματα και στη βιοπικιλότητα. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να πω ότι θα προτείνω ένα κέντρο καταπολέμησης της θαλάσσιας ρήπανσης σε αυτές τις άκρως απογνωρισμένες περιοχές πιθανότητα στη Μαδέρα να ιδρυθεί για να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να υιοθετήσουμε τρόπους καταπολέμησης της απειλής και αυτό ε, φυσικά σε συνεργασία με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα που βρίσκεται στην Πορτογαλία. Θα ήθελα να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, στους νέους που είναι παρόντες εδώ. Όλοι να δεσμευτούμε για την καταπολέμηση της, των θαλάσσιων απεριμάτων, αλλά να αγωνιστούμε και για το μέλλον μας, να έχουμε κάθε φορά καλύτερες θάλασσες και ωκεανούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. ακούσουμε τώρα ε, ενδιαφερομένους και ενεχομένους φορείς. Παρακαλώ να συστηθείτε. Uh, ε, το Διευθύνοντα Σύμβουλα ε, της... Ε, ε, του Ιδρύματος για τον ε, Γαλάζιο Ωκεανό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, Επίτροπε Βέλα, ε, πρώην μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, το σύστημα των ωκεανών είναι το πιο ευαίσθητο και ευπαθέ του πλανήτη. Όμω, ο η δυνατότητά του να παράγει βιομάζα, να διατηρήσει τη βιοπικιλότητα ή να παράγει οξυγόνο υποβαθμίζεται ε, διαρκώς. Ως ε, συνέπεια, ο ωκεανός τελικά αλλάζει και ως προς τη βιοχημική του ε, σύνθεση. Αυτό πιέζει τον ωκεανό σε μια βαθιά και τον οδηγεί σε μια βαθιά περιβαλλοντική κρίση, η οποία δεν γίνεται πλέον αρκετά κατανοητή ε, και δεν έχει γίνει ακόμα αρκετά κατανοητή από τον άνθρωπο. Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει προσφέρει αρκετέ ε, λύσει για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα αυτό. Το 2020 θα είναι ορόσημο, χρονιά ορόσημο όχι για την επιτυχία μα, αλλά για τον οργανισμό των ωκεανών που εκπροσωπώ φόβου μπορεί να είναι και ορόσημο δυσαρέσκειας για την έλλειψη εξέβρεση λύσεων. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα είναι πιο ισχυρά μεταξύ των νέων και είναι σαφή οι ενδείξεις της απογοήτευσής τους. Ε, το είδαμε και από τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων τους ε, προηγουμένως. Είναι απαραίτητο λοιπόν να λάβουμε δράση. Ο ΙΕ αυτή τη στιγμή συζητά αυτού της ε, νέα συνόδου που θέλουν να διοργανώσουν Πορτογαλία και η Κένια για το μέλλον των ωκεανών. οι ειδήσει, αλλά δεν είναι το τελευταίο βήμα που μπορούμε να κάνουμε, ε, διότι με την εφαρμογή του στόχου της χιλιετία 14 ε, δεν θα λυθούν τα προβλήματα των ωκεανών. Πρέπει να βρούμε τα κομμάτια του πάζλ και, να, και τη συνολική εικόνα, τη διασύνδεση των κλιματικών αλλαγών με το τι γίνεται στους ωκεανούς ή το μοντέλο οικονομικής μας ανάπτυξης που εξαρτάται από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στον πλανήτη και τον ανητικό αντίκτυπο που έχει αυτό το μοντέλο για τους ωκεανούς. Η διεθνή κοινότητα που εκπροσωπείται από τα μέλη του ΟΗΕ μεταξύ άλλων μπορεί να εγκρίνει στην επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ για τους ωκεανούς μια σχετική συμφωνία, αλλά έχει σοβαρές ευθύνες και η κοινωνία των πολιτών. Η ευθύνη αυτή είναι κάτι που συναισθανόμαστε πλήρως και ο οργανισμός μας προσπαθεί να σώσει ό,τι απομένει στους ωκεανούς προσπαθώντα να προωθήσει νέε προστατευόμενε περιοχέ με βιώσιμε αλληλευτικέ ε, δραστηριότητε και ενισχύοντα μια γαλάζια οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρόμαστε που μπορούμε να σα ανακοινώσουμε ότι η Περιφερειακή Κυβέρνηση των Αζωρών, σε, συνεργασία, σε εταιρική σχέση με, την, ε, με το Ίδρυμα ΟΕΤ και την, ε, τον δικό μα οργανισμό, πριν δύο μήνε, αποφάσισε να αφήσει σε ανάπαυση ένα μεγάλο μέρος τη θαλάσσια ζώνη των Αζωρών και να γίνουν αυτέ προστατευόμενε ε, περιοχέ. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό τη συνολική θαλάσσια έκταση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που εκπροσωπεί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η Πορτογαλία. Είναι τολμηρή και σημαντική απόφαση των Αζωρών, όχι μόνο για το δικό τους το αρχιπέλαγος ή για την Πορτογαλία μόνον, αλλά για ολόκληρο τον βόρειο δυτικό Ατλαντικό ωκεανό, τον βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό. Ο οργανισμός των γαλάζιων ωκεανών δεν πιστεύει ότι θα πετύχουμε να έχουμε γυρέστερους ωκεανούς μόνο με την διαφύλαξή τους. Και η οικονομία μας είναι θέμα. Η δική μας οικονομική ανάπτυξη και το μοντέλο που έχουμε καθορίσει φαίνεται ότι δεν είναι συμβατό με την ε, βιωσιμότητα του πλανήτη. Υπάρχει σοβαρότατη επίγουσα ανάγκη να αλλάξει το μοντέλο αυτό και γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τη φύση με άλλα μάτια. Είναι ένα κεφάλαιο ένα κεφάλαιο φυσικό και στο οποίο βασίζεται η ύπαρξη της κοινωνίας μας. Εάν γίνει κεφάλαιο η φύση, τότε οι δράσεις για να σώσουμε την φύση θα μπορούσε να θεωρηθεί οικονομική κίνηση. Είναι κεφαλαιακή επένδυση, όχι κόστος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το φυσικό κεφάλαιο να θεωρηθεί ως αντικείμενο που θα μπορούσε να το διαχειριστεί μια τράπεζα. Όπως είπε και η κυρία Δαμανάκη με το γαλάζιο ομόλογο ή με τη βιομάζα που με τι νέε προστατευόμενε θαλάσσιε περιοχέ. Κάτι που θα μπορούσε να το υπολογίσει στην τραπεζική του αξία Παγκόσμια Τράπεζα. Παρομοίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυχώ στην ενεργειακή τη πολιτική πρότεινε μέτρα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για μια ατζέντα για του ωκεανού που να προωθεί την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των ωκεανών. Κυρίες και κύριοι, ε, όσο αναβάλουμε ε, την δράση, τόσο πιο ριζοσπαστικές αλλαγές θα χρειαστούν. Οι νέες γενιές δείχνουν ότι δεν έχουν άλλη υπομονή. Ε, ο θυμός θα φουντώσει εάν οι θύνοντες παγκοσμίως δεν λάβουν αν δεν αναλάβουν ευθύνες και δεν αναλάβουν μέτρα για τις θαλάσσιες ε, περιοχές και τα διάφορα αρπακτικά ή τα κοράλια ή ε, για όλα τα είδη που ζουν στη θάλασσα. Πρέπει να σταματήσουμε την περιβαλλοντική υποβάθμιση και να σταματήσει ο φαύλο κύκλο όπου η περιβαλλοντική υποβάθμιση θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική ύφεση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Now I turn to Dr. Vladimir. Ευχαριστώ ο δόκτωρ ε, Βλάντιμιρ ε, ε, Ριάμπινιν, εκτελεστικός γραμματέας της Διακυβερνητικής Οκενογραφικής Επιτροπής και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO. Για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω να σας χαιρετήσω εξ ονόματος της κυρίας Όντρια Ζουλέ, Διευθυντού της UNESCO. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν Υπάρχει μια διάσταση παγκόσμια εδώ, διάσταση των Ηνωμένων Εθνών και θέλω να μιλήσω για το ρόλο της ωκεανογραφίας και της επιστήμης των ωκεανών για το μέλλον. Θέλω να απευθυνθώ στους νόους και να σας πω ότι είναι πραγματικά πολύ σπουδαία επιστήμη αυτή και επάγγελμα και θα βρείτε και δουλειά ε, ε, στον 21ο αιώνα να ασχοληθείτε με αυτά τα θέματα της ε, ωκεανογραφίας. Η Επιτροπή μας έχει ένα ρόλο καθοδήγησης ε, της επιστήμης για τους ωκεανούς από πλευράς ΟΗΕ. Παγκοσμίω. Η Ευρώπη όμως είναι ο υπαριθμόν ένα ηγέτης στην επιστήμη. Είναι τρία τα κέντρα ε, τα ισχυρά. Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και ε, Δυτικός Ειρηνικός. Συνεργαζόμαστε πολύ παραγωγικά και γόνιμα με την Ευρώπη Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης. Ε, υπάρχουν βάσεις δεδομένων στην Ευρώπη, όπως είναι η EMOTNET Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, για τον ειδικό σχεδιασμό για τη θάλασσα, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι το 1 τρίτο των ΑΟΣ παγκοσμίω μέχρι το 2030 να καλύπτεται από εγκεκριμένες από τις κυβερνήσεις ε, ε, προσπάθειες, δράσεις και σχέδια, ειδικά για τη θάλασσα. Συνεργαζόμαστε και με τη Γενική Διεύθυνση Επιστήμης και Έρευνας ε, και θα συνεισφέρει πολύ το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη, Horizon Europe, αλλά και πολλά υποσχόμενα είναι και τα παρατηρητήρια. Πού βρίσκονται επιστήμες των ωκεανών, η ωκεανογραφία. Ε, έχουμε μια πρόσφατη ανάλυση που λέει το εξής. Είναι αρκετά καλή επιστήμη για να φωτίζει ε, την κατάσταση. Ξέρουμε πόσο διοξίδιο του άνθρακα απορροφάει ο ωκεανός, πόσο θερμότητα απορροφάει ο ωκεανός, τι γίνεται με το οξυγόνο, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε καλές λύσεις. Η κατάσταση μας θυμίζει τα όσα συνέβησαν και για το κλίμα το 2008. Υπήρξε η επιστήμη και τα στοιχεία, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία για δράση και ούτε δράση υπήρχε. Και τώρα θα πρέπει να δράσουμε πραγματικά για να μπορέσει η επιστήμη να είναι αποτελεσματική. Η Επιτροπή μας ε, ε, έκανε προτάσεις ε, στον ΟΗΕ ε, για τις επιστήμες των ωκεανών που να προτείνουν λύσεις όμως προσανατολισμένες ε, στην ε, πράξη. Και πραγματικά συμμετέχουν πολλοί και ο κύριος Σάντος. Να σας πω ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι σε διάφορους τομείς να έχουμε ερηξικέλευθες δράσεις, χαρτογράφηση, παρατήρηση, δεδομένα, κατανόηση των οικοσυστημάτων και των μεγάλων βαθών τη δυνατότητα οικοδόμησης ικανοτήτων. Καταλαβαίνετε ε, πώς ε, έτσι αυξάνονται οι γνώσεις μας για τον ωκεανό ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είναι τομές. Είναι πολύ σημαντικά, καλά σχεδιασμένα και θα μπορέσουμε σε πολλούς τομείς να έχουμε ουσιαστικά ωφέλη. Διαχείριση παρακτήων ακτών, ε, προσαρμογή και μετρίαση του, της κλιματικής αλλαγής, ε, χωροταξικός σχεδιασμός στη θάλασσα. Όλα αυτά είναι τομείς δραστηριοτήτων ε, που μας οδηγούν να κάνουμε τους ωκεανούς παραγωγικούς, αποδοτικούς, με μια γαλάζια οικονομία και όχι ε, εις βάρος της υγείας των ωκεανών. Ακριβώς αυτή είναι η ιδέα της ωκεανογραφίας, της επιστήμης των ωκεανών και προσεχώς θα έχουμε μια παγκόσμια ε, διάσκεψη στην Κοπενχάγη το Μάιο. Αναφέρθηκε και ο Τιάγκο προηγουμένως ε, μια διάσκεψη για τις δράσεις που απορρέουν από την επιστήμη και τα δεδομένα. Ελπίζω πάρα πολύ η Ευρώπη να ε, στερνιστεί αυτό το μήνυμα και να βοηθήσει στην ωκεανογραφία και έχουμε για αυτή τη δεκαετία και έχουμε και ένα σλόγγαν «Ωκεανός που χρειαζόμαστε ε, για το μέλλον ε, που θέλουμε». Τώρα μιλάμε για την επιστήμη που χρειαζόμαστε για τον ωκεανό που θέλουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. τα εμπνευστικά τόσα μας είπατε. Και τέλος ε, θα δώσω το λόγο στον Πίτερ Χέρτσικ. Είναι εκτελεστικός διευθυντής ε, στο κέντρο GMR ε, στο Κίελο, στη Γερμανία. Για την έρευνα σου και παρακαλώ, έχετε το λόγο να σας ευχαριστώ Πρόεδρε για το λόγο. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τους καθαρούς ωκεανούς και θάλασσες από τη σκοπιά της έρευνας και θα ξεκινήσω με το 70%. Το ακούσατε πολλές φορές σήμερα. Το 70% καλύπτεται από ε, τους ωκεανούς. Έχουμε την, ε, διάφορους ωκεανούς, την Αυξηνοπόντο, τη Βαλτική, τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Θάλασσα, τον Ειδικό Κενό, τον Ατλαντικό, τον Ελληνικό. Και το 70% λοιπόν του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό ε, από των ωκεανών και γι' αυτό ζούμε σε ένα γαλάζιο πλανήτη. Είναι λοιπόν σημαντική η ωκεανή για μας, όχι μόνο ε, λόγω των μεγεθών τους, αλλά γιατί είναι ένα μεγάλο οικοσύστημα στον πλανήτη. Και έχουμε ακούσει και πάλι ότι υπάρχει πρόβλημα με το οξυγόνο. Παρέχει λοιπόν ο ωκεανό το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε και αυτό οφείλεται στη δραστηριότητα των μικροοργανισμών στον ωκεανό. Αν δεν μας κάνουν αυτή τη χάρη, δεν θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε, δεν θα ήμασταν εδώ σε αυτή την αίθουσα. Αυτό αποτελεί λοιπόν σημαντική λειτουργία και υπηρεσία των ωκεανών. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν, μάλλον απορροφούν το 30% των εκπομπών του άνθρακα από την αρχή της βιομηχανικής εποχής και το 30% σημαίνει ότι δεν θα μιλούσαμε σήμερα για το στόχο 1,5-2% ενώ θα ήμασταν σε μια πραγματικότητα 4-5 βαθμών Κελσίου. Μας έχει κάνει μεγάλη χάρη λοιπόν ο Γένος και πάλι εδώ, αλλά ε, ξέρετε... Ε, το ότι απορροφάτε το διοξείδιο του άνθρακα του ωκεανού ε, ουσιαστικά έχει και ένα τίμημα, προκαλεί τοξίνηση. Επίσης ε, και και ενός ε, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θερμότητας που παράγουμε και επίσης παρέχει τροφή για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η ωκεανοί είναι ζωτική για μας, το ακούσαμε και στο παρελθόν. Ο ωκεανός ε, ουσιαστικά αποτελεί το σύστημα στήριξη ζωή του πλανήτη. Πρόκειται για έναν ασθενή όμως την εντατική αλλά δεν είμαστε καλοί γιατροί, δεν προσέχουμε τους ωκεανούς μας, γιατί ε, εδώ με την πίεση που βάλουμε στους ωκεανούς ε, προκαλούμε οξύνηση στους ωκεανούς και φερούμε το οξυγόνο, αυξάνονται οι περιοχές που έχουν ελέγξει το οξυγόνο σε πολλές περιοχές του πλανήτη, αυξήνουμε την ε, θερμότητα των ωκεανών, ρηπαίνουμε τους ωκεανούς, τα πλαστικά. Ε, είναι ένας παράγοντα νικής, αλλά έχουμε και χημικού τύπου ρήπανση, βιολογικού τύπου ρήπανση. Επίσης, ε, ζημιώνουμε την βιοπικιλότητα των ωκεανών. Δεν έχουμε καν ανακαλύψει όλη τη βιοπικιλότητα, αλλά έχουμε προκαλέσει βλάβη σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτή. Αναφέρθηκε και η υπεραλίευση και το θέμα των χωροκατακτητικών ειδών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα βλέπουμε σήμερα, όμως υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα που ανακύπτει το 2050 θα έχουμε 50% περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη, δηλαδή 10 με 10,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι το 50% περισσότεροι άνθρωποι θα χρειάζονται 50% περισσότερα τρόφιμα, περισσότερη ενέργεια και 50% περισσότερους πόρους. Και κάποια θα πρέπει να έρθουν από τους ωκεανούς κάποια από αυτά. Έτσι λοιπόν η πίεση στους ωκεανούς αυξάνεται ε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα γη ωκεανό για υγιεί ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτό απαιτεί περισσότερη έρευνα που να προσανατολίζεται στη λύση. Η βασική έρευνα αποτελεί τη βάση, αλλά χρειαζόμαστε έρευνα που να προσανατολίζεται σε λύση, μεγαλύτερο συντονισμό της έρευνα και πιο στοχευμένη χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουμε να τάσουμε σε προϊόντα και δράσει. Η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα τη σωτηρία των ωκεανών μας για τις επόμενες γενιές στον πλανήτη. Νομίζω ότι αυτό έχει αναφερθεί και στο παρελθόν και θα ήθελα να είμαι κάπως πιο κλητικός στο σημείο αυτό γιατί πάντοτε αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τους ωκεανούς. Καθώς αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα και αφιερώσαμε όλο το απόγευμα σήμερα στη συζήτησή του, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ίσως λοιπόν θα χρειάζεται περισσότερη προβολή, περισσότερη ηγετική στάση και δράση από την ευρωπαϊκή πλευρά όταν ε, μιλάμε για τη διάσωση των ωκεανών μα και των θαλασσών μα. Σα ευχαριστώ. Well, thank you very much. We have now... Ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε στο τέλος του πάνελ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας που προσπάθησαν να μας δώσουν μια συνολική εικόνα του τι είναι το διακύβευμα τι μπορούμε να κάνουμε για τη διαφύλαξη των ωκεανών μας, πόσο σοβαρά παίρνουμε το θέμα αυτό και ότι παρά όλα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη χρονική πίεση. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να προσκαλέσω τον συνάδελφο Χένκελ που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια, να αναλάβει το επόμενο πάνελ για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. All over Europe, people are getting ready to vote in the European elections in May. Whoever you are, wherever you are, you can get involved and make sure everyone makes their voice heard. There is a movement of involved citizens, a diverse community of people who want to shape the Europe of tomorrow.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 because we want everyone to say, this time I'm voting. Hello. Good afternoon, ladies and... Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ας περάσουμε στο τελευταίο πάνελ για απόψε, το οποίο φέρει τον τίτλο μια υφόρος και βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα μειώσει την πίεση στους ωκεανού. Θα ήθελα καταρχά να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Μάισνερ για την όλη οργάνωση. Όπως είπε και ο κύριος Χέρτσικ από το ε, Γκέομαρ, ε, τόσο εύγλωτα, ε, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τους ωκεανούς μας σε καλή κατάσταση. Και πρώτη, ναι, αυτή τη φανταστική ιδέα ε, να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ωκεανών. Ξέρετε ότι ξέρουμε περισσότερα για την επιφάνεια της Ελληνής από ότι για το βυθό των ωκεανών και θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Θυμίζω ότι το τελευταίο αυτό πάνελ θα εστιάσει κυρίως ε, στο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην γαλάζια οικονομία, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση που υφίστανται οι ωκεανοί. Όπως είπε ο κύριος Χέρτσικ, το 50% των τροφοίμων μας, της ενέργειας που καταλαμβάνουμε και ε, των φυσικών πόρων του μέλλοντος θα πρέπει να παράγονται από τους ωκεανούς. Θα ήθελα να προσθέσω όμως ότι υπάρχουν πολλές χώρες που βρέχονται από ωκεανούς που έχουν τεράστια ποσοστά ανεργίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για τους Ευρωπαίους και την πολιτική του την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, να εξασφαλίσουν ότι ε, θα υπάρχει μια συνοχή στην πολιτική ε, παντού, σε όλους τους κλάδους γαλάζιας οικονομίας. Τώρα βέβαια πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά και θα ευθυγραμμιστούν με τρόπο επιτυχία. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Ε, ε, μειώνονται μεν οι ρυθμιστικοί φραγμοί και τα εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα ε, δίνεται και μεγάλη χρηματοδότηση και είμαι σίγουρος ότι τα ανέφερε προηγουμένως αυτά ο Επίτροπος Μοέδας. Και αυτή η χρηματοδότηση κυρίως θα προέρχεται από τα ερευνητικά προγράμματα και τα διαρθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία και τη Θαλάσσια Πολιτική. Ε, ο παράκτιος, ο αλευτικός τουρισμός, οι δατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, οι θαλάσσιες βιοτεχνολογίες, ε, η εξόριξη του βυθού Όλα αυτά είναι τομεί που θίγονται από τις διάφορες πολιτικές και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Και σε τούτο εδώ το πάνελ θα ασχοληθούμε με διάφορα από αυτά τα θέματα. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω και μια ανησυχία που έχω. Γνωρίζετε όλοι ότι η Βρετανία επί δεκαετίες ήταν θαλασσοκράτηρα. Ε, και μάλιστα ε, πολλοί ε, θεωρούσαν ότι δάμαζαν τη θάλασσα. Και η νομοθεσία που έχουμε για την ωκεανογραφία και πολλά ε, από όσα αφορούν τα σημερινά ζητήματα έχουν έμπνευση βρετανική. Καλωσορίζω την κυρία ε, Έμα Ναβάρο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της λέγω το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαι εδώ με όλους σας. Να συγχαρώ καταρχάς και να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την συζήτηση για το μέλλον των ωκεανών που τόσο πολύ τη χρειαζόμαστε. Ένα μέλλον που όπως μας θύμισαν και οι προηγούμενοι μιλητές αφορά τη ζωή όλων μας εδώ στον πλανήτη τους εξαρτάται. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προστατεύσουμε και θα χρησιμοποιούμε ή θα εκμεταλλευόμαστε με τρόπο βιώσιμο του ωκεανού μα. Ακούσαμε σήμερα ότι οι ωκεανοί συμβάλλουν τα μάλα στην παγκόσμια οικονομία και είναι ε, και ε, μια δύναμη που παράγει και θέσεις εργασία και καινοτομία και δίνουν οικονομικέ ευκαιρίε για το μέλλον. Ξέρουμε ότι πέραν των οικονομικών νόμος ωφελών, οι ωκεανοί είναι καθοριστική σημασία και για κρίσιμα θέματα του πλανήτη, από την ε, επιστηστική ασφάλεια, την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Όμως για να ε, εκμεταλλευτούμε το πλήρες δυναμικό των ωκεανών μας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία τους πρέπει την υγεία τους να την κοιτάξουμε γιατί κινδυνεύει πολύ. Η εικόνα είναι ζωφερή και πραγματικά ε, πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου τώρα, αμέσως. Χρειάζεται μια υπεύθυνη και βιώσιμη προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη των ωκεανών, για να βεβαιωθούμε ότι ο μεγαλύτερος φυσικός πόρος του πλανήτη παραμένει ζωντανός και από αυτόν μπορούν να ωφεληθούν και να αποφεληθούν οι ερχόμενες γενιές μια βιώσιμη γαλάζια ατζέντα είναι απαραίτητη. Τα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προωθήσουν αυτή την ατζέντα είναι ευπρόσδεκτα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το να προωθήσουμε μια τέτοια γαλάζια οικονομία που να είναι βιώσιμη, είναι προτεραιότητα. Είναι λογικό και αυτονόητο, διότι εφόσον υποστηρίξουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, και αυτά είναι στον πυρήνα τη δράση μα, έρχεται μαζί και η γαλάζια οικονομία. Ε, Ω μπούσουλα έχουμε ακολουθήσει φιλόδοξου κλιματικού στόχου. Ε, τουλάχιστον 25% των ε, κομμελίων μα, ε, τη χρηματοδότησή μα Επίσης, έχει να κάνει με την κλιματική δράση. Πέρσι έφτασε τα 16 δις ευρώ. Επίσης, θέλουμε να προσφέρουμε 100 δις δολάρια για κλιματικά προγράμματα παγκοσμίω και ε, θέλουμε να έχουμε εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη διάρκεια του χρόνου είμαστε ένα κέρια σημασία επενδυτή για την οικονομία των ωκεανών, κινητοποιώντα το κεφάλαιο του ιδιωτικού τομέα προ τους βιώσιμους στόχους και την επιδίωξή τους και στην Ευρώπη και εκτός. Ένα καλό παράδειγμα είναι το πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη των ε, γαλάζιων ακτών στην Ευρώπη. Έχουμε αναπτύξει πολλές δυνατότητες με επενδύσεις άνω των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια και θα συνεχίσουμε να ε, στηρίζουμε αυτόν τον τομέα ανάπτυξη. Επίσης η προστασία των ακτών αυτών έχει να κάνει και με το πρασίνισμα του τομέα της ναυτιλίας που είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα. Εργαζόμαστε για την προστασία των ωκεανών από την ρήπανση από τα πλαστικά έναν από τους μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα οικοσυστήματα πλέον. Γι' αυτό πέρσι μαζί με τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες επενδύσεων εγκαινιάσαμε την πρωτοβουλία για τους καθαρούς ωκεανούς. Τα ερχόμενα πέντε χρόνια θα προσφέρουμε 2 δις ευρώ για προγράμματα που θα αντιμετωπίσουν την αποκομιδή απορριμμάτων στους ωκεανούς, δηλαδή τα αστικά λίματα που δεν έχουν τύχη επεξεργασία και τα πλαστικά. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα σοβαρά που έχει τεράστια κοινωνική εμβέλεια. Ε, όμως η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας δεν έχει να κάνει μόνο με λεφτά και χρήμα, έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της καινοτομία και την άρση των φραγμών για νέα προγράμματα. Η γαλάζια οικονομία και τα προγράμματά τη ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση στα ιδιωτικά κεφάλαια διότι πολλές φορές έχουν να κάνουν με τεχνολογικές λύσεις που είναι τελείω καινοτόμε ή με άγνωστες αγορές. Γι' αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέψαμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των προγραμμάτων και να προσελκύσουμε ιδιωτικού επενδυτές. Αυτό είναι καθοριστική σημασία γιατί η καινοτομία και η επιστήμη είναι κρίσιμη σημασία για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της βιωσιμότητα. που ε, έχουν να κάνουν με την ε, περαιτέρω ανάπτυξη και την προστασία των ωκεανών. Όμω για να ανθίσει η γαλάζια οικονομία πρέπει να εντείνουμε την ε, χρηματοδότηση. Οι ανάγκε χρηματοδότηση είναι προφανώ πέραν των κρατικών συλλογισμών. Θα πρέπει ο ιδιωτικό τομέα να ανασκουμποθεί και να έρθει να συμμετάσχει. Θα πρέπει η δική του συμβολή να ληφθούν υπόψη στι ανάλογε αποφάσει μα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τι βιώσιμε επενδύσει για του ωκεανού μα για να καθοδηγήσουμε τους επενδυτές προς τη βιωσιμότητα και την βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές της. Ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την βιώσιμη χρηματοδότηση των ωκεανών που αναπτύξαμε από κοινό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το το ΒΒΕΦ και την, το Ίδρυμα για τους βιώσιμους πόρους είναι μια αρχή. Φέτος οι αρχές αυτές θα βρεθούν στην καρδιά μιας νέας πρωτοβουλίας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Περιβάλλοντος του ΙΕ. Αυτό ξεκίνησε ε, ως μια πρωτοβουλία 12 θεσμών και τώρα γίνεται ο κατεξοχήν κανόνας για την ε, επένδυση στους καθαρούς ωκεανούς με τρόπο βιώσιμο. Όμως ο χρόνος περνάει και έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Προκλήσεις που θα απαιτήσουν δράση ε, συνδυασμένη και πολυμερή, αλλά και ατομικέ πρωτοβουλίες όλων μας. Υπ' αυτήν την έννοια, η σημερινή εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για να να προβάλλουμε ιδέε και να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε ευθύνη για την εξέβρεση λύσεων για αυτές τις προκλήσεις. Σας διαβεβαιώ ότι η ΕΤΕ παραμένει πλήρω δεσμευμένη στον αγώνα της προώθησης της γαλάζιας οικονομίας που θα κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και για την σύναψη εταιρικών σχέσεων με άλλους προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ναβάρο. Και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Πιέρ Ντελσό, τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις να πάρει το λόγο. Για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ μεγάλος τίτλος για μια γενική διεύθυνση. Θα συνοψίσω με λίγα λόγια αυτά που θέλω να πω το Sky, το Copernicus, ε, ε, και η Αρκτική. Ο είναι ένας, ένα όριο, αλλά αποτελεί ε, και ένα εργαλείο για να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει στη γη. Και το είπε και ο πρόεδρος Σταγιάννη, ότι μαζί με το Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσω του Κοπέρνικου τι συμβαίνει στη Γη. Το Κοπέρνικος είναι ένα σύστημα δορυφόρων που βασικά παρακολουθεί τον πλανήτη και παίρνει φωτογραφίες και μας δίνει φωτογραφίες για τις διάφορες καταστάσεις του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, φυσικά, οι ωκεανοί είναι πολύ σημαντικό μέρος της παρατήρησης που υλοποιούμε με το Κοπέρνικος και θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το Κοπέρνικους ε, αξιολογείται από όλου, ακόμη και από τη ΣΥΠΑ, ως το καλύτερο σύστημα παγκοσμίω. Έτσι λοιπόν, ε, ως Ευρωπαίοι μπορέσαμε να ε, συνάψουμε ένα σύστημα, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που είναι το καλύτερο για την παρατήρηση της γης. Τι κάνουμε τώρα με τις εικόνες που παίρνουμε από το Κοπέρνικους, αναπτύσσουμε υπηρεσίες που παρακολουθούν επίσης τι συμβαίνει στους ωκεανούς. Έτσι λοιπόν έχουμε αναπτύξει την θαλάσσια υπηρεσία που μας δίνει κάποιες προβλέψεις για τους ωκεανούς και πληροφορίες για το κλίμα στους ωκεανούς. Και επίσης ε, μέσω των δορυφόρων μπορούμε να έχουμε μία έκθεση σε θέματα που αφορούν ε, την ε, αύξηση του επίπεδου των υδάτων στη θάλασσα ή το λιώσιμο των πάγων. Μία άλλη πολύ σημαντική πτυχή και συνιστόσα του Κοπέρνικου είναι η παρατήρηση ε, στη θάλασσα. Χρησιμοποιείται για να παρακολουθούμε όλες τις δραστηριότητε του ωκεανού, παραδείγματο χάρη τα σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα που βρίσκονται και τι κάνουν. Αλλά και κάτι πολύ σημαντικό να ανοιχνεύουμε τη ρήπανση και να μπορούμε να αντιδράμε γρήγορα. Μία άλλη πολύ σημαντική, σημαντική υπηρεσία είναι η υπηρεσία εκτακτη αναγκη ε, Χρησιμοποιείται όταν έχουμε μία κατάσταση κριση πρέπει χάρη στη Μεζανβίκη όταν έχουμε πλημμύρε, παρακολουθεί την κατάσταση του Κοπέρνικους και μπορούμε να, μπορεί να μα βοηθήσει για να βοηθήσουμε και να σώσουμε του ανθρώπου επί τόπου. Χρησιμοποιείται δυστυχώ σε τακτική βάση και θέλω να αναφέρω τον Δίας. Το Κοπέρνικους είναι ο μεγαλύτερος πάροχος δεδομένων στον κόσμο. Έτσι λοιπόν όλες ε, οι εικόνες, φωτογραφίες ε, που παίρνουμε μέσω του Κοπέρνικους είναι δωρεάν για όλους. Αλλά η δυσκολία είναι ότι επειδή υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα και ακόμη και αν είναι δωρεάν, είναι δύσκολη η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων. Τι κάναμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσαμε να πληρώσουμε ιδιωτικούς ε, παραγωγούς και να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες με όλα αυτά τα δεδομένα. Ε, και ε, όλα τα δεδομένα διατίθεται δωρεάν σε όλους. Έτσι λοιπόν και είναι η ιδέα. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν αυτά τα δεδομένα και να αναπτύξουν υπηρεσίες και λύσεις, προϊόντα βάσει αυτών των εικόνων. Έτσι λοιπόν, αν ε, δεν ξέρεις πια τι να κάνεις, ε, Κυριακή βράδυ βρέχει στις Βρυξέλλες, ε, πας στον Τάιας, είναι δωρεάν και δημιουργείς κάτι, μπορείς να παρακολουθήσεις τι συμβαίνει στον ωκεανό. Το παρουσιάζω ως αστείο, αλλά αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι βασικά να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα από όλου και στην Ευρώπη βέβαια και ότι αναπτύσσουμε υπηρεσίες που μας βοηθούν να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και στους ωκεανούς. Και τέλο ε, Αρκτική. Γιατί αναφέρω την Αρκτική. Γιατί ακόμη η ΕΝ και το Κοπέρνικους είναι ένα πολύ επιτυχές πρόγραμμα. Πρέπει να το συνεχίσουμε, να το αναπτύξουμε και να το συντηρήσουμε στο μέλλον. Και τώρα, ε, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ένα νέο διαστημικό πρόγραμμα για το μέλλον. Και ένα από τα στοιχεία που θέλουμε να αναπτύξουμε στο Κοπέρνικου, αν έχουμε υποστήριξη φυσικά από τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, είναι η λεγόμενη Αρκτική Αποστολή. Τι θέλουμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε το Κοπέρνικου για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση στην Αρκτική. Γιατί ξέρουμε ότι η κατάσταση στην ε, Αρκτική επηρεάζει πάρα πολύ το κλίμα παγκοσμίω, ε, αλλά και στου ωκεανού. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιε αποστολέ. Θέλουμε να τι αναπτύξουμε χρησιμοποιώντα του δορυφόρου. Και επίσης ε, θέλουμε να αναπτύξουμε μια αποστολή για την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να παρακολουθούμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Και πάλι αν θες να το κάνεις, το καλύτερο εργαλείο διαθέσιμο είναι το διάστημα. Έτσι λοιπόν, κάποιε φορέ παραπονιόμαστε ότι δεν είναι σε ηγετική θέση Ευρώπη σε πολλού τομεί, αλλά μπορώ να σα πω ότι με το Κοπέρνικο έχουμε ένα εργαλείο ιδιαίτερα ισχυρό. Είναι εξαιρετικό και επίσης θα είναι ένα ισχυρό μέσο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στους ωκεανούς. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Δερζού. Σε μία πρόταση, όταν μιλάτε για τον Κοπέρνικο, έχουμε την εντύπωση ότι έχει επιτευχθεί αυτό που πρότεινε ο κύριος Χέρτσικ. Τι λέτε για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλασσών και Οκεανών. Μα έχουμε ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος που τον ανέφερα. Γιατί να μην κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τους ωκεανούς. We uh, this and maybe we can <laughs> this Ωραία, το σημειώνουμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ότι δεσμεύεται ένας ε, υψηλός αξιωματούχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε κάποιους συναδέλφους μας, η κυρία Ισάσκου Πιλπάου Μπαραντίκα από την Άλτε, για τρία λεπτά. Η κυρία Πιλπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας σε όλες και όλους. Καλησπέρα και ευχαριστώ ε, τους επισκέπτες, αλλά και εκείνους που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση όπως η Γκέινέ Μάισνερ που είναι τόσο ερωτευμένη όπως πάντα με τους ωκεανούς. Η στρατηγική αυτή η γαλάζια που αναλύουμε σήμερα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες χειροπιαστές δράσεις του μοντέλου 2020. Από την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 σήμανε σημαντική και οριστική αλλαγή της σχέσης μας με τη θάλασσα. Μια μετατροπή των παραδοσιακών ε, δραστηριοτήτων, διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος, δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, και εκμετάλλευση της ενέργειας στη θάλασσα. Όλα αυτά βασίζονται στην βιωσιμότητα. Αναπτύσσουμε ε, την οικονομία μας μειώνοντας την πίεση στη θάλασσα. Και αυτό είναι προς όφελος των παράκτιων ε, κοινοτήτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε, ε, να παρακολουθούμε και να οργανώνουμε την προσπάθειά μας. Ε, οι παραδοσιακές δραστηριότητες τώρα βασίζονται ε, σε πολύ αυστηρές εκθέσεις ε, για τα αποθέματα. Έχουν βελτιωθεί τα αλευτικά εργαλεία και οι τεχνικές. Αναπτύσσεται η υδατοκαλλιέργεια και μετατρέπονται οι στόλοι και ο αλευτικός και ο Ξεφεύγουμε από το διοξίδιο του άνθρακα. Προχωρούμε στην αυτόνομη πλοήγηση. Έχουμε ευκαιρίε για τα ναυπηγεία που είναι παραδοσιακή δραστηριότητα. Η γνώση επίσης οδηγεί και σε καινοτομία και σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες ε, και μπορούμε να μετατρέψουμε τις απειλέ, όπως είναι η ρήπανση από τα πλαστικά σε ευκαιρίε και στη στεριά με νέε δραστηριότητε και προϊόντα ε, για υποκατάσταση αυτών των ρηπαντών και άλλες ε, δραστηριότητες στη θάλασσα με τεχνικές καθαρισμού και συλλογής που ήδη δίνουν καρπούς. αιφόρος εκμετάλλευση λοιπόν ε, ενός μεγάλου θαλάσσιου πόρου που είναι η ενέργεια. Εγώ ως Βάσχα είμαι πολύ περήφανη που η μικρή μας χώρα είναι πρωτοπόρα στην έρευνα για την ενέργεια από τις παλήριες. Στο Μουτρίκου καταφέραμε να ε, παράξουμε 1,3 γιγαβάτ ε, ώρες ε, το 2016, συνδεδεμένα στο δίκτυο. Αυτό μπορεί να είναι χαμηλή παραγωγή, αλλά κανένα άλλο εργοστάσιο που χρησιμοποιεί την ενέργεια από τις παλήριες δεν το έχει καταφέρει. Χρησιμοποιεί και δοκιμάζει νέα μοντέλα μηχανών ε, έτσι ώστε ε, να ε, εκμεταλλευτεί αυτή την ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τις Κανάρια, την Κανάρια νησιά με την αιωλική ενέργεια. Άλλο κλειδί για τη στρατηγική μας είναι η οργάνωση των νέων δραστηριοτήτων. Έτσι μειώνονται συγκρούσεις και δημιουργούνται συνέργειες με την ευφυή εξειδίκευση ή την εγκύτητα. Και τέλος η παρακολούθηση και επιτήρηση ε, κλείνει αυτό το κύκλο για να ε, μπορούμε να ελέγχουμε αυτές τις πρακτικές και τις αποκλίνουσες πρακτικές από αυτό το αηφόρο και βιώσιμο μοντέλο στις νέες πολιτικές μας. Γι' αυτό χαιρετίζω αυτή τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου, έτσι ώστε να εδρεωθεί αυτή η σημαντική εξέλιξη της σχέσης μας με τη θάλασσα. Και το λέω ως Ευρωβουλευτής, αλλά και ως μέλος μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας που έζησε, ζει και φιλοδοξεί να συνεχεί να ζει από τη γαλάζια οικονομία και που έχει ζήσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αηφορία και βιωσιμότητα. Γι' αυτό σας φέρνω ένα μήνυμα από την ακτή. Σε όλη αυτή την προσπάθεια μετασχηματισμού, αυτέ οι τοπικέ κοινωνίε, οι παρακτηε θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν. Η συμμετοχή του είναι εκ των όνου κάνευ, έτσι ώστε αυτή η αλλαγή να προοδεύσει και να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε αιώνες γνώσεων και συμβίωσης με τη θάλασσα. Και αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να αποδίδουν στα μέλη τους ευκαιρίες, υπηρεσίες και αναγνώριση για την προσπάθεια που κάνουν έτσι ώστε να πρωταγωνιστούν σε αυτή τη βελτιωμένη σχέση με τη θάλασσα. Ελμαρ, που είναι η θάλασσα στα ισπανικά, αλλά Λαμάρ στο θηλυκό τη λένε οι άνθρωποι της θάλασσας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνάδελφος είναι η Κλάρια Ουτζίνα Αγγιλέρα Γκαρσία από τους Σοσιαλιστές και δημοκράτε για τρία λεπτά. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μια καλή συζήτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα το απόγευμα. Σε αυτό το πάνελ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σκέψεις για να δώσω ενάφησματα στη συζήτηση. Η γαλάζια οικονομία δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο μια απλή έννοια ακόμη. Όταν πριν χρόνια αρχίσαμε να μιλάμε για τη βιωσιμότητα, όλα ήταν βιώσιμα. Αυτό που συνεισέφερε στη βιωσιμότητα και αυτό που δεν συνεισέφερε, αλλά όλα έφεραν την ετικέτα βιωσιμότητα. Προσοχή. Ο κίνδυνο της γαλάσιας οικονομίας είναι να γίνει μια έννοια που να καλύπτει τα πάντα. Όλα τα κάθε τι καινούριο. Κάθε τι καινούριο πρέπει να είναι διαφορετικό. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε πάντα. Θα πρέπει να δρούμε και με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την οπτική για στην πράξη. Και σε σχέση και με τον κυρία Ναβάρο, θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με την οποία χειριζόμαστε τις επενδύσεις μας, ε, ιδιωτικές και δημόσιες, για να ευνοήσουμε και να προωθήσουμε αυτή τη γαλάζια οικονομία. Αυτό είναι σαφές. Μπορούμε να έχουμε τους ίδιους στόχους ή παρόμοιους στόχους, αλλά θα πρέπει να πράττουμε με διαφορετικό τρόπο και να έχουμε ξεκάθαρα πού κατευθύνουμε τις επενδύσεις μας, ιδιαίτερα τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές. Οι ωκεανοί περιλαμβάνουν τεράστιο πλούτο σε πόρους και έχουν μια τεράστια δυναμική για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνία και την απασχόληση. Αν και είναι τεράστιο το δυναμικό τους, υπόκειται σε υπερβολικές πιέσεις υπερβολική εκμετάλλευση των πόρων τους, ρήπανση, αυξανόμενη βιοπικιλότητα και κλιματική αλλαγή. Όλο αυτό, όλο αυτό το μεγάλο δυναμικό μπορεί να καταλήξει διαφορετικά. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους δράσης. Εγώ νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που θέλω να αναφερθώ, πολλοί απόψε αναφέρθηκαν και στα πλαστικά και στη ρήπανση των ωκεανών. Εγώ θέλω να μιλήσω για την ελευτική δραστηριότητα. Η τομεακή πολιτική της Ελίας, της, ε, η κοινοτική πολιτική, έφερε μεγάλες αλλαγές. Ίσως να μην ε, το αξιολογούμε επαρκώς. Γιατί μένουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όμως έχουμε εγκρίνει σχέδια διαχείρισης ε, των ελευτικών πόρων ε, στα πλαίσια της κοινή ελευτικής πολιτικής και ε, για τη Δυτική Μεσόγειο αλλά και στον Ατλαντικό, στα Δυτικά ύδατα όπως και στη Βαλτική ή στη Βόρεια Θάλασσα. Απομένουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά γίνονται ήδη πράγματα για καλύτερη εκμετάλλευση και κατάργηση της υπερελίας. Και επίσης υπάρχουν μεγάλες θυσίες που γίνονται από όλους τους κλάδους. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες αρχές ε, που θα ήθελα να καταθέσω εδώ στη συζήτηση. Κάποιες αρχές ε, που είναι απαραίτητες ε, για αυτή την βιώσιμη γαλαζία οικονομία. Καταρχήν, για να την υλοποιήσουμε τη γαλαζία οικονομία θα πρέπει να έχουμε τη συμμετοχή και τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών στους ωκεανούς. Όλων. Κανένας δεν πρέπει να αποκλείεται. Θα πρέπει να δεσμευτούμε και να εμπλέξουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων για τη βιώσιμη γαλαζική οικονομία. Δεύτερον, να έχουμε κατά νου κάτι που χρησιμοποιούμε πολύ, αλλά ενίοτε με αντιφατικό τρόπο. Την ε, υποστήριξη, τη στήριξη της καλύτερης δυνατής παροχής συμβουλών. Δηλαδή, να αξιολογούμε με τον κατάλληλο τρόπο την αξία των επιστημονικών αναλύσεων. Γιατί πολλές ε, φορές ε, αν ε, δεν μας κάνει για την υιοθέτηση μιας θέσης, την απορρίπτουμε. Και το βλέπουμε εδώ και στο Κοινοβούλιο. Η επιστημονική αξία των κομματήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εφαρμογή της γαλάζιας οικονομίας. Και τρίτον, θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλες τις στοιχείες της βιωσιμότητας οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πτυχή. Και τις τρεις. Αν ξεχάσουμε μία εξ αυτών, τότε δεν θα τα κάνουμε καλά τα πράγματα. Και τα τρία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη ενός καλύτερου μέλλοντος σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική πτυχή, την κοινωνική και την, και την οικονομική. Με συγχωρείτε. Κανένα δεν θα πρέπει να μείνει εκτός. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι η γαλάζια οικονομία προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε πού θα την κατευθύνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις που θα ήθελα να σας καταθέσω εδώ σήμερα. Βλέπουμε πολύ μεγάλες αλλαγές και δεν ε, θα ήθελα να ε, ξεχάσουμε την πρόταση να υπάρχει μια νέα υπηρεσία για τους ωκεανούς. Εμένα πολύ καλή μου φαίνεται, αλλά ξέρετε τι σκέφτεται το Συμβούλιο. Λιγότεροι πόροι για όλες τις πολιτικές για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να δούμε πώς θα κάνουμε περισσότερα, πώς θα έχουμε περισσότερα εργαλεία και μέσα με λιγότερους πόρους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει τους πόρους που έχουμε να τους χρησιμοποιήσουμε και να τους κατευθύνουμε καλύτερα. Δεν μας διευκολύνουν βέβαια τη ζωή, αλλά νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Now I would like to... Ευχαριστώ. Και θα ζητήσω τώρα την κυρία Τομά από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες να παρέμβει για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Θα ήθελα να πω αν ήμουν ωκεανό σήμερα το απόγευμα και έβλεπα τόσοι πολλοί να σκύβουν πάνω από το λίκνο μου θα ανησυχούσα. Τόσες επενδύσεις και θα έλεγα πω πω λιγάκι μαζευτείτε. Είναι σαν να παρουσιάζεται ένα νέο Ελντοράντο για πολλούς επενδυτές. Και υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι. Καλοί λόγοι υπόθηκαν, δεν θα τους επαναλάβω το δυναμικό για την ανανεώσιμη ενέργεια από τη θάλασσα, το δυναμικό για τη ρομποτική που επιτρέπει να πάμε και να αντλήσουμε σε εκατοντάδες χιλιόμετρα κάτω από τη στάθμη. Ξέρετε ότι το σκάφος που είναι το πιο ε, γνωστό στο στόλο μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό που πηγαίνει να κάνει εξορίξεις ε, στη θάλασσα ε, για πετρέλαιο σε μεγάλα βάθη. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και εδώ υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να φαίνεται τόσο ελκυστική η γαλάζια οικονομία. Καλή και κάποιοι λιγότερο καλή. Έχουμε ένα πληθυσμό που αυξάνεται. Έχουμε έλλειψη φυσικών πόρων στη γη, στην ξηρά. Έχουμε οικονομική παγκοσμιοποίηση που εντείνεται και θα συνεχίσει να εντείνεται. Έχουμε μεταφορές εμπορευμάτων και όπως είπα έχουμε και τεχνολογικά μέσα που επιτρέπουν φοβερά κατορθώματα σε σχέση με κάποια χρόνια. Αυτά είναι τα θετικά. Όμως κατά τη δική μου αντίληψη εδώ προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες επιτακτικές ανάγκες. Πρώτα απ' όλα να μην ξανακάνουμε στη θάλασσα αυτό που κάναμε στην ξηρά στη γη. Επίσης για αυτό το λόγο να αλλάξουμε ε, μοντέλο εκμετάλλευση θα έπρεπε να ξεχάσουμε τελείω τον όρο μοντέλο εκμετάλλευση. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο όρο. Και γιατί. Γιατί στην γη, στην ξηρά, τι κάναμε. Κατασπαταλήσαμε, διαπράξαμε σφάλματα που δεν διορθώνονται, οικοκτονίες θα τις έλεγα, οικολογικές οικοκτονίες, εγκλήματα κάτω του περιβάλλοντος, κατασπατάληση, κατασπατάληση φυσικών πόρων που δεν μπορούν να ανανεωθούν. Πρέπει να αλλάξουμε εντελώ λοιπόν μοντέλο, πρότυπο. Και εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που προηγουμένω η Κλάρα Αγγιλέρα. Στην Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε στην Αλία και την μέγιστη απόδοση, ακόμη και αν δεν είναι η καλύτερη, ακόμη και αν βελτιώνεται. Ε, πρέπει να το πιστέψουμε παρόλα αυτά, ε, γιατί θα πρέπει από του φυσικού πόρου να παίρνουμε αυτό που μπορεί να, να παραχθεί. Δεν μπορούμε να επιτιθέμεθα στο κεφάλαιο των φυσικών πόρων και να παίρνουμε ό,τι μα ενδιαφέρει ε, και να μην ε, τραβάμε για να, όπως από ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση των ε, καπιταλιστών. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τις λαπερέ συνέπειες για τα αποθέματα και τους φυσικούς πόρους εν γέννη. Χρειάζονται πολλά εδώ, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είναι δύο οι βασικές απαιτήσει. Πρώτα απ' όλα, να κοιτάξουμε την καλή διαχείριση των πόρων και των οικοσυστημάτων. Διότι δεν είναι δεδομένα αυτά, και εδώ θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές, και ναι, το θέμα των ελέγχων, το θέμα της αστυνόμευσης. Πρέπει να κοιτάμε ποιο κάνει τι. Συχνά δεν αρκεί η εμπιστοσύνη, δεν γεννάει έλεγχο ω προ την παραγωγή και την παραγωγή πλούτου, καθώ και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ο έλεγχο είναι ε, κέρια σημασία. Για να ολοκληρώσω, να πω <clears throat> για να είμαστε αποτελεσματικοί και σοβαροί και να φτάσουμε στο τέρμα ε, των όσων λέμε, των υποχρεώσεων του δρόμου μας, θα πρέπει να βγούμε από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και την λογική των, οικονομικ... εθνικών εγωισμών. Θα πρέπει να αφήσουμε τα 10 και τα 12 μίλια και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι υπήρξε χερσόνησος, κατακαιρματισμένο ήπειρος και μια από τις πιο θαλάσσιες, τις ναυτικές ήπειρους. Μας περιβάλλει νερό δεν είναι και λίγο αυτό για τα θεσμικά μας όργανα, κύριε Επίτροπε. Έχουμε μια γενική διεύθυνση που ασχολείται υποτίθεται μόνο με την Αλία, τη Μάρε. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε μια επιτροπή, την Επιτροπή Αλίας, που υποτίθεται ότι ασχολείται με την Αλία. Αλλά έχουμε και τι θαλάσσιε μεταφορέ την Επιτροπή Μεταφορών, λόγο. Δεν θα σας τα πω όσα υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουμε συνέστηση, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι η Ευρώπη είναι θαλάσσια και ναυτική. Τι θα γίνει λοιπόν με τη θαλάσσια κυβέρνηση, το είπα και για να ολοκληρώσω πρόεδρε, δυο λόγια για την ανθρωπότητα. Να μην ξεχνάμε την ανθρωπότητα στους ωκεανούς και να μην ξεχνάμε κατά κύριο λόγο το δικαίωμα, μάλλον την υποχρέωση, το καθήκον της διάσωσης στη θάλασσα. Η διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι αρχή, αξία που ισχύει από αιώνες απαράβατη και τώρα την εγκαταλείπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. And now uh, we have a couple of speakers. Uh, each one uh, I would like to ask to really stick to the... Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρείτε το πεντάλεπτό σας. Ο κύριος Βίτο Βερτέλιο από την Ένωση ατυπιομάζας στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για τρία θέματα. Πρώτον, να σας εξηγήσω ε, τι είναι τα φύκια. Ποιο είναι το πρόβλημα ε, στην υγεία των ωκεανών και τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα φύκια για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Τι είναι η βιομάζα από τα φύκη. Είναι μικροφύκη, πολύ μικροσκοπικά, που καλύπτουν όλους τους ωκεανούς ε, και ε, με τη φωτοσύνθεση τους ε, παράγουν οξυγόνο όπως ακούσαμε. Αυτή τη μορφή έχουν. Είναι το ένα χιλιοστό του ενός χιλιοστού. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίε και είδη με διάφορα ονόματα. Αυτά είναι από τα πιο διοδομένα μικροφύκη στον πλανήτη ε, καλύπτει το 5% της φωτοσύνθεσης των ωκεανών. Και ποια είναι τα πολύ μικροσκοπικά φύκη. Είναι αυτά τα φύκη που βλέπετε εδώ, στις ακτές επίσης. Ε, ε, σας δείχνω μερικές φωτογραφίες. Αυθονούν στην Ευρώπη. Στην Ασία καλλιεργούν αυτά τα φύκια. Στην Ευρώπη τα συλλέγουν από τους ωκεανούς, τις οδιές. Ε, έχουν διαφορετικές δραστηριότητες ε, και ε, ιδιότητες τα διάφορα φύκια. Μπορούν να παράγουν πολλοί σακχαρίτες, μπορούν να επεξεργάζονται σε βιολογικό καθαρισμό ε, τα αλήματα. Ε, αυτό το φίκι που σας δείχνω τώρα, το κόκκινο, αυθονούσε στην Πορτογαλία, στη χώρα μου, αλλά ε, υπερεκμεταλλεύτηκαν αυτό το είδος οι άνθρωποι και τώρα σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Να σας πω δύο λόγια και για το πρόβλημα ποιο είναι. Της υγείας των ωκεανών ουσιαστικά από την μη βιώσιμη εκμετάλλευση των ωκεανών. Εδώ βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια ότι δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η ρήπανση και το δεύτερο είναι η υπεραλίευση. Η ρήπανση έχει πολλές εκφάνσεις και πτυχές. Ε, έχει υπερβολική έκκληση διοξιδίου του άνθρακα ε, στην ατμόσφαιρα, αλλάζει το κλίμα και αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα στους ωκεανούς. Άλλο πρόβλημα είναι τα πλαστικά που αναφέρθηκαν για τη ρήπανση και η υπεραλίευση έχει σχέση με αυτά. Το θέμα των πλαστικών κατά την προσωπική μου άποψη είναι από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Όχι τα μεγάλα πλαστικά αλλά τα πολύ μικροσκοπικά πλαστικά γιατί αυτά τα πλαστικά δεν προέρχονται μόνο από την αποσύνθεση των ίδιων των πλαστικών από τη διάσπαση αλλά και από ε, την πλήση όλων των ρούχων που χρησιμοποιούμε και εγώ τα χρησιμοποιώ που δεν είναι όλα βαμβακερά αλλά είναι συνθετικά. Κάθε φορά που πλένουμε ένα ρούχο συνθετικό, δηλαδή πλαστικό, απελευθερώνονται σωματίδια μικροσκοπικά πλαστικών και καταλήγουν στον ωκεανό. 6 με 9 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Εκατομμύρια τόνοι. Αυτό είναι τεράστιο ε, ποσό. Και αυτά τα μικροπλαστικά για να διασπαστούν χρειάζονται χίλια χρόνια και δεν μπορούν να απομακρυνθούν με κανένα τρόπο από τους ωκεανούς. Είναι τόσο μικροσκοπικά, ε, ε, αυθονούν, είναι ε, παντού και τα τρώνε τα αμαλάκια, οι πολύ μικρές γαρίδες, τα ψάρια και περνάνε στην τροφική αλυσίδα και τελικά καταλήγουν και στον άνθρωπο. Αλλά α είμαστε λίγο πιο θετικοί και αισιόδοξοι. Πώς μπορούν να συνεισφέρουν τα φύκη λοιπόν. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα στον ωκεανό. Το ένα είναι τι βάζουμε, τι ρίχνουμε δηλαδή, τι πετάμε στους ωκεανούς και το άλλο είναι τι βγάζουμε από τους ωκεανούς. Τι ρίχνουμε εκεί. Ένα σωρό ε, χημικούς ε, και τι βγάζουμε με την υπεραλίευση ψάρια, αλλά και, θηλαστικά, δελφίνια, ε, φάλαινες ε, και ε, μα, μαλάκια και οστρακοειδή, πολύ μικρές γαρίδες, ακόμα και στην Αρκτική. Σε τρία επίπεδα είναι η δράση μας. Το πρώτο είναι η πρόληψη. Το σημαντικότερο είναι να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Όχι απλώς να καθαρίσουμε τους ωκεανούς, με την πρόληψη να τα σταματήσουμε όλα αυτά και να έχουμε μια οικονομία πιο κυκλική, χωρίς πλαστικά, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα και ε, μια δεσμευτική βιωσιμότητα και ε, πολύ δρακόντια φορολογία για οτιδήποτε ρηπαίνει τους ωκεανούς. Μετά, ενημέρωση. Κατά την άποψή μου είναι το σημαντικότερο. Οι πολίτες, αν δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει, δεν πρόκειται να πιέσουν τους πολιτικούς και οι πολιτικοί θα δρανήσουν. Και τέλος, χρειάζεται να έχουμε ισόρροπη εκμετάλλευση των θαλασσών και των ωκεανών. Ε, με την υπερεκμετάλλευση δεν προστατεύεται ο ωκεανός. Τι μπορούν λοιπόν τα φύγη να κάνουν για όλα αυτά τα πράγματα. Τέσσερα κυρίως. Τα δύο πρώτα είναι ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τις ε, ηχθειοτροφές, στις ηχθειοκαλλιέργειες. Στην ιδιατοκαλλιέργεια χρησιμοποιούμε 7 εκατομμύρια τόνους το χρόνο ηχθιέλαια και ηχθιάλευρα και 200 εκατομμύρια τόνους ε, ε, αλεύρια από σόγια και σογέλαιο μπορούν τα φύκια αυτό να το αντικαταστήσουν όταν παράγονται σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Και έτσι ε, θα αλλιεύουμε λιγότερα ψαράκια για να τα κάνουμε ηχθιάλευρα. Και έτσι θα σωθούν και δάση στη ξηρά. Ε, μπορώ να σας δείξω πολλές εφαρμογές στην επόμενη διαφάνεια. σας πω ότι τα φύκη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ε, για ε, επιλεκτική αποκατάσταση βιολογική. Δηλαδή, τα φύκια μπορεί να είναι φορείς βακτηρίων που διασπούν τα πλαστικά. Επίσης, άλλη ιδιότητα να είναι η λίπανση των ωκεανών, όπου έχουμε νεκρές ζώνες χωρίς οξυγόνο μπορούν τα φύκη να δημιουργήσουν ζώνες που να παράγεται οξυγόνο και αυτό να αλλάξει ριζικά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος είναι οχτώ οι βασικές εφαρμογές των φυκών και των πολύ μικροσκοπικών και των κανονικών φυκιών που φυτρώνουν στη θάλασσα. Ε, τροφές, ζωοτροφές, ε, λιπάσματα, χημικά, καλλιντικά κλπ. Και η Ευρώπη είναι ηγέτης εκεί. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη ε, σε όλους αυτούς τους τομείς. Αυτά και τελείωσα και σας ευχαριστώ. Thank you. And now, uh, σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ασίν, διευθύντρια του Policy Office του WWF. Για πέντε λεπτά παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οργάνωση της διάσκεψης αυτής. Χαίρομαι εκπροσωπώ εδώ την οργανώσή μου που έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αρχής, των αρχών μάλλον, της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Κάποιοι είπαν ότι ο ωκεανός μοιάζει σαν το και εκτιμήσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία στην οικονομία, περίπου 24 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία μπορεί να, να μεταφραστούν σε κέρδη περίπου σε 2,5-3 εκατομμύρια χωρίς να μιλήσουμε για όλα τα άλλη ωφέλη, το οξυγόνο, τα τρόφιμα, αλλά αποτελεί και ε, αναχέτηση, παράγοντα αναχέτηση της κλιματικής απειλής. Επίσης, ε, η οικονομία του ανακαινού αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030 κατά μέγεθος και ε, δημιουργεί ένα προηγούμενο για τις μεταφορές, τη βιοτεχνολογία, την ενέργεια. Ε, αλλά πέρα από ότι εμεί είμαστε οργανώσεις ενδιαφερόμαστε για τη βιοποικιλότητα, όταν βλέπουμε του δείκτες τη υγεία των ωκεανών, δεν οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, Αντιθέτω, ε, κινούνται προ τη λανθασμένη κατεύθυνση. Περίπου το ένα τμήμα, το ένα τρίτο συγγνώμη, των ελευτικών επελευμάτων ε, οι λιμόνες, ε, η μαγκρόβια βλάστηση ε, αποψηλώνονται δύο-τρεις φορές ε, ταχύτερα από τα τροπικά δάση. Μιλάμε για τα τοξικά, τα πλαστικά και την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά έχουν πολύ σοβαρό αντικτύπο στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για την οξύνηση των πιο κρυών υδάτων έχουν αντίκτυπα, αντίκτυπο στην τροφική αλυσίδα. Και κάτι ακόμη που αφορά τον την οργάνωσή μου αφορά την ελεύκανση των κοραλιών. Γιατί είδαμε πριν δύο χρόνια το πιο σοβαρό περιστατικό λεύκανση των κοραλιών. Χάσαμε σχεδόν το ίμιση των κοραλιογενών υφάλων και αν συνεχίσουμε με την ε, σημερινή τάση θα τους χάσουμε όλους τους υφάλους μέχρι το 2050. Και όχι απλώ χάνουμε ένα πολύ όμορφο είδος, αλλά έχει αντίκτυπο αυτό σε εκατομμύρια ανθρώπους από το οποίο εξαρτώνται για το εισόδημά τους και για την προστασία των ε, παράκτων περιοχών αν έχουμε καλή διαχείριση των ωκεανών, τότε θα συνεισφέρει στο να πετύχουμε όλους τους 17 στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξης και αυτά είναι καλά νέα. Αλλά για να επανέλθω σε ό,τι είπε προηγούμενο ομιλήτη οι φιλοδοξίες μας για την οικονομική ανάπτυξη εξαρτώνται από υγιή οικοσυστήματα και τις υπηρεσίε που προσφέρουν. Για να τα πούμε πολύ απλά λοιπόν. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τη φιλοδοξία μας, ε, για την ε, γαλάζια ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για την ανάγκη ελαχιστοποίηση του κινδύνου και να δημιουργήσουμε ανθεκτικότητα στους ωκεανούς ε, εν ώψη της κλιματικής απειλής. Αυτό απαιτεί να προστατεύσουμε πολλά από αυτά τα οικοσυστήματα πριν από το να σκεφτούμε πώς θα τα εκμεταλλευτούμε και να λάβουμε υπόψη τα όρια του πλανήτη, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μόνο ένα πλανήτη και αυτό θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να αποκαταστήσουμε αυτό το φυσικό κεφάλαιο που είναι υποπηλή σήμερα. Θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό Μέρο όλη ε, τη επιχειρηματική πρόταση. Είμαστε λοιπόν σε σημαντικό σταυροδρόμι και αναφέρθηκε αυτό και από νεότερου συναδέλφους. Ε, από την ε, μία πλευρά έχουμε πολιτέ που ζητάνε όλο και περισσότερο δράση και από την άλλη έχουμε τι δημόσιε πολιτικέ και είναι ένα βήμα μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχει ήδη τα νομοθετικά εργαλεία για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία αλλά τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα εργαλεία και θέλω να αναφέρω τρία. Το πρώτο αφορά τη στόχους της κοινή ελευθερικής πολιτικής για την επίτευξη βιώσιμης αλίας μέχρι το 2020, αλλά και την οδηγία πλαίσιο για ε, την θαλάσσια στρατηγική 2020 και αυτό πολύ σύντομα. Και μια άλλη πολιτική σημαντική είναι η σύμβαση για την βιοπικιλότητα, ο στόχος 11 που καλεί για την προστασία τουλάχιστον 10% ε, των ε, παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών. Λέχθα τον ε, αυτών, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπούμε τώρα καλούμε για δράση. Το 2020 θα κάνουμε μία αποτίμηση πολλών διεθνών συμφωνιών, της Συμφωνίας των Περισσίων, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Σύμβαση για την βιοτοπική βιοπικιλότητα, τη CBD. Και γι' αυτό καλούμε για μια νέα όθηση για τη φύση, μια νέα συμφωνία, ένα νέο deal για τη φύση και για τους ωκεανούς και τη βιοπικιλότητα. Πρέπει να ενταχθούν πολύ περισσότερο στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου. Και θα κλείσω με τα τρία μήνυματά μου και θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, να απαντήσει την παγκόσμια Κλίση για βιώσιμε επενδύσει και ανάπτυξη στην παγκόσμια Γαλάζια οικονομία. Δεύτερον, και παγκοσμίω και εσωτερικά να προωθήσει τη βιώσιμη ελεία και την κυκλική οικονομία και να προστατεύσει τρίτον την αρθεκτικότητα των ωκεανών εγκαίρως για την προθεσμία του 2020. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου. Ο κύριος Ζανεμιγκρούτσε, πάλι για πέντε λεπτά. Από τη Ocean Energy Europe. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, Επίτροπε, κύριοι Ευρωβουλευτές, συνάδελφοι. Η δική μας οργάνωση εκπροσωπεί την ενέργεια στους ωκεανούς. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επικεντρωθώ στην Παλήρια και στα παλιριακά κύματα. Εδώ λοιπόν στις εικόνες βλέπετε τι συμβαίνει Πατήστε το ένα παρακαλώ. Μπορεί να ρωτηθείτε. Τι τους χρειαζόμαστε, τους... Τι, τι χρειαζόμαστε την ενέργεια από τους ωκεανούς. Έχω μια διπλή απάντηση. Η πρώτη είναι το κλίμα και η άλλη η βιομηχανική ανάπτυξη. Το κλίμα προφανώς, διότι ξέρουμε ότι έως το 2050 δεν μπορούμε να ε, έχουμε την παραμικρή εκπομπή άνθρακα πλέον για την παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να υπάρχει ανανεώσιμη παραγωγή. Εάν δείτε την έκθεση του IPPC, τα σενάρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τα περισσότερα πιστεύουν ότι πρέπει να φτάσουμε το στόχο της ανανεώσιμης ε, ενέργειας μέχρι το 2050 κατά 100%. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι βιώσιμη και ζήτηση και προσφορά. Για να εξορροπήσουμε τις δύο αυτές ε, διαστάσεις χρειάζεται η κατάλληλη παραγωγή ενέργειας και αποτελεσματικότητα στην ενέργεια, απόδοση στην ενέργεια μάλλον και η σωστή αποθήκευση και γι' αυτό χρειαζόμαστε καταπληρωτικά κύματα. Γιατί? Διότι παράγουμε πολύ διαφορετικό ρυθμό από τη ολική και ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να ελαφρύνουμε τα σχετικά συστήματα. Μέχρι το 2050 μπορούμε να φτάσουμε 10% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα παλιωτικά κύματα των ωκεανών. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η ενέργεια των ωκεανών. Α, να το λέει. Η ενέργεια των ωκεανών σημαίνει και επενδύσει. Και κέρδο. Η Δανία, η Γερμανία έχουν ήδη ωφεληθεί στην διεθνή αγορά, αξιοποιώντα του ωκεανού. Αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλε περιοχέ, σε άλλε χώρε τη Ευρώπη που είναι παραθαλάσσιες μπορούμε να δημιουργήσουμε 400.000 θέσει εργασία στην Ευρώπη. Και αρκετέ και εκτό. Έχουμε πετύχει αρκετά στι διάφορε ακτέ. Αυτά που δείχνουμε προ στιγμή είναι ακριβά, ίσω. Αλλά έχουμε κατεβάσει το κόστο για την νεολική και την ηλιακή ούτω ή άλλω και ανάλογο μπορούμε να κάνουμε, κάτι ανάλογο μπορούμε να κάνουμε για, για του ωκεανού. Λίγο τσιμέντο, λίγο μπετόν ε, κάποια καλώδια και κάτι άλλα εξαρτήματα χρειαζόμαστε και μετά μπορούμε με απλά μηχανήματα να αρχίσουμε να παράγουμε. Η πράσινη ανάπτυξη χρησιμοποιείται ήδη στην ε, ηλιακή και την αιωλική. Θέλουμε το ίδιο να γίνει και στους ωκεανούς λοιπόν. Ε, το γαλάζιο κατά κάποιο τρόπο είναι το νέο πράσινο που θα έλεγε κάποιος, όπως και το όνομα της σειράς εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι και γι' αυτό, για τον περιορισμένο αντίκτυπο ανάλογα με το ποια σκοπιά υιοθετήσει κανείς και το τι αντικτύπους βλέπει στο τοπικό περιβάλλον. Έχουμε τη δυνατότητα να ε, ε, ενεργοποιηθούμε σε περιοχές όπου υπάρχουν ισχυρά ρεύματα. Εκεί όπου υπάρχει λιγότερη βιοποικιλότητα γιατί ο πυθμένης τη θάλασσα είναι βράχια, σκληρά βράχια. Ε, συμπαγή. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι περισσότεροι δακτύλοι, περισσότεροι περισσότερες άγκυρες που να μην καταστρέφουν το θαλάσσιο πυθμένα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για την παραγωγή ενέργειας. Ε, για τα θηλαστικά, ε, για μια σειρά από ενέργειες στη θάλασσα, ειδικά για τις φώκες ας πούμε, και γιατί για την ώρα δεν έχουμε παρατηρήσει να υπάρχουν ε, άλλου είδους προβλήματα μεταξύ της προστασίας των ειδών. Εδώ λοιπόν το νέο πράσινο είναι το γαλάζιο. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να πάμε ως εκεί με τρόπο βιώσιμο και για την αίμα που ζητά να έρθει ο ιδιωτικό τομέα και να αναλάβει πρωτοβουλίες και να επενδύσει, τα ξέρει καλά, φαντάζομαι, αλλά οι επενδυτέ χρειάζονται δύο πράγματα για να επενδύσουν σε νέε τεχνολογίε. Χρειάζονται προβλεψιμότητα και χρειάζονται και κίνητρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν εδώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ κύριε Βέλα, κύριε Μοέδα, για τα πέντε χρόνια σκληρής δουλειά πολιτικού και οικονομική ενίσχυση. Χωρί εσά κάποιε από αυτέ τι διαφάνειε, κάποιε από αυτέ τι τεχνολογικέ λύσει, δεν θα έπλεαν σήμερα στους ωκεανούς όπως σήμερα. Έχουμε πάρει λίγη χρηματοδότηση από τον ορίζοντα 2020. Κάποιες από τις συσκευέ αυτές δεν θα υπήρχαν στη θάλασσα, δεν θα τις είχαμε τρέξει εάν δεν είχατε βοηθήσει κι εσείς. Έκλεισε ε, για δράση, προ ε, για δράση προς τα κράτη-μέλη λοιπόν εδώ, ιδίω στη χώρα των Βράσκων ας πούμε, που έχει πετύχει ιστορικά βήματα πρόοδου. Ε, σε εθνικό επίπεδο χρειαζόμαστε προβλεψιμότητα στην αγορά ε, και προβολή και κάτι που να προσελκύσει τους επενδυτές. Δεν θα επενδύσουν αλλιώς οι επενδυτές σε ένα καπιταλιστικό κόσμο χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία. Εάν είναι κανείς λοιπόν εκπρόσωπο κάτω μέλους, βουλευτή από κάτω μέλους παρατηρούμε, δείτε τι γίνεται με την ενέργεια ε, και τι γίνεται με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε. Αν δεν το κάνετε για τις βιομηχανίες, κάντε το για τις κοινότητες που ζουν σε παράκτηρες περιοχές. Έχουν υποφεληθεί ε, πάρα πολύ από αυτό το είδος την επιχειρηματική δράση, το ίδιο και θα υποφεληθούν από την παραγωγή ενέργειας. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Εάν σας ενδιαφέρουν όσα κάνουμε, κοιτά, ψάξτε μας στο Google. Θα... Είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τις επόμενες δεκαετίες για τα θέματα αυτά και την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τρουέ. Και τώρα θα παρακαλούσα τον τελευταίο ομιλητή να πάρει το λόγο, Κρίστοφ Τούτκατ, Γενικός Γραμματέας της Sea Europe. Thank you, Chairman. Um, Commissioner. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, κύριε Μάισνερ, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του διοργανωτέ τη σημερινή συνεδρίαση που κάλεσαν ε, το Σιγηρόπα. Για όσου δεν μα ξέρετε, είναι οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ναυπηγείων και όσους κατασκευάζουν εξοπλισμό συλλογικά. Είμαστε πάνω από 8.000 εταιρείε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και ε, εκπροσωπούμε τον ευρωπαϊκό τομέα τεχνολογίας. Τώρα τι κάνει ε, μια τέτοια οργάνωση σε μια σύνοδο για τους ωκεανούς. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ότι είναι καταρχήν η συντήρηση, η μετατροπή ε, και η επισκευή του εξοπλισμού πολύπλοκων ε, πλατφόρμων offshore ε, και πλέον και εξακολουθούμε να έχουμε στην Ευρώπη μια παγκόσμια ηγετική θέση και είμαστε περήφανοι, αλλά πάμε και λίγο παραπέρα. Εξετάζουμε περισσότερο την τεχνολογία και τις υποδομές ε, που είναι κατάλληλες για τις ε, ε, δραστηριότητες της γαλλικής οικονομίας. Αν δείτε τα κρουαζερόπλια, πιστεύουμε ότι είναι ένα αυτό πολύ σημαντικό ε, τμήμα των δραστηριοτήτων ε, και κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, ο τομέα μα ε, έχει στην καρδιά του του ωκεανού και τι θάλασσε και θέλει να συνεισφέρει σε βιώσιμη γαλάζια οικονομία και να μειώσει την πίεση που υπάρχει στους ωκεανούς. Και αυτό θα το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε με τους συναδέλφους, με την Waterboard Technology Platform. Αυτή η πλατφόρμα είναι ε, μια νέα στρατηγική ε, ερευνητική ατζέντα και ε, εκεί καλύπτει όχι μόνο τις κλασικές μεταφορές και θα αναφέρω πιο συγκεκριμένα. Καταρχήν, τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό σημαίνει τα παντοπόρα πλοία, αλλά και την εσωτερική ναυσιπλοεία. Εδώ θέλουμε ένα καθαρό ε, τρόπο μεταφορών. Θέλουμε μέχρι το 2030 να φτιάξουμε νέα ποντοπόρα πλοία αλλά και εσωτερική ναυσιπλοεία ε, με μηδενικέ εκπομπέ. Ενώ για τα άλλα σκάφη θέλουμε μείωση 50% των εκπομπών ενώ θα πλέον στη θάλασσα. Και μέχρι το 2050 πιστεύουμε ότι μπορούμε για κάθε πλοίο να έχουμε μηδενικέ εκπομπέ. Και όταν μιλάμε για μηδενικέ εκπομπέ, δεν μιλάμε μόνο για τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά μιλάμε και για τη μείωση τη ρήπανση στη θάλασσα και τη συγχωρήπανση. Και με αυτή την ε, φιλοδοξία ε, θέλουμε να πάμε πέρα από αυτά που συζητάτε, συζητώνται σήμερα στο πλαίσιο ε, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας ε, στο Λονδίνο, αλλά πέρα από το να έχουμε πλωτές μεταφορές, ε, καθαρές και πράσινες, θέλουμε να δούμε και τις γαλάζιες δραστηριότητες, τις δραστηριότητες γαλάζιας οικονομίας. Προηγούμενη ομιλήτρια αναφέρεται, προηγούμενος ομιλητής, συγγνώμη, αναφέρθηκε σε αυτό, οπότε δεν θα αναφερθώ και εγώ αλλά θα επικεντρωθώ σε άλλα πράγματα. Καταρχήν, θέλουμε να προωθήσουμε την προστασία των ωκεανών και των εσωτερικών πλωτών οδών. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει η Ευρώπη να έχει πλήρη ε, ολοκληρωμένη ένα πλήρω ολοκληρωμένο σύστημα ε, παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών και να έχουμε μία ολιστική εικόνα όλων ε, των πλωτών επιχειρήσεων και έτσι θα μπορούμε να έχουμε επιχειρήσεις για απορρίμαση από τα πλαστικά. Επίσης θέλουμε να διευκολύνουμε ε, στις offshore ε, πλατφόρμες ε, να αναπτύξουμε πολλαπλά συστήματα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους στις, παράκτης, στις πλατφόρμες να έχουμε καλές συνθήκες διαβίωσης στη θάλασσα. Ε, και με τέτοιους συνδυασμούς με υπεράκτιες πλατφόρμες ε, θέλουμε να παράγουμε στην Ευρώπη τα πρώτα πλωτά νησιά ε, για κάποιε βιομηχανικέ δραστηριότητε ή ψυχακέ δραστηριότητε και κατοικία μέχρι το 2050. Ε, βέβαια, πρέπει να πληρούνται πολλέ προποθέσει και καταρχήν και τον έφεραν και κάποιοι προηγούμενοι ομιλητέ, η ανάγκη για σημαντικέ επενδύσει ε, στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην κοινοτομία και στο πλαίσιο του Horizon Ευρώπη, αλλά και εκτό του πλαισίου Horizon Ευρώπη. Σήμερα ο τομέα ε, τη ελεύθερη τεχνολογία επενδύει το 10% σε δραστηριότητε έρευνα και ανάπτυξη ε, και είναι ένα από του πρωτοπόρου σε βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη. Αλλά αν θέλουμε να αναπτύξουμε το δυναμικό τη γαλάζια ε, ανάπτυξη ε, πλήρω και θέλουμε καθαρέ θαλάσσιε μεταφορέ, σίγουρα χρειάζονται περισσότερε επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη. Δεύτερον, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων ενιών θα πρέπει να υποστηρίζονται πλήρω με κατάλληλε πολιτικέ και κανονισμού. Αυτά είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο συγκεκριμένα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει για να είμαστε καινοτόμοι και το να, είμαι καινοτό, να είμαστε καινοτόμοι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο σημαίνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο κλίμακα. Τρίπον, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κυρίως ε, για ε, κεφαλικές επενδύσεις ε, και, και επενδύσεις με ένταση κινδύνου. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται καινοτόμα πλοία και πλατφόρμες και για δραστηριότητες γαλάζιας ανάπτυξης. Τέταρτον, ο κλάδος θα πρέπει ε, να απασχολεί νέους με ενθουσιώδη κίνητρα και ε, με υψηλά προσόντα για να παράγουν καινοτόμες τεχνολογίες και να μπορούν να προσαρμοστούν σε έναν ε, κόσμο τεχνολογικό που αλλάζει γρήγορα. Και τέλος, για τον ευρωπαϊκό ε, τομέα τεχνολογία στη θάλασσα, χρειαζόμαστε μια στρατηγική που την αποκαλούμε leadership strategy. Αυτό θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας ε, στον ε, παρασκευή, στην κατασκευή ε, του εξοπλισμού αλλά και την αφήγηση πλοίων και θα πρέπει να ωφεληθεί όχι μόνο ο τομέας αλλά και όλη η πλωτική κοινότητα όπως και οι δραστηριότητες της γαλάζιας ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, ε, το μήνυμά μου με δύο λόγια είναι ότι θέλουμε γαλάζια ανάπτυξη και για τα ναυπηγεία. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, είναι πολύ σημαντικό και για τις μελλοντικέ γενιές και για τον πλανήτη και θέλουμε να βάλουμε τα δυνατά μας να αναλάβουμε και τη δική μας ευθύνη προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται το τελευταίο πάνελ υπαριθμών 3. Ξέρω ότι Ορισμένοι είναι έτοιμοι να κάνουν ερωτήσεις, αλλά με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε ερωταπαντήσεις για τον το λόγο ότι σε λίγο μας τελειώνει η διερμηνία. Και βεβαίως θέλετε να ακούσετε και το κλείσιμο και σας παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. κυρία Μάισνερ, κυρίες και κύριοι, ακόμα παραμένουν πολλοί στην αίθουσα. Θα φανταστικό. Μην φοβηθείτε ότι θα υπάρξει άλλο πάνελ που θα μακρηγορήσει. Απλώς τα καταληκτικά σχόλια και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Βέλα να κάνει τις θεματικές ε, ε, καταληκτικές παρατηρήσεις και εγώ τις ευχαριστίες για να κηρύξουμε το πέρας αυτής της διοργάνωσης. Ευχαριστώ πολύ Γκεζινέ, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το απόγευμα. Μεγάλη πηγή έμπνευση οι παρουσιάσεις και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση. Και πολύ ενθαρρυντικό είναι να βλέπουμε ότι όποιες κάνουν είναι οι προτάσεις μας, οι πολιτικές μας απόψεις, συμφωνούμε όλοι για το εξή ότι χρειαζόμαστε μια δράση ισχυρή και συντονισμένη για τον κανονισμό, για τον, τους ωκεανούς μας, αλλιώς ε, η οικονομία μας κινδυνεύει και οι ζωές μας οι ίδιες και το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πολύ φιλόδοξη δράση για να μειώσει την παραγωγή πλαστικών, να καταπολεμήσει τη λαθρέα αλληλεία και να καταστήσει τα αποθέματα βιώσιμα, έτσι ώστε να υποστηρίξει την γαλάζια οικονομία να αναπτύξει τη θαλάσσια έρευνα και την επιτήρηση των ωκεανών. Όπως γνωρίζετε, παραμένουν μεγάλες όμως οι προκλήσεις. Τα ωκεάνια συστήματα είναι περίπλοκα και είναι πολλές οι πιέσεις, κλιματική αλλαγή, ρήπανση, βιοπικιλότητα και απώλειά της και υπεραλίευση. Όλα αυτά θα εξακολουθήσουν να ε, πλήττουν τους ωκεανούς. Μέχρι το 2050 θα είμαστε 9 με 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη και θα αυξηθούν οι πιέσεις όλες αυτές. Θέλω να σας ε, ε, διαβεβαιώσω ότι είναι προσιλωμένη σε αυτή την προσπάθεια πλήρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει ε, τις δράσεις είτε πρόκειται για το νέο πρόγραμμα Horizon ε, Europe με εστίαση στους ωκεανούς, είτε ε, στη νέα θαλάσσια στρατηγική και το Ταμείο μετά το 2020 για τη θάλασσα και την αλία. Και επίσης ε, για την εξωτερική χρηματοδότηση και το αντίστοιχο μέσο μετά το 2020. Είναι παγκόσμιο ηγέτης, αξιόπιστος η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι προσιλωμένη και παραμένει στο να πρωταγωνιστεί διεθνώς. Ε, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, τη ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην εφαρμογή της συνθήκης του Παρισιού, της συμφωνίας μάλλον, και για την προστασία της θαλάσσιας βιοπικιλότητας στις ανοιχτές θάλασσες και τους ωκεανούς. Και ξέρουμε ότι για να παραμείνουν υγιείς οι ωκεανοί θα πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε στενότερα. Για το λόγο αυτό και μαζί με τη συνάδελφό μου Γκερίνη χαράσουμε ένα φόρουμ για τη διακυβέρνηση των ωκεανών παγκοσμίω, με εμπειρογνώμονε, με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακούς ερευνητές και ε, ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις για να δώσουν συνέχεια στις δικές μας προτεραιότητες, για να συζητήσουμε τις διεθνείς προκλήσεις και προβλήματα και πιο σημαντικό για να συστήσουμε δράση. Αυτό θα είναι ένα ακόμα βήμα στις προσπάθειές μας για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, προς τους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους Οκεανούς. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια επιτροπή Οκεανών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια μόνιμη επιτροπή. Και χρειάζεται και περαιτέρω δράση. Φυσικά θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό και ελπίζω και εσείς να συνεχίσετε και να συναντηθούμε για να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο γαλάζιο ωκεανό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Καρμενουβέλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που παραμείνατε μέχρι το τέλος. Καλά και εγώ παρέμεινα. Αλλά Ήθελα να γίνει αυτή η διάσκεψη εδώ και πάρα πολύ καιρό και φυσικά θα παραμείνω, αλλά ε, συνήθω οι επίτροποι έχουν τόσε πολλέ υποχρεώσει και αντισταθήκατε σε όλου του πειρασμού και παραμείνατε εδώ. Είναι θαυμάσιο αυτό και πραγματικά ένα ε, προσεκτικός παρατηρητής καταλαβαίνει ότι τα λαμβάνετε αυτά σοβαρά υπόψη και το ξέρω εγώ φυσικά ότι τα λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, πρέπει να σας κάνω ένα σχόλιο επειδή είπα ότι ορισμένοι ρωτούσαν γιατί έχει πλαστικό καπάκι αυτό το μπουκάλι. Έχει μια ιστορία το μπουκάλι αυτό. Συνήθως εδώ έχουμε παντού πλαστικά μπουκάλια. Και το δικό μας Intergroup αρνήθηκε να έχει. Έχει μόνο ποτήρια και γυαλί. Αυτό είναι ένα συνδυασμός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ε, καπάκι είναι πλαστικό, αλλά είναι ανακυκλούμενο. Το άλλο είναι γυαλί. Και το κοπάνισα. Πάντως θα πρέπει να ε, σκεφτούμε πώς ε, να ε, αποφύγουμε να έχουμε μπουκάλια πλαστικά μιας χρήσης. Θέλω να πω κι άλλα. Ήταν συναρπαστική αυτή η διάσκεψη. Ικανοποιήθηκα πάρα πολύ και είμαι πανευτυχής που το καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τόσο κόσμο. Ε, ε, χίλιοι εγγεγραμμένοι είναι πολύ. Εγώ θα προτιμούσα ένα εκατομμύριο. Θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ε, να γνωρίζει ένα εκατομμύριο κόσμο τι γίνεται με τους ωκεανούς είναι μια καλή αρχή πάντως και η χίλιοι. Και ως ε, ιδέα είναι θαυμάσια και λαμπρή ιδέα ε, για έναν οργανισμό για τους ωκεανούς εκτός από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Και τώρα έχω τη χαρά και την ευχαρίστηση να σας ευχαριστήσω όλους. Όλους τους προσκεκλημένους, τους ε, ισταμένους, γιατί χωρίς κοινό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διάσκεψη. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ομιλητές, ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ποτέ δεν έχω δει διάσκεψη με υψηλού επίπεδου με τόσους πολλούς ευρωβουλευτές. Έτσι δεν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί θα πρέπει να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό ρόλο. Ευχαριστώ όλους όσοι διοργάνωσαν, ιδιαίτερα το ιδιαίτερο γραφείο ε, του Προέδρου Ταγιάννη και κυρίω την κυρία Μαγδαλένα Πιόρουν και Γκοσάλ Μεντόσα Ασένση, αλλά κυρίως την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, Ραμόν Βαν Βάλτεβελ και την Αλεξάνδρα Λαμόρ που είχαν πολλή δουλειά και εκτός αυτού θα ήθελα και πάλι να αναφέρω γιατί ξέχασα μια γενική διεύθυνση στα εισαγωγικά μου σχόλια Γενική Διεύθυνση Director, Directorate General είναι στα αγγλικά ΜΑΡΕ και RTD αλλά και περιβάλλοντος ε, ε, ξέχασα να την αναφέρω αυτή τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Και τώρα, χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, ένα τελευταίο. Όλοι εσείς εδώ παρόντες αγαπάτε τους ωκεανούς. Για μένα είναι κρίσιμο να βλέπουμε ότι χρειάζεται προστασία ωκεανός. Ε, ένα πλανήτη έχουμε μόνο. Αυτό το πλανήτη έχουμε, αυτούς τους ωκεανούς. Πρέπει να τους προστατεύουμε. Και ο κόσμος προστατεύει ό,τι αγαπάει. Λοιπόν, φεύγοντας από εδώ θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να βγούμε και να κάνουμε τους άλλους ανθρώπους να αγαπήσουν τους ωκεανούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή επιστροφή και στο επανειδήν. Κάποια άλλη φορά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.